Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, καθίστε παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε. Για όσους δεν παρακολούθησαν ε, την συνεδρίαση από το πρωί, να σας πω Όταν μια σπουδαία μέρα έχουμε μια συνεχιζόμενη ακρόαση, πολλή δουλειά, πολλή ουσία, πολύ σημαντικά θέματα και τώρα ξεκινάμε το δεύτερο ήμιση αυτής της σκληρής μέρας δουλειάς. Με αυτή την ακρόαση θέμα την κατάσταση στην Ουγγαρία. Έχουμε διοργανώσει αυτή την ακρόαση για την κατάσταση στην Ουγγαρία, πράγμα που ζήτησαν διάφορες ομάδες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Και βεβαίως σας καλωσορίζω όλους. σε αυτή τη συνεδρίαση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή μας που είναι αρμόδια για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις και καλωσορίζω και τους διακεκριμένους ε, προσκεκλημένους και συμμετέχοντες που βρίσκονται εδώ στο Προεδρείο. Επίτροπος Νέλη Κρούς, καλωσορίσατε, είναι τιμή μας που είστε σήμερα εδώ. Τον ε, ε, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κύριο Χαραντάκη, τον κυρία Λεβάη, που είναι γενική διευθύντρια αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τους προσκεκλημένους μας που έχουν έρθει για να συμβάλλουν στην συζήτηση που θα ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να θυμίσω την κατάσταση ως έχει. Στις 19 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, η διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσε την ε, ΛΥΜΠΕ, την Επιτροπή μας, να διοργανώσει μια δημόσια κρόση για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Η κατάσταση αυτή βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ που έγιναν στις 25 Μαΐου και 12 ε, Ιανουαρίου. Ο κύριος Τόμας Μάρκετ, ο γραμματέας της Επιτροπής βάνος του Συμβουλίου της Ευρώπης, παρουσίασε τα συμπεράσματα της έκθεσης που έγινε σε αυτή την Επιτροπή. Στις 18 ε, Ιανουαρίου δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπής έγινε με και μετά ακολούθησε η συζήτηση για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία, στην Ολομέλεια τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την παρουσία της δανικής κυβέρνησης ε, της, του Προέδρου Μπαρόζο της Επιτροπής, του ε, Αντιπροέδρου της Επιτροπής κυρίας Ρέντινγκ και του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, κυρίου Βίκτορ Όρμπαν. Και έχει προγραμματιστεί ένα ψήφισμα για την Σύνοδο της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου Φεβρουαρίου, της δεύτερης δολομέλεια δηλαδή, που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Γι' αυτό και προσβλέπω σε μια καρποφόρα συζήτηση. σα καλωσορίζω όλου, και θα ήθελα απλά να σα πω ποια είναι η δομή αυτή τη ακρόαση. Θα ακούσουμε τέσσερι σειρέ από εισηγήσει. Όλοι οι ομιλητέ θα πρέπει να τηρήσουν, σας ε, παρακαλώ εξ αρχής, όλοι οι ομιλητές θα πρέπει να τηρούν τα χρονικά όρια που τους έχουν δοθεί, ώστε να μπορέσουμε να χειριστούμε την κατάσταση, γιατί έχουμε μια τάση εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να μακρηγορούμε λίγο στις συζητήσεις, πέρα από τα λογικά χρονικά όρια. Οπότε σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας τα το χρόνο που σας έχει δοθεί. Κάθε μια από τις εισηγήσεις θα ακολουθηθεί από συζήτηση. Πάντοτε ως πρόεδρος προσπαθώ να διευρύνω το μάκρος της συζήτηση και βεβαίως το πεδίο για όσους περισσότερους γίνεται. Σας καλώ λοιπόν από τώρα όσους θέλετε να συμμετέχετε να προβλέψετε δύο λεπτά έκαστος για την ε, ομιλία σας και να παρακολουθήσετε και να τηρήσετε μάλλον το χρόνο ερωτήσεων, να υποβάλλετε ερωτήσεις και όχι να κάνετε αγορεύσεις. Σας θυμίζω λοιπόν ότι θα γίνει ένας πρώτος γύρος συντονιστών και μετά θα υποβάλουν ερωτήσεις τα υπόλοιπα μέλη. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη συνεδρία. Ο πρώτος ομιλητής είναι η κυρία Νέλη Κρούζ, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα. Είναι τιμή μας που βρίσκεστε εδώ, κυρία Κρούζ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης κύριε Πρωθυπουργέ. Ε, ξέρω, ναι, σας ε, έδωσε έναν ε, ακόμη τίτλο. κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω σήμερα εδώ. Ξεκολουθώ να έχω σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουγγαρία. Και το ίδιο ανησυχεί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό αφορά τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι, ε, είμαι ευτυχής που είμαι εδώ και θα έχω την ευκαιρία να το συζητήσω άμεσα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και το συζήτησα σήμερα το πρωί πριν από αυτή την ακρόαση. Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα στείλαμε τρεις επιστολές επί παραβάσεις γκρικές αρχές όσον αφορά την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, την ε, ηλικία συνταξιοδότηση των δικαστών και την ανεξαρτησία της αρχής προστασίας των δεδομένων. Και για αυτά τα σημεία οι ουγγρικές αρχές δεν έχουν ακόμα απαντήσει. Οπότε δεν θα σχολιάσω περαιτέρω αυτές τις διαδικασίες. Ωστόσο, οι ανησυχίες μας είναι ευρύτερες σε σχέση με την οικονομική πολιτική της Ουγγαρίας, την ποιότητα της δημοκρατίας και την πολιτική νοτροπία της. Γι' αυτό θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία σήμερα για να μιλήσω για το περιβάλλον των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυτή τη στιγμή, καθώς και τη δομή της ε, νομοθεσίας περί ελευθεροτυπίας. Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί είναι θεμελιώδες δικαίωμα η ελεύθερη έκφραση. Υπάρχει και ε, οικονομική σημασία, διότι οι ιδιώτες επενδυτές καθώς και τα διεθνή θεσμικά όργανα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν πρόσβαση στα ανεξάρτητα αναλύσει των μέσων μαζικής ενημέρωση. Οι Ουγγρικέ αρχέ θα πρέπει να προσέξουν ώστε να μην δώσουν οποιαδήποτε άλλη εντύπωση. Αντιθέτως, χρειαζόμαστε θετικά μηνύματα. Όπως ε, τόνισε ο πρόεδρος Μπαρόζο στην τελευταία σύνοδο τη Ολομέλεια του Κοινοβουλίου πριν από τρεις εβδομάδες, ενεργώντας με υπεύθυνο και ε, δημοκρατικό τρόπο προς το συμφέρον όλων των Ούγγρων πολιτών, οι Ουγγρικές αρχές μπορούν να κερδίσουν και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, των φορέων και των επενδυτών μέσω ενός ε, νομικά σταθερού περιβάλλοντος που βασίζεται στο κράτος δικαίου, στις δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιπλέον, απειλέ ε, στον τύπο θα πρέπει να θεωρηθούν μέρο μια ευρύτερη εικόνα. Εγώ η ίδια έχω μιλήσει με ανθρώπου από την Ουγγαρία. Μόλι τι προάλλε συνομίλησα με έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο επιχειρηματία του δικτύου, έναν από τους νέους ε, συμβούλους μου για τα ψηφιακά θέματα και η εικόνα που μου παρουσίασε είναι πολύ ανησυχητική. Για παράδειγμα, μιλά για μια χώρα όπου διακρίσεις κατά των μειονοτήτων είναι πολλές και η κατάσταση επιδεινώνεται. Μου είπε επίσης πως οι άνθρωποι των μειονοτήτων είναι, γίνονται θύματα διακρίσεων όταν αναζητούν ε, απασχόληση. Μιλά για ισχυρισμούς ότι η αστυνομία έχει λάβει διαταγές να παρακολουθεί τις μειονότητες, ότι ο ρατσισμός στα σχολεία γίνεται πιο ανοιχτό και γίνεται και πιο αποδεκτός και ότι μάλιστα υπάρχουν φόβοι για βίες επιθέσεις. Το συγκεκριμένος άνθρωπος, ο ίδιος από την κοινότητα των Ρωμά, σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει τη χώρα. Δεν θέλησα να βιαστώ και να προβώ σε κρίσεις επί τη βάση αυτών των δηλώσεων. Όμως, ο περιορισμό τη ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση θα πρέπει να εξεταστεί σε αυτό το, υπό αυτό το πρίσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πλουραλισμό των ΜΜΕ, η δυνατότητα να ακούγονται διάφορε απόψει και φωνέ είναι ακόμα πιο σημαντική. Τον Ιανουάριο της περασμένης χρονιά, εγώ ασχολήθηκα με τα πιο σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την νομοθεσία ΜΜΕ της Ουγγαρίας. Η συμβατότητά τους με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εν γέννη και με την οδηγία περί υπηρεσιών. Και έχουμε συνεργαστεί στενά με τούτον εδώ τον Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα μαζί του έχουμε συνεργαστεί για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην συμμόρφωση με την περιορισμένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωση σε αυτό το τομέα. Και υπογραμμίζω ότι είναι περιορισμένη η σχετική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά επίσης κατέστησα σαφές ότι παρακολουθώ τις εξελίξεις και ότι θα ε, ε, υψώνω τη φωνή μου όταν αυτό χρειάζεται. Και γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ένας από τους λίγους ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν απομείνει και που δίνουν μια ανεξάρτητη φωνή στην τελευταία, ε, στον τελευταίο διαγωνισμό για τις συχνότητες στην Βουδαπέστη φαίνεται πως δόθηκε προτεραιότητα ε, σε σταθμούς ποικίλου περιεχομένου και όχι σε σταθμούς ε, πολιτικής ανάλυσης. Εγώ Ανησυχώ όταν γίνεται τέτοιο είδου διάκριση ει βάρο των ΜΜΕ και του πλουραλισμού. Για να είμαι ομή, εάν θεσπίζονται τεχνικές διατάξεις που είναι κατά των πολιτικών συζητήσεων στο ραδιόφωνο, να μην εκπλαγείτε όταν γίνεται λιγότερη πολιτική συζήτηση στο ραδιόφωνο. Φυσικά εγώ δεν είμαι εκπρόσωπο για κάποιο συγκεκριμένο ΜΜΕ, αλλά Είχα λεπτομερή συζήτηση με τον κύριο Αράδο πριν από δύο εβδομάδες και είμαι βέβαιος πως ο ίδιος μπορεί να μιλήσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση του ραδιοφώνου κλαμπ. Αλλά χρειάζεται να βρούμε μια βιώσιμη λύση που θα επιτρέπει ένα πλουραλιστικό τοπίο για τα ΜΜΕ που θα μπορούν να σχολιάσουν και να προβούν σε πολιτικές αναλύσεις ε, ε, στα ΜΜΕ και στο ραδιόφωνο πιο συγκεκριμένα. Όπως πολύ γνωρίζετε, στις 19 Δεκεμβρίου 2011 ε, το Ουγγρικό Συνταγματικό Δικαστήριο βρήκε ότι η νομοθεσία περί ΜΜΕ περιόριζε το συνταγματικό δικαίωμα των, των ΜΜΕ και κάλεσα τις ουγγρικές αρχές να διορθώσουν αυτά αυτά τα προβλήματα. Φαίνεται πως τώρα προετοιμάζεται σχετική νομοθεσία ευθυγραμμισμένη με αυτές τις αποφάσεις και σίγουρα είναι αυτό ευπρόσδεκτο, αλλά όχι αρκετό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο σεβασμός της ελευθερίας των ΜΜΕ και ο πλουραλισμός δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι να αφορά μόνο τα τεχνικά ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας. Αφορά επίσης την εφαρμογή και την προώθηση θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών στην πράξη. Τέλος, είναι επίσης ε, ο πλουραλισμός των ΜΜΕ και η ελευθεροτυπία που προσφέρουν στην σωστή ατμόσφαιρα και την πολιτική νοοτροπία. Μια πρόσφατη μελέτη, κυρίες και κύριοι βουλευτές, υποδεικνύει ότι η νομοθεσία περί ΜΜΕ της ε, Ουγγαρίας ξεπερνά τις ευρωπαϊκές πρακτικές και προδιαγραφές, ιδιαίτερα εάν εξετάσουμε το πεδίο εφαρμογής και τις επιπτώσεις, αν δούμε τον συνδυασμό των διατάξεων όσον αφορά τις αρχές ε, των ΜΜΕ και την κεντρική δομή, τις ε, αρμοδιότητες της εξουσίας της, ιδιαίτερα η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, καθώς και το πεδίο εφαρμογής των, μέσων, των νομοθεσιών περί ΜΜΕ για τα οπτικοακουστικά, το ραδιόφωνο, online και τον έντυπο ε, τύπο και τα εξή είναι γεγονότα και όχι μύθος. Ο κίνδυνος παραβίασης ασαφών κανόνων μπορεί να οδηγήσει στην αυτολογοκρισία, ακόμα και αν δεν επιβληθούν ποτέ πρόστιμα. Επίσης, ίσως θα γνωρίζετε την ανεξάρτητη ομάδα ευρωπαϊκού επίπεδου για την ελευθερία του τύπου και του πλουραλισμού με πρόεδρο τον ε, κύριο Φράιμπεργκ, πρώην πρόεδρο της Λετωνίας, η οποία ομάδα αφού μελέτησε την υπόθεση της Ουγγαρίας 25 Ιανουαρίου, κατέληξε στην αξιολόγηση και παραθέτω ότι η Ουγγαρία έχει θέσει τον εαυτό του σε μια θέση δυνητικού κινδύνου όσον αφορά την ελευθερία του τύπου και η κυβέρνηση σοφό θα ήταν να σκεφτεί πώς θα βγει από αυτή την κατάσταση. Τέλος παράθεσης. Και γι' αυτό και η Ουγγρική κυβέρνηση χρειάζεται να κάνει περισσότερα και να δράσει γρήγορα ώστε να καθησυχάσει την Κομισιόν, την Επιτροπή και όλους όσους ανησυχούν και να δείξει πως είναι σοβαρή σε σχέση με την προστασία της ελεύθερης έκφρασης και του πλουραλισμού των ΜΜΕ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει θεσπίσει προδιαγραφές για να προστατεύσει την Ευρώπη εδώ και 50 χρόνια και περισσότερο. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά μαζί του για πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της ελευθερίας των ΜΜΕ. Πρόσφατα μίλησα με τον κοινωνικό γραμματέα Γιάκλαντ του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι έτοιμοι να ενεργήσουν. Η Κομισιόν περιμένει δύο βασικά πράγματα από την Ουγγρική κυβέρνηση. Και τις τελευταίες εβδομάδες και πάλι σήμερα έχουμε καταστήσει σαφή αυτά που επιθυμούμε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στους συναδέλφους του. Και σήμερα θα, πρέπει, θα σας τα αναφέρω ρητά. Πρώτον, η Ουγγρική κυβέρνηση θα πρέπει ρητά και με διαφάνεια να ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης μια συνολική γνωμοδότηση για τη συμμόρφωση της νομοθεσίας περί ΜΜΕ και την πρακτική της εφαρμογή και την συμμόρφωσή της με τις θεμελιώδεις αξίες όπως ε, συμπεριλαμβάνονται στην ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεύτερον και εξίσου σημαντικό είναι ότι οι Ουγγρικές Αρχές θα πρέπει να δεχτούν και να εφαρμόσουν οποιαδήποτε συγκεκριμένη σύσταση θα προκύψει από τα πορίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποσχέθηκε ε, ότι αυτά τα δύο θα γίνουν στην συνεδρίασή μας στην διαπροσωπική πριν από δύο εβδομάδες και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι με επιμονή θα, παρατη... θα παρακολουθώ την επίτευξη αυτών των στόχων. Εγώ περιμένω λοιπόν από πλευρά τη Ουγγρική κυβέρνηση δημόσια δέσμευση και για τα δύο αυτά, τους δύο αυτούς στόχους, όσο γίνεται πιο ζητήμα. Ιδανικό θα ήταν σήμερα να γίνει η δέσμευση αυτή και η Κομισιόν δεν είναι ικανοποιημένη με την κατάσταση μέχρι ότου οι ανησυχίες του Συμβουλίου της Ευρώπης να αντιμετωπιστούν. Δεν έχουμε χρόνο να σπαταλήσουμε. Θα πρέπει η Ουγγρική κυβέρνηση να άρει όλες τις αμφιβολίες όσον αφορά την ε, προσήλωσή της στις ευρωπαϊκές αρχές. Και τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στις συνομιλίες μας ήταν σαφής. Ελπίζω πως και στη σημερινή μας, στην τωρινή του ομιλία θα είναι το ίδιο σαφής. Ε, χρειάζεται λοιπόν σαφήνεια χωρίς αντίσταση και αυτό ελπίζω πως θα γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Γανέλη Κρούς. Τώρα θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στη κυρία Λεμπάιτ της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω μέρος σε αυτή τη συζήτηση για ένα μάλιστα τομέα που είναι πολύ σημαντικός και ενώ το τομέα της δικαιοσύνης. Και στο πλαίσιο αυτό, ο προβληματισμός και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από την Επίτροπο Νέλη Κρούς ε, είναι τα ίδια με της Επιτρόπου ε, Ρέντινγκ για το τομέα της δικαιοσύνης. Συμμεριζόμαστε αυτές τις ανησυχίες και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη δήλωση του Προέδρου Μπαρόζο στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Είπε τότε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο και θα πρέπει να είμαστε σαφείς ε, στις αξίες μας, ε, ε, στεναροί στις αρχές και δίκαιοι στη μέθοδό μας. Και στον τομέα της δικαιοσύνης αυτό ακριβώς έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν στις 17 Ιανουαρίου αποφάσισε να γύρει δύο διαδικασίες επί παραβάση κατά της Ουγγαρίας ζητώντας διευκρινήσεις για ένα επιπλέον θέμα την ανεξαρτησία δηλαδή της δικαστικής εξουσίας της δικαιοσύνης στην Ουγγαρία. Θα ήθελα τώρα να σας απαριθμίσω τις συγκεκριμένες ανησυχίες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, ως προς την πρώτη υπόθεση επί παραβάση που αφορά την ε, ανεξαρτησία της αρμόδιας αρχής προστασίας των δεδομένων. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί εδώ στεματοφύλακα της συνθήκης και προσπαθεί να εξασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών με την κοινοτική νομοθεσία, την ενωσιακή νομοθεσία. Υπό αυτό το σκεπτικό δηλαδή δράει η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων. Γνωρίζετε όσοι είστε εξοικειωμένοι με τα θέματα της προστασίας δεδομένων ότι η ανεξαρτησία της αρμόδιας αρχής, αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων κατοχυρώνεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην σχετική οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Αυτά είναι τα τρία ερίσματα της ανεξαρτησίας της εποπτικής αρχής. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και αναθεώρηση ε, πρόσφατα της ε, ε, προστασίας των δεδομένων. Η νέα Ουγγρική Εποπτική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων για να πληρεί πλήρω αυτό το, αυτή την απέτηση, θα πρέπει να πληρεί πλήρως την απέτηση αυτή της ανεξαρτησίας. Μία πτυχή της ανεξαρτησίας τη εποπτική αρχής ε, αφορά τη θητεία του Προέδρου αυτής της εποπτικής αρχής. Δεν μπορεί ε, χωρίς λόγο και αιτία να ε, περατώνεται η θητεία του Προέδρου της εποπτικής αυτής αρχής. Θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένοι λόγοι και μάλιστα η ε, ε, ε, ο πρόορος τερματισμός της θητείας του πρώην πια Προέδρου της Εποπτικής Αρχής της Ουγγαρίας αποτελεί δημιουργεί μάλλον εύλογες ανησυχίες για το κατά πόσο είναι όντως ανεξάρτητη αυτή η Εποπτική Αρχή. Στα πλαίσια του συντάγματος υπάρχει εγγύηση για την ανεξαρτησία της νέας ε, εποπτικής αρχής προστασίας των δεδομένων. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη ανησυχία μας για την πρώτη απόλυση του διευθυντού της ε, εποπτικής αρχής. Δεύτερο πρόβλημα αφορά την πρώτη συνταξιοδότηση των δικαστών, εισαγγελέων και δημοσίων συμβολογράφων. Ένα δεύτερο ζήτημα που μας προβληματίζει. Η Ουγγαρία τροποποίησε το την ηλικία πρόορης δεξιοδότηση για τις κατηγορίες αυτές από τα 70 χρόνια που ήταν αρχικά στα 62 χρόνια που ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Το πρόβλημα είναι ότι η ηλικία συνταξιοδότηση, ε, η γενική, η βασική, δεν είναι υποχρεωτική για όλου του εργαζόμενου. Αν διαβάσουμε την Ουγγρική νομοθεσία, διαπιστώνουμε ότι θα ήταν υποχρεωτική όμω για του δικαστέ, του εισαγγελεί και του ε, συμβολογράφου που σημαίνει ότι μετά τα 62 οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν πλέον να εργάζονται. Και για τους υπόλοιπους, ενώ για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους ο κανόνας είναι πιο ελαστικός. Δεν ε, δόθηκε καμία αξιόπιστη αιτιολόγηση για την ε, μεταρρύθμιση αυτή του, όρου, του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των τριών αυτών κατηγοριών δικαστών, εισαγγελέων και συμβολογράφων. Μάλιστα, φαίνεται υπάρχει αντίφαση με το γεγονός ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που αποφασίστηκε το 2009 από τις Ουγγρικές Αρχές θα αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 65 χρόνια. Και μάλιστα αυτό θα γίνει σε μία οκταετή περίοδο. Ενώ οι τροποποίησεις του όρου του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότηση για του ε, δικαστέ από τα 70 στα 62, η μείωση θα γίνει μέσα σε ένα χρόνο μόνο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο μεταρρυθμίσεων, τη ειδική για του δικαστέ εισαγγελεί και συμβολογράφου και τη γενική. Για όλα σε αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι το μέτρο αυτό δεν ήταν ε, ανάλογο με το σκοπό, ούτε, συνάδει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που απαγορεύει την ε, διακριτική μεταχείριση για λόγο ηλικίας στον τομέα της απασχόλησης. Η τρίτη ανησυχία που είχαμε και που εκφράστηκε σε μια επίσημη προειδοποίηση που στείλαμε όταν η Επίτροπος Ρέντινγκ ζήτησε διευκρινήσεις από την Ουγγρική κυβέρνηση αφορούσε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης του δικαστικού κλάδου. Πρόκειται για ένα θέμα που σχετίζεται με την πρόορη ε, διακοπή της εντολής του πρώην Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου που είχε αρχικά εκλεγεί για μία εξαιτία, τον Ιούνιο του 2009 και ευνίδια διακόπη η θητεία του στα τέλη του 2011. Επιπλέον, ο πρόεδρος του νέου Εθνικού Δικαστικού Γραφείου ε, ε, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους πόρους, τον προπολογισμό και την κατανομή των υποθέσεων δημιουργεί κάποιου προβληματισμού για εκεί. Δεν υπάρχει καμία νόμιμη διαδικασία λήψη αποφάσεων για την επιχειρησιακή διαχείριση των δικαστηρίων ή άλλε ασφαλιστικές δικλείδε ή εχέγγυα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης Και μάλιστα η πρόορη διακοπή του πρώην Προέδρου του Ανατάτου Δικαστηρίου καθώς και η συγκέντρωση των εξουσιών στο γραφείο αυτό δημιουργεί αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και αποτρέπει τους πολίτες από την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους ενώπιον του δικαστηρίου, όπως κανονικά κατοχυρώνεται από το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ ζήτησε διευκρινήσεις για το σημείο αυτό και επιπλέον ενημέρωση από τις Ουγγρικές Αρχές. Τώρα, τι ρώτησε η... και τι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις Ουγγρικές Αρχές. Ε, Ζήτησαμε λεπτομεριακές απαντήσεις και προτάσεις για να επιλυθούν τα προβλήματα και μάλιστα σε το χρόνο που δικαιολογείται φυσικά από τον αντίκτυπο που, θα, που είχαν όλες αυτές οι αποφάσεις για τους ε, θυγωμένους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκτιμήσει τα μέτρα που θα ανακοινώσουν οι Ουγγρικές Αρχές και θα αποφασίσει με βάση αυτές τις επίσημες απαντήσεις ε, τι πορεία θα ακολουθήσει. Προς το παρόν συνεχίζονται οι τεχνικές επαφές με τις Ουγγρικές Αρχές προκειμένου να βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα αυτά. Είναι σαφές πάντως ότι δεν πρόκειται να διστάσουμε και θα συνεχίσουμε τα διαβήματά μας, αν το κρίνουμε απαραίτητο. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τις επίσημες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις που περιμένουμε από τις Ουγγρικές Αρχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λεμπάχη. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση που μας κάνατε. Τώρα περνάμε στην ομιλία του Αντιπροέδρου της Ουγγρικής Κυβέρνησης και Υπουργό Δικαιοσύνης και Πολιτικής Διοίκησης, τον κύριο Ντούνταξ να βράξει. Καλώ ήρθατε και έχετε το λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ο τίτλος της ακρόασης αυτής είναι αρκετά ευρύς. Η κατάσταση στην Ουγγαρία. Η κατάσταση δηλαδή συνολικά στην Ουγγαρία. Και η κυρία Γενική Διευθύντρια και η κυρία Επίτροπος μόλις μίλησαν για το θέμα αυτό. Αλλά από τις εισηγήσεις αυτές αποκρισταλώθηκε ότι πρόκειται για πολύ συγκεκριμένους τομείς. Να εξετάσουμε λοιπόν καταρχάς το πρώτο τμήμα να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίδεται να τοποθετηθώ, να παρουσιάσω συνοπτικά τα όσα έχει πράξει και εξακολουθεί να πράττει η κυβέρνηση. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι ακόμα ρευστά. Έχουμε καλές επαφές με την ε, Επίτροπο, είμαστε σε διαρκή επαφή. Το πράξαμε αυτό άλλωστε και στο παρελθόν σε ό,τι αφορά το νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα, έγινε εδώ πέρσι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο στην Επιτροπή σας μια σχετική συζήτηση, η οποία και οδήγησε στην εφαρμογή των παρατηρήσεων στις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα όμως το θέμα είναι διαφορετικό. Επιτρέψτε μου στην ακρόαση αυτή να ξεκινήσω από τον τίτλο, από την επιγραφή αυτή. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ευρύ στην κάλυψή του ο τίτλος αυτός, η επιγραφή αυτή. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να περιοριστεί κάπως. Το θέμα είναι η συνεργασία α, εσωτερικών επιτροπών και οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, αυτή τη συνεργασία βρίσκομαι και εδώ σήμερα έχω παραστεί και στο παρελθόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο ε, Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν έχει μιλήσει ενώπιον της Ολομέλειας και θεωρώ ότι μεταξύ δημοκρατών θα πρέπει να είναι δυνατόν να διεξαχθεί ένας επικοδομητικός διάλογος, ακόμη και αν δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία σε όλα τα θέματα, σε όλες τις λεπτομέρειες. Θέλουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε τη δική μας θέση, τη δική μας τοποθέτηση, να σας παρουσιάσουμε πώς καταλήξαμε στι δικές μας αποφάσεις και νομίζω ότι υπάρχει διάθεση ε, να εισακουστούμε. Συνεργαζόμαστε, όπως σας είπαμε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Προσπαθούμε ε, ως επιτοπλίστων να ε, εξεύρουμε και κοινέ λύσεις ακόμα και για αμφιλεγόμενα ζητήματα. Προσπαθούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε, ακόμα και αυτό δεν είναι εύκολο γιατί πολλές φορές οι απόψεις είναι διαφορετικές. Το προσπαθούμε πάντως η Ουγγρική κυβέρνηση και η Ουγγαρία θεωρεί ότι έχει υποχρέωση σε ό,τι αφορά την αρχή του κράτους δικαίου. Αυτό άλλωστε ανταποκρίνεται και στην ιστορία μας. Η κυβέρνηση και η ίδια η χώρα έχουν μια ιστορία στο πρόσφατο και το παλαιότερο παρελθόν που καταδεικνύει ότι η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου αποτελούν αξίες για τις οποίες πάντα αγωνίστηκε η Ουγγαρία. Αξίες τις οποίες πάντα προασπίστηκε η Ουγγαρία. Κοιτώντα πώς έχει η κατάσταση σήμερα στην Ουγγαρία, διαπιστώνουμε το εξή. Η τελευταία 25 ετία η ιδέα αυτή η αγάπη για την ελευθερία και για το κράτος δικαίου έχουν περάσει ίσως σε δεύτερη μοίρα, αν θέλετε, εν μέρη. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να αντιληφθούμε το τι συζητάμε. Μιλάμε για τα θεσμικά συμφέροντα, μιλάμε για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Έχουμε δημοκρατικούς θεσμούς οι οποίοι έχουν συχθεί στη χώρα μας. Όπως σας είπα, έχουμε ταχθεί υπέρ της δημοκρατίας και όπως σας είπα, τα τελευταία 25 έτη έχουν επιτευχθεί πολλά. Έχουμε ένα νέο σύνταγμα, έχουμε θέσει τα σημεία βάρους της πολιτικής μας και από την αρχή του 2010 στην Ουγγαρία έγινε διακριτή και η οικονομική κρίση αλλά και μια πολιτική κρίση. Κρίθηκε αναγκαίο να βρεθούν οι απαραίτητες ισορροπίες, οι οποίες είναι απαραίτητες σε μια δημοκρατία και σε αυτή συγκαταλέγονται διάφορα σώματα, όπως το Συνταγματικό Δικαστηρίο. Πάρα πολλές λοιπόν νομοθεσίες ε, εκδόθηκαν και αναλόγως προσαρμόστηκε και ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης όπως αναφέρθηκε. Η Ουγγαρία λοιπόν λειτουργεί ως δημοκρατία. Είμαστε ταγμένοι υπέρ της δημοκρατίας και τη δημοκρατία τη θέλουμε να τη τηρήσουμε. Εγώ ανήκω σε ένα κόμμα, το κόμμα του Πρωθυπουργού, που για πρώτη φορά μπήκε στο κοινοβούλιο, μάλλον που έβαλε στο κοινοβούλιο για πρώτη φορά με βουλευτή με καταγωγή Ρωμά. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω. Στο σημερινό λοιπόν κοινοβούλιο, στο κόμμα μας, έχουμε τους πιο πολλούς ε, συναδέλφους, βουλευτές με καταγωγή Ρωμά. Αυτό θέλω να τον τονίσω, αλλά ασφαλώς ε, είμαστε υπέρ και άλλων ομάδων, όπως είναι για παράδειγμα τα άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη δημοκρατία, ότι αισθανόμαστε όλοι ε, από κοινού υπεύθυνοι για όλες τις ομάδες και δεσμευόμαστε υπέρ αυτών. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την υπόθεση την οποία παρακολουθούμε και την οποία θίξατε σε ό,τι αφορά καταρχάς το Σύνταγμα. Συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία σημειώνει ότι η αρχή προστασία των δεδομένων θα πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητη. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Συμφωνούμε απόλυτα. Και ξεκινήσαμε σε ό,τι αφορά τον ορισμό των συγκεκριμένων προτύπων. Συμφωνήσαμε ως προς αυτά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι πλέον η αρχή προστασία των δεδομένων κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τώρα του δικαστέ και σε ό,τι αφορά την ηλικία συνταξιοδότησή του. Δεν είναι δικαστικό το θέμα, δεν είναι θέμα δικαιοσύνη, είναι μάλλον θέμα ε, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματο. Στην Ουγγαρία το σύστημα συνταξιοδότηση βρίσκεται υπό μεταρρύθμιση. Όντως, στην Ευρώπη αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης. Το ίδιο και στην Ουγγαρία. Θέλαμε λοιπόν να μην υπάρχουν διακριτικές με, ε, συμπεριφορές και να υπάρχει μια σύνδεση του ορίου συνταξιοδότησης των δικαστών με το γενικότερο όριο συνταξιοδότηση. Βρήκαμε λοιπόν ένα συμβιβασμό. Ελπίζω και πραγματικά πιστεύω ότι με το συμβιβασμό αυτό θα εξαλειφθούν όλα τα προβλήματα τώρα σε ό,τι αφορά το νόμο για τα μέσα ενημέρωσης. Η κυρία Επίτροπος ε, ανέφερε ότι το συνταγματικό δικαστήριο ε, επέκρινε πάρα πολλά στοιχεία της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης. Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση και βάσει της απόφασης του δικαστηρίου θα γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις της νομοθεσίας να εξασφαλίσουμε, να διαβεβαιώσουμε την Επίτροπο ότι θα γίνουν λοιπόν όλες αυτές οι αλλαγές και φυσικά όλα αυτά θα διαβιβαστούν και στο Συμβούλιο της Ευρώπης γιατί ε, τοποθετήθηκε και ε, υπέβαλε γνωμοδότηση σχετικά και το Συμβούλιο της Ευρώπης και όλες αυτές τις παρατηρήσεις λοιπόν κατά ανταπόκριση σε όλες αυτές τις ε, παρατηρήσεις θα διεξάγουμε τις σχετικές τροποποιήσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις στο θέμα αυτό και σίγουρα ασφαλώς θα λάβουμε υπόψη τις ε, απόψεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για να βρούμε μια σωστή λύση. Τώρα σε ό,τι αφορά την εξαρτησία της δικαιοσύνης, επεξεργαζόμαστε μία απάντηση στα ερωτήματα που μας τέθηκαν και εδώ είμαστε ανοιχτοί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρισκόμαστε σε ένα διαρκή διάλογο άλλωστε και θα ακολουθήσουν περαιτέρω πληροφορίε. Να προσθέσω όμω και κάτι άλλο, ιδιαίτερα συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά τον νόμο για, τις ενημερ... για μέσα ενημέρωση. Μιλήσατε για το ραδιόφωνο για το Club Radio. Μιλάμε για θέματα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Μιλάμε για θέματα διατήρησης, προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνη. Σας παρακαλώ λοιπόν στο σημείο αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε το σωστό δρόμο, δεν είναι πολιτικού τύπου οι αμφισβητήσεις μας, ε, οι σκέψεις που κρύβονται πίσω από την υπόθεση αυτή. Ελήφθη μια απόφαση και αυτό γίνεται χωρίς καμία οποιαδήποτε πολιτική πίεση. Ευχαριστούμε. Κύριε Αντιπρόεδρε Ναυράξης για την παρουσίαση της ουγγρικής ε, κατάστασης. Ως εκπρόσωπος της Ουγγρικής Κυβέρνησης μας εκθέσατε την κατάσταση. Σημειώνουμε όλες τις λεπτομέρειες και για την ίδια την ε, ΛΥΜΠΕ και προς χάρη των πρακτικών της σημερινής ακρόσης θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι παρόν εδώ ο η δικαιοκριμένη εκπρόσωπος ε, της κοινότητας των Ρωμά που εδώ και χρόνια το Ευρωκοινοβούλιο έχει μέλος της Σοσιαλιστικής ο ε, κ. Χαντριό Ραμίρε Σεγέρα, που ήταν ένα Ισπανό ε, σοσιαλιστή, εκπρόσωπο της κοινότητας Ρωμά και μάλιστα πρόεδρο για χρόνια της ε, ομοσπονδία των Κοινοτήτων Ρωμά τη Ισπανία. Και σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά για να εκφράσουμε και να αντιπροσωπεύσουμε, εκπροσωπήσουμε σωστά την ποικιλομορφία τη Ευρώπη. των ευρωπαϊκών λαών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούσαμε λοιπόν τι εισηγήσει και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει η συζήτηση. Θα ακούσουμε λοιπόν τι συμβολέ των συντονιστών. Σύμφωνα με την αριθμητική του εκπροσώπηση. Θα αρχίσουμε με το ΕΛΚ. Να σα θυμίσω ότι για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συζήτηση και να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερου ομιλητέ, θα ήταν καλό αν ο καθένα σα περιοριστεί σε δύο λεπτά για να υποβάλει τις ερωτήσεις του, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα δεύτερο γύρο μετά από τις απαντήσεις των μελών του Προεδρείου. Κύριε Μπουζουτήλ, έχετε το λόγο. Έχουμε πολλά προσωπικά αισθήματα λόγω της κατάστασης στην Ουγγαρία. Ωστόσο, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρασυρθούμε από τα συναισθήματα, αντί να κάνουμε αυτό που είναι λογικό και να βασιστούμε στα γεγονότα. Ας σας ε, παρουσιάσω τη θέση του ΕΛΚΑ για αυτό το θέμα. Καταρχήν, υποστηρίξαμε την πρόταση για διοργάνωση αυτής της ακρόσης, παρά το γεγονός ότι κυβέρνηση τη Ουγγαρίας είναι όπως όλοι γνωρίζουμε είναι από κόμμα μέλος του ΕΛΚ. Το υποστηρίξαμε διότι δεν έχουμε καμία δυσκολία να συνεργαστούμε πλήρως με οποιαδήποτε πρωτοβουλία ώστε να εξασφαλιστεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία και σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης. Δεύτερον, υποστηρίξαμε άμεσα και χωρίς κανένα δισταγμό την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξεκινήσει διαδικασίες κατά παράβαση κατά της Ουγγαρία στους τρει τομείς που αναφέρθηκαν και προσμένουμε το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών. Τρίτον, καλωσορίζουμε τις σαφείς δηλώσεις ε, των Ουγγρικών Αρχών διαστόματος του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας ε, στην Ολομέλεια του Σώματος και τώρα από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ότι οποιαδήποτε νομοθεσία που δεν είναι σύμμορφη προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα αλλάχτεί και θα εφηγραμμιστεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είμαστε πεπισμένοι πως οι Ουγγρικές Αρχές θα τηρήσουν αυτή τους τη δέσμευση διότι γνωρίζουμε πως ήδη πέρυσι το έκαναν όταν προέκυψαν προβλήματα προβλήματα με τον ε, νομοθεσία περί ΜΜΕ και κατόπιν αιτήματο τη Κομισιόν άλλαξαν όντω αυτή την νομοθεσία. Εμεί καλούμε την Επιτροπή να διερευνήσει πλήρω οποιασδήποτε ανησυχίε ανέφερε ο Αντιπρόεδρο και αυτό να το κάνει σε σχέση με την Ουγγαρία, αλλά και άλλα κράτη-μέλη τη Ένωση. Αλλά κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό που ε, ισχύει στην Ουγγαρία μπορεί να αντιστοιχεί σε μια κατάσταση του άρθρου 7 που κάνει λόγο για σαφή κίνδυνο σοβαρής παράβασης από πλευράς του κράτους, κάποιου κράτους μέλους των αρχών των αξιών της Ένωσης θα υπήρχε κίνδυνο σοβαρής παράβασης από την Ουγγαρία αν η Ουγγαρία δεν είχε δεσμευθεί για μεταρρύθμιση οποιαδήποτε νομοθεσία που είναι ασύμβατη. Όμως το έκπραξε, ε, δεσμεύθηκε και δεσμεύθηκε επανελειμμένος. Οπότε υποστηρίζουμε πλήρως τη θέση της Κομισιόν, αλλά εντόνως διαφωνούμε με την πολιτική χειραγώγηση και με κρίσεις που γίνονται πριν να ολοκληρωθεί η κατάλληλη διαδικασία. Αυτή η Επιτροπή και αυτό το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να μετατραπούν σε δημόσιο δικαστήριο για την Ουγγαρία, διότι αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Οι αβάσιμες καταγγελίες, οι κατηγορίες είναι ε, λανθασμένες, υποβαθμίζουν την θέση του γκρικού λαού και γι' αυτό δεν θα μας εντυπωσιάσει αν το αποτέλεσμα είναι αυξημένος ευρωσκεπτικισμός. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Μπουσούτιλ. Κυρία Κόνς, από πλευρά των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, θα μιλήσω και εγώ ουγγρικά, καθότι μιλάμε άλλωστε και για την Ουγγαρία. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Έλλη Κρούς, που ήρθε πραγματικά στην Επιτροπή μας. Θα προσπαθήσω να μην επισέλθω ε, στις λεπτομέρειες της νομοθεσίας, αλλά πιο πολύ στο πνεύμα της νομοθεσίας. Ε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, μιας και είναι εδώ και η Γενική Διευθύντρια και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και η Επίτροπος. Ελπίζω και στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά. Νομίζω ότι τα βασικά ε, θέματα είναι τα εξή. Το βασικό ζήτημα. Πώς θα συνεχίσουμε, τι θα γίνει στο μέλλον. Το θέμα λοιπόν είναι η ποιότητα της ε, Ουγγρικής Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι η Ουγγρική κυβέρνηση εφαρμόζει κατά γράμμα τα, τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό αποτελεί λοιπόν το πρώτο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Βλέπουμε λοιπόν, εξετάζοντας το θέμα αυτό, ότι υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ο κύριος Ορμπάν είπε πολύ υπερήφανα στην Ολομέλεια ότι από τότε που ε, εκλέχθη Πρωθυπουργό έχουν περάσει 300 νόμοι και ότι υπάρχουν, ε, ε, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στον τομέα της παιδείας και του καθεξής. Θα πρέπει να ρωτηθούμε κατά πόσο όλο αυτό όλοι αυτοί οι νόμοι προέκυψαν με δημοκρατικό τρόπο αυτός ο υψηλός αριθμός νομοθεσιών. Αυτό λοιπόν είναι, αυτή λοιπόν είναι ένα από τα ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω και έχω και άλλα ερωτήματα να θέσω. Δεν ξέρω κατά πόσο η κυβέρνησή μας ε, έχει πίστη και δεσμεύεται για την διαδικασία ενοποίησης. Ιδάλλως δεν μπορώ να φανταστώ πως έχουν προκύψει κάποιες από αυτές τις νομοθεσίες. αλλά όντως απέστειλε ερωτηματολόγια η, κυβέρνηση πριν από την ε, επεξεργασία του συντάγματος. Αλλά όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολλά προβλέχτηκαν τα οποία δεν ταιριάζουν για το σύνταγμα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε διατάξεις για το οικογενειακό δίκαιο και πρέπει να πω ότι υπάρχει και έλλειψη δικαιοσύνης. Μία συγκεκριμένη ερώτηση έχω να θέσω ιδιαίτερα προς την κυρία Γενική Διευθέντρια. Μιλήσατε για την υπηρεσία προστασίας των δεδομένων και για την ανεξαρτησία της υπηρεσίας αυτής. Ως τώρα, ο διαμεσολαβητής απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του πριν από τη λήξη των, της ε, περίοδου θητείας τους. Και τελικά ο, ε, ο θα επανέλθει στη θέση αυτή και αυτό θα το αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστήριο. Και εδώ τύφεται το θέμα της ε, τήρησης της νομοθεσίας, αν θέλετε, ε, στο γράμμα, του γράμματος της νομοθεσίας και του πνεύματος της νομοθεσίας. Και στο τέλος του έτους πέρασαμε κάποια νομοσχέδια τα οποία δεν κινούνταν απαραίτητα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κύριος Ναυρατσής. Ε, να σας ρωτήσω το εξής, γιατί δεν ε, αποδεχτήκατε πλήρως την κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού λέτε ότι είσαστε σε τόσο διαρκή επαφή με την Επιτροπή. Γιατί δεν ε, έχετε συμμορφωθεί ως τώρα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα και την νομοθεσία περισταθερότητας. Αν είσαστε λοιπόν τόσο πεπισμένοι ότι τα επιχειρήματα είναι σωστά, γιατί δεν πράτεται και αναλόγως. Γιατί, για παράδειγμα, περικόψατε τις αρμοδιότητες του συνταγματικού δικαστηρίου. Όλα αυτά πώς μπορούν πρακτικά να συγκυραστούν. Thank you very... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι κανένα μυστικό ότι εδώ και αρκετό καιρό η ομάδα των φιλελευθέρων ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να κινήσει διαδικασίες κατά τη Ουγγαρία με βάση το άρθρο 7 παράγραφος 1 της συνθήκης. Και ακούω συνεχώ ότι αυτό είναι κάτι ε, πολιτικά μεροληπτικό υποκειμενικό, ότι θα πρέπει να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάση και να δούμε τη συμπεριφορά της Ουγγαρίας. Θα ήθελα προς ενημέρωση να διαβάσω για όσους το γνωρούν ακόμη και το, το, για τον Επίτροπο Μπαρόζο, ότι η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το άρθρο 7, ανακοίνωση του 2003 που μιλούσε για σεβασμό και προαγωγή των αρχών που αποτελούν τις βάσεις της Ένωσης, ήδη στην ανακοίνωση του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 δεν περιορίζεται σε τομείς που καλύπτονται από την Ενωσιακή Νομοθεσία. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει όχι μόνο για παραβίαση των κοινοτικών αξιών στο, σε περιορισμένο τομέα, αλλά ακόμη και όταν παραβιαστούν δικαιώμα, δικαιώματα σε τομεί που έχουν αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη αποκλειστική, που είναι αυτόνομα. Επιπλέον, η ανακοίνωση αυτή λέει ότι με τον κίνδυνο του ε, σαφούς κινδύνου, εφανούς κινδύνου, το άρθρο 7 της συνθήκης δίνει ένα προειδοποιητικό μήνυμα σε ένα κράτος μέλος πριν την ε, υλοποίηση της επικίνδυνης κατάστασης. Και επίσης υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν την επαγρύπνησή τους εφόσον αυτός ο πιθανός κίνδυνος πηλεί το οικονομικό κοινωνικό περιβάλλον και για, όλη την περίοδο από τη στιγμή της εμφάνισης των συμπτωμάτων, ρατσισμού, ξενοφοβίας κλπ. Και από τη στιγμή που τα συμπτώματα αυτά έχουν γίνει ορατά. Το άρθρο 7 λοιπόν μιλάει για καθήκον, για χρέο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προασπίσει τι θεμελιώδει αρχέ και αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ξεχάσουμε λοιπόν αυτή την εθνικιστική προσέγγιση που τη βλέπω να ευδοκιμεί όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δηλαδή μια χώρα έχει αποκλειστική κυριαρχία για το τι κάνει εντό επικράτειάς της. Λάθος. Αν σε μια χώρα, όποια και αν είναι αυτή, κάτι πάει στραβά, αυτό επηρεάζει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε εδώ. Γιατί υπάρχουν πολλά πραγματικά περιστατικά που μας ε, υποχρεώνουν να δηλώσουμε ότι η κατάσταση στην Ουγγαρία έχει επιδεινωθεί σοβαρά. Η κυρία Λούνατζε για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Εκ μέρους ε, των Πρασίνων θα ήθελα να αποταθώ στον κύριο Μπουσουτήλ, τον συντονιστή του ΕΛΚ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και να του συστήσω να ακούει πρώτα, να ακούσει πρώτα τους προσκεκλημένους μας και τι θα μας πούν και μετά να λάβει μια απόφαση στην ομάδα για το άρθρο 7 και όχι από την αρχή, γιατί γι' αυτό γίνεται η ακρόαση. Και η ομάδα μας ζήτησε εφαρμογή του άρθρου 7 για να αξιολογήσουμε τι συμβαίνει στην Ουγγαρία. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την ακρόση. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε ε, Μπουσουτήλ. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε. Μην αρχίσετε τώρα να ανησυχείτε. Μετά θα λάβουμε απόφαση. Μην προδικάζετε. Τώρα, ως προς τους πρασίνους. Αυτά που ακούμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, τα νέα από την Ουγγαρία, είναι πολύ ανησυχητικά και ευχαριστώ την Επίτροπο Κρούς που διευκρίνησε ότι και για το θέμα του νόμου των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουμε ένα, μία μόνο έκφαση ενός ευρύτερου ε, φάσματος ανησυχιών και της ε, υπόνοιας ότι η Ουγγαρία παρεκκλίνει προς ένα πολιταρχικό, αυταρχικό καθεστώς που δεν έχει α, όμοιό του στην Ευρώπη. Σε, σε ό,τι αφορά κάτι που είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Σνόβατσης, ε, Είπατε σαφώς και ευχαριστούμε που το κάνατε ότι η ε, χώρα σας είναι προσιλωμένη στη δημοκρατία και ότι έχετε όλε τα απαραίτητα συστήματα ελέγχου και επιτήρηση για να το εξασφαλίσετε. Το είδαμε όμως και αυτό με τον Πρωθυπουργό σας. Άλλα λέτε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλα λέτε ε, στην πατρίδα σα. Χθε μόλι ο Πρωθυπουργό σα, ε, ο Όρμπαν, σε ένα συνέδριο του Φίντες χθες, αναφέρθηκε σε μια δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος στο Κούτσε το Σεπτέμβριο του 2009 που δήλωσε ότι για τα επόμενα 15-20 χρόνια ο διτός χαρακτήρας το, τον, της ουγγρικής πολιτικής με ισχυρό κυβερνών κόμμα και ισχυρή αντιπολίτευση θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ισχυρό κυβερνό κόμμα που θα είναι σε θέση να προσδιορίζει το εθνικό πρόγραμμα που σημαίνει ότι το κόμμα αυτό θα είναι το φίδες για τα επόμενα 15-20 χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος ε, του Πρωθυπουργού και του κόμματό σας. Οδεύεται προ ε, ένα ενιαίο ισχυρό κόμμα. Πού είναι λοιπόν η έλεγχη που κάνετε στην Ουγγαρία και η προσήλωση προς τη δημοκρατία. Έχετε ε, τον κύριο Ισαγγελέα, τον αρχηγό του ανώτατου δικαστηρίου, είναι μέλη του κόμματό σα. Το νέοι ε, δικαστική, ε, δικαστική του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο επικεφαλής του Γραφείου για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Έχετε ημετέρους στα πιο σημαντικά θεσμικά πόστα. Αυτή είναι η έλεγχη και αυτή είναι η εγγύηση για τη δημοκρατία. Checks and balances, αυτή η έλεγχη ε, για την εφαρμογή της δημοκρατίας σημαίνει ότι αν ένα κόμμα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων, τότε είναι που θα πρέπει να αναμίξει την αντιπολίτευση και να έχει συνομιλίες με την αντιπολίτευση. Και χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση και χρειάζεται πλουραλισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να ακουστεί και η άλλη φωνή. Τώρα, κεντρικό πεδίο ισχύω αυτό που ζήτησε ο Πρωθυπουργό σα στο συνέδριο του ΦΙΔΕΣ σημαίνει ε, κατεύθυνση προ ένα αυταρχικό καθεστώ, ε, το οποίο ε, στυλιτεύουμε όλοι. Θα θέλαμε να μα πείτε τι ελέγχου κάνετε, τι σεβασμό εξασφαλίζετε όταν το ΦΙΔΕΣ, το κόμμα σας, έχει μονοπολίσει ουσιαστικά όλα τα ισχυρά αξιώματα στη χώρα σας. Θα ήθελα να σας υπογραμμίσω τη σημασία που έχει η τήρηση του χρόνου. Γιατί είμαστε ήδη εδώ όλες ολόκληρες και έχουμε ακόμη πολλές ώρες μπροστά μας. Θα είναι πολύ μακριά αυτή η μέρα. Και έχουμε και πολλούς προσκεκλημένους στην δημόσια αυτή ακρόαση και κανονικά στις 6.30 πρέπει να τελειώσουμε. Η διερμηνία θα σταματήσει στις 6.30. Δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Γι' αυτό θα πρέπει να τηρούμε πιστά το χρόνο αγόρευσης. Η κυρία Μακιντάιρ της ε, ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Όποιο θέλει το λόγο, παρακαλώ, στον πρώτο κύριο ερωτήσεων να, να το δηλώσει από τώρα. Η κυρία Μακιντάιρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τίποτα αν δεν είναι προασπιστή των δικαιωμάτων. Η ομάδα μου πιστεύει ιδιαίτερα στην κυριαρχία κάθε κράτου μέλου και το δικαίωμα κάθε δημοκρατική χώρας να καθορίζει το σύνταγμά του και του νόμους του. Επίσης πιστεύουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τιμούν τις δεσμεύσεις τους ε, που έχουν αναλάβει στις ε, ευρωπαϊκές συνθήκες, όπως έχουν τεθεί θέματα για το δικαστικό θέμα, για το νόμο, για τα μέσα ενημέρωσης, ε, για το, την αρχή προστασίας των δεδομένων. Όλα αυτά μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Ωστόσο, η ομάδα μου θεωρεί ότι όλες οι ε, έρευνε θα πρέπει να γίνουν σε πνεύμα δικαιοσύνη και ισορροπία. Μόνο με συνεργασία θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στα σωστά αποτελέσματα. Ζητώ λοιπόν να μην αντιμετωπίζουμε την Ουγγαρία ω εχθρό, ως, αλλά ω μέλος της Ένωσης, τον οποίο θα πρέπει να εισακούσουμε και να βοηθήσουμε προκειμένου να προσαρμοστεί στις ε, ε, προδιαγραφέ. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώθηκε και η ακρόαση, όχι μόνο για να εξαπολύσουμε κατηγορίες, αλλά για να ακούσουμε και την Επιτροπή και την ίδια κυβέρνηση. Γιατί τα θέματα αυτά, ξέρετε, προκαλούν έντονα πάθη. Αλλά θα σας ζητούσα να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να διατηρήσουμε και ένα πνεύμα ισορροπίας, αν θέλετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τόνισε και έχει εντοπίσει ποιοι είναι οι τομεί όπου χρειάζεται προσαρμογή του συντάγματο και ελπίζουμε να ακολουθήσει δράση, ενέργεια από πλευρά τη ε, Ουγγρική κυβέρνηση. Θα πρέπει να περιμένουμε πρωτού το Κοινοβούλιο αναλάβει περαιτέρω δράση. Θα ξέρετε ότι είμαι νέο μέλο του Κοινοβουλίου και τα τελευταία έξι χρόνια έχω συνεργαστεί τακτικά στη Βουδαπέστη στο γραφείο μου με θέα το Δούναβη και αγαπώ ιδιαίτερα την Ουγγαρία και το λαό της Ουγγαρίας. Θαυμάζω ιδιαίτερα τον τρόπο εξυγχρονισμού και ανάπτυξης της Ουγγαρίας, διατηρώντας παράλληλα την κληρονομιά της. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να μάθω την ε, γλώσσα. Το μόνο που έχω μάθει είναι τη λέξη «κέσονα» που σημαίνει «ευχαριστώ». Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τις παρουσιάσεις σας σήμερα και θα ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε ποια είναι πραγματική, το πραγματικό επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ σας, επαφών μεταξύ σας και, κα, και κατά πόσον υπάρχει όντως μεγαλύτερη κατανόηση από αμφότερες πλευρές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρες. Και τώρα η κυρία Βερζιάτ για την ΚΟΕ. Ναι, με συγχωρείτε, δεν έβρισκα το μικρόφωνο. Εγώ ήθελα να συμφωνήσω με τους φιλελεύθερους και πράσινους συναδέλφους όσον αφορά το επίμονο αίτημα εκπόνηση έκθεσης επί τη βάση του άρθρου 7 από πλευρά του Κοινοβουλίου, αλλά επειδή πολλά υπόθηκαν δεν θα επαναλάβω. Θα προσπαθήσω μόνο να δώσω κάποια παραδείγματα που εμένα μου δημιουργούν πρόβλημα και που δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής. Το θέμα της προστασίας των μειονοτήτων ε, είναι προβληματικό. Και έχω την εντύπωση μάλιστα ότι ο ορισμός που δίνεται από, την, από το νέο Ουγγρικό Σύνταγμα στην υπηκότητα, στην εθνικότητα, δεν μπορεί παρά να τονίσει τις εντάσεις στην περιοχή ανάμεσα στις μειονότητες. Πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Επιπλέον διάβασα, αλλά σίγουρα δεν είναι βάσιμο αυτό, ότι είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα απέναντι στους ε, άστεγους ότι μέτρα ποινικοποίησης είχαν ψηφιστεί με πολύ μεγάλα πρόστιμα που προβλέπονται για ανθρώπους που έχουν ε, την ατυχία να μην μπορούν να ζήσουν εξυπροπώ. Τα πρόστιμα είναι τόσο βαριά που δεν έχουν καμία δυνατότητα να πληρώσουν τα πρόστιμα αυτά και άρα καταδικάζονται σε φυλάκιση. Έχω την εντύπωση πως μια τέτοια αντίληψη περί προστασίας των ε, πιο ενδεών είναι αντίθετη με τις αρχές, ε, τις αξίες της ευρωπαϊκές, που τις λέμε εμείς ευρωπαϊκές, αλλά μάλλον είναι καθολικές. Έπειτα υπάρχουν διάφορε διατάξει που εγώ θα μπορούσα να σχολιάσω από πολιτική άποψη, αλλά οι πολιτικέ επιλογέ είναι αυτέ που είναι και καθο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 έχουν ανυψωθεί σε επίπεδο συνταγματικών αξιών, όπως για το γάμο για παράδειγμα. Μπορεί να, έχουμε, να κάνουμε πολιτικές επιλογές, δεν έχουμε τις ίδιες πολιτικές επιλογές, αλλά αυτός ο ορισμός του γάμου δεν έχει θέση σε ένα σύνταγμα. Όταν λέει ότι ένας γάμος δεν μπορεί να συναυθεί παρά μόνο μεταξύ ανδρός και γυναικός στο, μέσα στο σύνταγμα, αυτό ε, δημιουργεί νομικό πρόβλημα στις αξίες που εμείς υποστηρίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ίδιο και για την άμβλωση, γιατί θεωρείται ότι το έμβριο είναι άνθρωπος και αυτό αναφέρεται στο ίδιο το σύνταγμα. Το ίδιο και για την ισόβια κάθεξη. Όλα αυτά, νομίζω, και έχω σχεδόν τελειώσει, Πρόεδρε, μετατρέπουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στενές χριστιανικές αρχές που, αξίες που νομίζω δεν μπορούν να αναγνωρίζονται μέσα στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καθολική τους ε, έννοια όπως αυτές εννοούνται εδώ σε αυτό το σώμα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του EFT, ο κύριος ο δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην ε, λεπτομερή σας ε, παρουσίαση, Επίτροπε Κρούς, στην ουσία κάνατε μια ιερά εξέταση απέναντι στην Ουγγρική κυβέρνηση αναφερόμενη σε πολύ με λεπτομερή προγράμματα και εισάγοντας αμφιβολίες. Εγώ προς αυτό διαρωτώ με λοιπόν αν η Κομισιόν στην ε, δράση της για εξέταση της υποψηφιότητας της Τουρκίας όπου αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο βάσιμα και πολύ άριθμα τα περιστατικά θα χρησιμοποιήσει τα ίδια κριτήρια και θα τα παρακολουθήσει με την ίδια προσοχή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το ειδικό μας σπίτι και με μια χώρα που με περηφάνεια ε, ε, διεκδικεί την ε, γέννησή της ε, το 1848 και ε, περήφανα υψώνει την σημαία της ελευθερίας. Και μάλιστα εντάξει να εξετάσουμε το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε να κάνουμε τη δημοκρατία, την κυριαρχία και την αρχή της επικουρικότητας που καθιστούν εξαιρετικά σημαντική τη σημερινή συζήτηση. Δημοκρατία. Εγώ διαβάζω στις εφημερίδες από ανεξάρτητα μέσα ότι η γκουρική κυβέρνηση κάνει ένα δημοψήφισμα σε όλες τις οικογένειες για 12 ζητήματα, 12 σημεία μάλλον, πριν να νομοθετήσει. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει ως υπόδειγμα αυτή την κυβέρνηση και να ρωτήσει κάμια φορά και τους Ευρωπαίους πολίτες για σημαντικά θέματα. Το κάνει ποτέ. Ε, ε, ερωτηματικό αυτό για τη δημοκρατία. Και έπειτα υπάρχει και το θέμα της επικουρικότητας που τίθεται, για παράδειγμα, για το ζήτημα που αναφέρθηκε του ραδιοφωνικού σταθμού. Υπάρχει ένα ζήτημα όπως αναφέρθηκε, υπάρχει μάλλον υπόθεση στα δικαστήρια. Νομίζω λοιπόν πως είναι απίστευτο να τίθεται σε, στην, στην προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα θέμα τέτοιο διοικητικό ενώ είναι ένα απλό θέμα το οποίο θα πρέπει κάθε κυρίαρχο κράτο να το αντιμετωπίζει μόνο του. Και έπειτα το θέμα της, κυριαρχίας, τη εθνικής κυριαρχίας είναι αυτή ασύμβατη με το κοινοτικό δίκαιο. Πού είναι τα όρια. Γιατί με μεγάλη εξωπρέπεια λέει αυτή η χώρα. Έχουμε και κρατούμε την κυριαρχία μας. Και υπάρχει και η εξή αμφιβολία. Ίσως η αντίστασή τη στι δυνατέ δυνάμει μπόρεσε να βρει την σταθερότητά της στην οικονομική και την χρηματοπιστωτική χωρίς να υποστεί τους φρικτούς κανόνες του, της διεθνούς ε, ε, οικονομικής εξουσίας ε, το καθιστά αντιπαθητική σε διάφορες άλλες δυνάμεις. Ευχαριστώ. Θα σας ειδοποιήσω ότι η ώρα έχει πάει 3 και 4 και έπρεπε ήδη να περάσουν, έχουμε περάσει στο δεύτερο πάνελ. Σε καμία περίπτωση φυσικά δεν θα τα καταφέρουμε. Ωστόσο έχουν έρθει κάποια μέλη του δεύτερου πάνελ, γιατί το χρονοδιάγραμμα έλεγε ότι θα ξεκινήσουν στις 3. Ε, Έχω ένα κατάλογο των ομιλητών που θέλουν να πάρουν το λόγο για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Να προτείνω η Επίτροπος, η Γενική Διευθύντρια και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αν δεν έχετε αντίρρηση, να δώσουμε 1,5 λεπτό για τους βουλευτές που είναι ήδη στον κατάλογο και κλείνει η λίστα, 8 μέλη, 8 βουλευτές, προκειμένου να απαντήσει και, ε, να απαντήσει το πρώτο πάνελ, πρωτού περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Αν δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Θα ακούσουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. 1,5 λεπτό θα είμαι αυστηρός. Πριν πάρετε το λόγο, σας παρακαλώ κοιτάξτε τις σημειώσεις σας, τα χαρτιά σας, προκειμένου να μην ε, τα διαβάσετε και να μην ξεπερνάτε το όριο χρόνου, γιατί το λέω εγώ 1,5 λεπτό, αλλά τελικά πολλοί μιλούν 2,5 λεπτά. Δεν πρέπει να προλάβουμε. Σας παρακαλώ. Η κυρία Γιάννοκα. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και την Επίτροπο για την ομιλία της και την παρουσίασή της. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση και να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Σε ό,τι αφορά την προστασία των μειονοτήτων στην Ουγγαρία. Πριν από μερικά χρόνια, τους, οι, Ούγγροι, οι, τσιγκάνοι, οι υπέστησαν πολλές επιθέσεις και σωματικές και μάλιστα πρόσφατα είχαμε απόπειρες εκφοβισμού των Ρωμά στην Ουγγαρία. Ε, μάλιστα η κυβέρνηση ε, Φίντες ενέκρινε μια νομοθεσία που απαγορεύει τον εκφοβισμό των μειονοτήτων και έτσι σταμάτησαν οι προσπάθειες εκφοβισμού κατά των ε, Αθηγάνων. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε τους Αθηγάνους με τους Ρωμά στην Ουγγαρία και στην Ευρώπη. Πολλά άλλαξαν τα τελευταία δύο χρόνια στην Ουγγαρία, ακριβώς χάρη στην κυβέρνηση του Φίδες έχουμε επιτέλους μια στρατηγική προστασία στον Ρώμα χάρη στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή προστάτευσε ε, την, την, ε, τις μειονότητες ε, που ούτως έως και πριν από την κρίση είχαν πρόβλημα. Η στρατηγική αυτή, μάλιστα που έχει υπογραφεί από 27 χώρες μέλη υπέρ των μειονοτήτων, είχε υποβληθεί με, από την Ουγγαρία. Ήταν, ήταν ουγγρική πρόταση και η Ουγγαρία είναι ίσως η μόνη χώρα που την εφαρμόζει αποτελεσματικά. Και νομίζω ότι την Ουγγαρία θα πρέπει να τη μιμηθεί και η Ρουμανία. Πρόβλημα με τους Αθηγάνους και Ρωμά έχουν και άλλες χώρες, Ιταλία, Γερμανία. Θα πρέπει και αυτές οι χώρες να πραγματοποιήσουν αποφασιστικά βήματα προκειμένου να επιτρέψουν στις μειονότητες και στην Ρωμά μειονότητα μεταξύ άλλων να βρουν το δρόμο τους προς την οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να προστατεύσουμε τις μειονότητες και να περιορίσουμε τις εξτρεμιστικές ε, εκφάσεις. Η κυρία Μποσκούρτ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση έχω να απευθύνω στον εκπρόσωπο της Ουγγρικής Κυβέρνησης, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Άκουσα ότι η συζήτηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό το, της Ουγγαρίας, ότι στην Ουγγαρία περιγράφηκε ως ε, νίκη του Ουγγρου Πρωθυπουργού. Πειράζει το ότι παρουσιάζεται έτσι στα μέσα ενημέρωσης. Όχι. Αλλά αυτό που πειράζει είναι ότι δεν υπάρχει πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης και δεν παρουσιάζεται καμία άλλη άποψη. Σε ένα έτο ε, πέρασαν γρήγορα, γρήγορα 230 ε, νόμοι, 99 μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Μπορεί να θεωρείτε την αντιπολίτευση ενοχλητική, αλλά εκπροσωπεί ένα τμήμα του γκρικού πληθυσμού, ξέρετε, όπως και εσείς. Σε μια δημοκρατία, επίσης, ξέρετε, ε, θα πρέπει να υπάρχει και ο υπεύθυνο η υπηρεσία προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι βασικό πρόκειται να δώσετε την απόλυτη ανεξαρτησία στην υπηρεσία αυτή, γιατί και αυτό είναι πολύ βασικό για τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισελ, 1,5 λεπτό. Oui. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επίτροπο Νέλη Κρούς γιατί ήταν πολύ εύστοχα τα σχόλιά της ε, και τιμούν την Επιτροπή. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος της. Ήθελα να απευθυνθώ στον συντονιστή του ΕΛΚ. Και να του πω ότι δεν με συγκίνησε καθόλου, απλώς με ανησύχησε. Για να μην πω ότι με συγκλώνησε κιόλα. Με σοκάρατε κύριε συντονιστά με, αυτό που, με αυτή τη στρατηγική ε, που ακολουθείτε με το ΕΛΚ κατά της Ουγγαρίας, σαν να μην συμβαίνει τίποτα δηλαδή, σαν να είναι μια μπανάλ κατάσταση ε, και ενώ βλέπουμε ότι η δημοκρατία, και ξέρουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι η τυραννία της πλειοψηφίας, δεν έχει ε, το κυβερνών κόμμα ή η πλειοψηφία να περιθωριοποιεί την αντιπολίτευση, αλλά χρέος έχει να τη σέβεται. Κάτι που δεν ε, φαίνεται ότι γίνεται. Τρίτη παρατήρηση. Φυσικά και συντρέχουν όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 7. Φυσικά και δεν πρέπει να περιμένουμε να διερευνήσουμε περαιτέρω τα κριτήρια και τα πραγματικά περιστατικά, γιατί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 7 και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Προσπαθείτε τώρα να κερδίσετε χρόνο εξηγώντα μας ότι ε, δεν είναι και πολύ σοβαρή κατάσταση, ε, η Ουγγρική κυβέρνηση είναι καλοπροαίρετη και ούτω καθώς. Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο. Καταλαβαίνω ότι μερικέ κυβερνήσει μπορεί να μπερδεύτηκαν ή να έσπευσαν. Αυτό που με ανησυχεί είναι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά τη κυβέρνηση. Γιατί όταν έρχεται εδώ ο κύριο Ορμπάν, μα τα λέει όλα πολύ χαλαρά και επίκη. Όταν πηγαίνει όμως στην Ουγγαρία τα λέει πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτό είναι εύλογο να κλονίζει την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχουμε προς λοιπόν την Ουγγρική κυβέρνηση. Ανάμιση λεπτό κύριε Λουκαρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να χαιρετήσω την παρουσίαση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης και της Επιτρόπου. Μιλάμε για θέματα οικονομικά, θέματα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής, μιας και συζητάμε θέματα παγκοσμιοποίησης ε, η αλλαγή είναι κάτι το αναγκαίο, ακόμα και στην Ουγγαρία. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θέλουν να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον οι πολιτικοί λόγοι, οι πολιτικές αιτίες που αναφέρονται στέκουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και Ερωτώ λοιπόν τον Αντιπρόεδρο της ε, Ουγγρικής Κυβέρνησης. Ποια είναι η θέση της Ουγγρικής Κυβέρνησης, ποιες είναι οι σχέσεις με την αντιπολίτευση, με τους σοσιαλιστές, προκειμένου να σχηματίσουμε μια σαφή εικόνα, προκειμένου να κατανοήσουμε ποιες είναι οι πηγές, οι αιτίες μιας τέτοιας απόφασης. Κατά δεύτερον, ποια ήταν η εθνική αντίδραση, μάλλον ποια ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράστηκαν και εξαπολύθηκαν τέτοιες κατηγορίες. Θα μπορούσατε λοιπόν εν συντομία να μας αναφέρετε ποια ήταν η επίσημη ανταπόκριση της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητή Επίτροπο, αξιότιμη Αντιπρόεδρε τη κυβέρνηση. Μιλήσαμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα να θέσω άλλο ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα στην Ουγγαρία, το θέμα της κατάστασης των ετούντων άσυλο. Η Επιτροπή του Ελσίνκη διαπίστωσε πολλές φορές παραβιάσεις ε, φυλακίσεις ε, ανηλίκων, οικογενειών. Το 2010, το Δεκέμβριο του 2010, εισήχθη ένα καινούριο σύστημα ασύλου στην Ουγγαρία και διαπιστώθηκαν παραβιάσεις ε, των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εγώ από τη Γερμανία έχω ζήσει ότι η Ουγγαρία ήταν χώρα υποδοχής ε, των προσφύγων. Αυτό θα ήθελα να ξαναγίνει. Πώς λοιπόν θεωρείτε, ποια είναι η στάση σας για την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποια προοπτική υπάρχει να εφαρμοστούν πλήρως αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σόκουρ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, θα μιλήσω γκρικά. Ακούστε δεν μπορώ να λάβω σοβαρά υπόψη τις κατηγορίες των σοσιαλιστών και φιλελευθέρων. Είναι αβάσιμες, για να μην πω και γελίες αυτές οι κατηγορίες. Γιατί το 2006 ε, ξυλοκοπούσαν τους, Ευρωπα... τους ε, Ούγγρους πολίτες στην Ουγγαρία, κανένας ε, φιλελεύθερος ή σοσιαλιστές ε, δεν διαμαρτυρόταν. Το, το, ράδιο, το ραδιόφωνο κλαμπ δεν έκλεισε. Μάλιστα, ε, ρωτάτε γιατί σε μια χώρα που παραβιάζονται οι κανόνες των γλωσσών κλείνουν, κλείνουν κάποιους ε, ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έκλεισε ένας ε, ραδιοφωνικός αγγλικός σταθμός και ξέρετε για ποια χώρα μιλάω. Αυτό όμως δεν τα λέτε τίποτα. Άλλωστε δεν επιτράπει είσοδος του Προέδρου της Ουγγρικής Δημοκρατίας στη χώρα αυτή και κανένας τότε δεν είπε τίποτα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά λοιπόν. Στην Ουγγαρία έχουμε πολλέ μειονότητε. έχουμε πολύ τακτικέ επαφέ μαζί του. Καμία μειονότητα δεν αισθάνεται φόβο. Ενώ στι γειτονικέ χώρε της Ουγγαρίας εκεί είναι που οι μειονότητε ε, ε, φοβούνται. Αλλά κανεί δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Ευχαριστώ κυρία Ιντβελ. The... Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο σύντομε ερωτήσει προ τον αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση. Καταρχήν, με εξέπληξε το γεγονός ότι έμαθα ότι κατά μέσο όρο 2.500 Ούγγροι πολίτες ε, ζητούν άσυλο στον ε, Καναδά, κυρίως Ρωμά. Θα ήθελα να μου δώσετε την εξήγηση αυτού του φαινομένου. Δεύτερη ερώτηση. Ε, από ό,τι κατάλαβα, ένας ε, συνδυασμός μετα... νομοθετικών μεταρρυθμίσεων με την οικονομική κρίση οδήγησε στο ότι πολλά δημόσια σχολεία δόθηκαν από τους Δήμους στην Καθολική Εκκλησία. Αυτό ήταν ε, δυνατόν και παλιότερο. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά που είναι γραμμένα σε ένα δημόσιο σχολείο, από τη μια μέρα στην άλλη, βρίσκονται να φοιτούν σε ένα καθολικό σχολείο όπου ισχύουν καθολικοί κανόνες, κανόνες της Καθολικής Εκκλησίας, να δίνονται διαφορετικά, να κάνουν καθημερινά την προσευχή τους και μάλιστα πολλοί διευθυντέ σχολείων αντικαταστάθηκαν από διευθυντέ σχολείων που ακολουθούν το καθολικό δόγμα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κύριος Άντερ, τελευταία ερώτηση, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Εμένα με ενοχλεί το εξή. Δεν με ενοχλεί αυτό το διτό, αν θέλετε, αυτή η υποκρισία στη γλώσσα και στις δηλώσεις. Άρα αυτά τα διπλά μέτρα και σταθμά. Ο καθένας λέει αυτά που τον συμφέρουν, αυτά που τον ευνοούν. Όλα αυτά τα οποία ε, συζητήθηκαν είχαν ήδη συζητηθεί με την αντιπολίτευση και με τους σοσιαλιστές προς, τα ποια κατεύθυνση, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι μεταρρυθμίσει. Φυσικά. Το Κοινοβούλιο είναι τελικά το αρμόδιο σώμα για την νομοθεσία αυτή. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Τώρα, σε ό,τι αφορά θέματα δικαιοσύνη και σε ό,τι αφορά θέματα διοικητικά της δικαιοσύνης. Κυρία Γκέντς, να σας ε, διαβεβαιώσω ότι ο πρόεδρος ε, του Ανώτατου Δικαστηρίου υπόκειται σε πολύ αυστηρούς κανόνες. Αυτό δεν ίσχυε στο παρελθόν. Πλέον είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες αυτοί. Και αυτό ισχύει για όλο το δικαστικό σώμα. Θα πρέπει να πληρούν υψηλές προδιαγραφές. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Γιατί όπως σας είπα, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχε πολύ πιο πολλές ελευθερίες στο παρελθόν. Και έγινε και μια ολόκληρη συνδιάσκεψη με διαβούλευση σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και θέματα α, κατανομής των εξουσιών συζητήθηκαν και υπήρχε λοιπόν συνένεση και μετά από τη συνένεση αυτή προτάθηκαν οι σχετικές τροποποιήσεις. Το Κοινοβούλιο που κινούμε το Συνταγματικό Δικαστήριο ε, συμφώνησαν και ανέκριναν την διαδικασία. Ο Πρόεδρος ξέρω ότι δεν είναι εύκολο γιατί ήταν έντονε ε, οι συζητήσει και ήταν ε, και πολλέ ερωτήσει. Μια και ακούσαμε δύο γύρου ερωτήσεων. Δεν θα είναι εύκολο να απαντήσετε, αλλά είμαι βέβαιο ότι τα αξιότιμα μέλη του πάνελ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να απαντήσουν ε, άμεσα στι ερωτήσει που άκουσαν. Και να μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσει. Η κυρία Κρούς να ακολουθήσουμε την ίδια σειρά όπως και στο πρώτο γύρο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέντε ερωτήσεις τέθηκαν προς ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να τις συνδυάσω, να τις συγκεράσω για να απαντήσω. Μία ερώτηση που προβλημάτισε πολλούς βουλευτές είναι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όλα τα κρατημέλη και τα δυναμει κρατημέλη. Η απάντηση είναι καταφατική. Σίγουρη η αντιμετώπιση είναι ίση προς όλους. Δεύτερη ερώτηση. Το άρθρο 7. Το άρθρο 7 μιλά για τον, κατάλληλο, καταλληλότερο τρόπο ε, αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και διαδικασία επιπαραβάση στόχο έχει να πει στην Ουγγαρία να ευθυγραμμίσει το εθνικό της δίκαιο με το κοινοτικό δίκαιο πριν να προσφύγουμε στο δικαστήριο, για να μην χρειαστεί να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Αλλά συνεχίζουμε την επαγρύπνηση. Και αν υπάρξουν περαιτέρω ανησυχίες ή αν δεν διασκεδαστούν οι ανησυχίες μας, θα δούμε και, θα δούμε και άλλους τομείς της ε, νομοθεσίας και το πώς ε, ε, εφαρμόζει ποιο είναι το νομικό πλαίσιο της Ουγγαρίας και αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του 7 θα αναλάβουμε δράση. Σε ό,τι αφορά τους Ρωμά. Αν σας ενδιαφέρει θα μπορούσα να ζητήσω από, το, από ένα μέλος του της Συμβουλευτικής μου Επιτροπής που πρόσφατα πήγε για προσωπικούς λόγους στην Ουγγαρία και σχημάτισε εντύπωση για το τι συμβαίνει εκεί. Μπορώ να σα στείλω γραπτή, απάντηση, ε, γραπτή ενημέρωση. Δεν είναι συγκινησιακά φορτισμένο, δεν είναι μεροληπτικό. Ένα απλό άνθρωπο, πολύ αντικειμενικός, που συγκέντρωσε πληροφορίε και εντυπώσει από προσωπικό ταξίδι στην Ουγγαρία. Και τέλο θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα μία απάντηση από τον Αντιπρόεδρο της Ουγγρικής Κυβέρνησης. Η Ουγγρική Κυβέρνηση ρητά και διαφανώς ε, θα ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης μία εκτενή και περιεκτική γνωμοδότηση ό,τι αφορά την συμβατότητα της ε, νομοθεσίας περί ε, μέσω μαζικής ενημέρωσης και την εφαρμογή της με τρόπο που να ε, τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές και την, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και η δεύτερη ερώτηση, επίσης σημαντική, οι ουγγρικές αρχές, η, ουγγρικές η ουγγρική κυβέρνηση δέχονται και εφαρμόζουν τις θα δεχθούν και θα εφαρμόσουν τις συγκεκριμένε συστάσει του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αν η απάντηση και στις δύο ερωτήσεις είναι απερίφραστο ναι, θα θεωρήσω ότι αυτή η συνάντηση έχει πραγματικά μεγάλη επιρροή στη δημοκρατία στην Ευρώπη. Η Γενική Διευθύντρια κυρία Λεμπάγη. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το κεντρικό ερώτημα που ετέθη στον τομέα της δικαιοσύνης είναι πού οδεύομαι. Πολύ σημαντικό θέμα. Διότι ως Επιτροπή εμείς αναζητούμε την πλήρη συμβατότητα της εγκρικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή. Εμένα με ενθάρρυναν οι δηλώσεις του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, ωστόσο Όλα αυτά θα πρέπει πλέον να μετατραπούν σε συγκεκριμένες νομοθετικές τροπολογίες έτσι ώστε η ουγγρική νομοθεσία να συμμορφωθεί πλήρως με την ευρωπαϊκή περί αρχών ε, προστασίας των δεδομένων που αναφέρθηκε, θέμα που αναφέρθηκε από πολλούς από εσά και είναι σημαντικό τομέα. αλλά και το θέμα του δικαστικού τομέα και της νομικής προστασίας. Αυτά, μαζί με την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου, που είναι ένα στοιχείο κλειδί για τη δημοκρατία, θα πρέπει πλέον να τροποποιηθεί και ευχόμεθα οι ουγγρικές αρχές να μπορέσουν να απαντήσουν στα ερωτήματα και στις τροποποιήσεις που ζητήσαμε. Οι προθεσμίες είναι πολύ σύντομες, 17 Φεβρουαρίου, την επόμενη εβδομάδα. Και θα θέλαμε να έχουμε πολύ συγκεκριμένες δράσεις σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ, κυρία Λεμπάη. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος, κύριος Ναυράξης, θα κάνει ό,τι μπορεί για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ετέθησαν στην Ουγγρική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν. Κάποια από αυτά θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω άλλωστε. Με ρωτήσατε αν και κατά πόσο ήμασταν σε επαφή με το Συμβούλιο της Ευρώπης και κατά πόσον ε, ε, συμμορφωθήκαμε με τις συστάσεις του. Να σας πω ότι η απάντηση είναι καταφατική. Δεν θεωρούσαμε ότι πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλε κριτικέ, ε, όπω σα είπα, πάντα ήμασταν σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θεωρούσαμε ότι το θέμα του διαμεσολαβητή πρόκειται να ξανατεθεί. Όπω και να έχει, προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε για να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων και σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματο, ε, σε ό,τι αφορά το ανώτατο δικαστήριο, σε ό,τι αφορά το συνταγματικό δικαστήριο τώρα. Οι θέσει είναι. Οι απόψει είναι διχασμένε και θα μπορούσαμε επί ώρες να το συζητάμε το θέμα. Τα συζητήσαμε όλα αυτά εκτενώ όμω. Και όντω. Διαγράφησαν κάποιες από τις ρήτρες που αναφέρατε, όντως, αλλά αυτό έγινε μετά από συνένεση οι αρμοδιότητες του συνταγματικού δικαστηρίου σε καμία περίπτωση δεν περιορίστηκαν, αντιθέτως διευρύνθηκαν, κυρία Λούνατσεκ. Με κατηγόρησε ότι μιλώ υποκριτικά και ότι άλλα λέω εδώ και άλλα λέω αλλού. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Προσπαθώ να σας πω, να σας λέω ακριβώς τα ίδια που λέω και στη Βουδαπέστη. Σας διαβεβαιώ. Σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες τώρα. Για τον Πρωθυπουργό. Δήλωσε απλά ότι το κυβερνητικό κόμμα, το ΦΙΔΕΣ, επρόκειτο να είναι στο επίκεντρο και τώρα που υπάρχει κυβέρνηση του ΦΙΔΕΣ και του KDNP, Ασφαλώς και υπάρχει αντιπολίτευση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ε, στο δεξί τμήμα του πολιτικού φάσματος. Προσπαθούμε να μείνουμε στο κέντρο. Επίσης, μια άλλη κατηγορία που ακούσαμε ήταν ότι δεν υπάρχει πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης. Εγώ διαφορετικά πράγματα έχω ακούσει. Και σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει απόλυτο απόλυτος πλουραλισμός ε, στον έντυπο τύπο, στο ραδιοφωνικό φάσμα. Ανεξάρτητα από την μορφή της έκφρασης, ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του και ραδιοφωνικός ε, σταθμός Club Radio. Δεν ήταν μοναδικός σταθμός της αντιπολίτευσης, δεν μπορούμε να τον ρίσουμε έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μοναδικός σταθμός. Υπάρχουν διάφορα μέσα ενημέρωσης ε, στην Ουγγαρία που βρίσκονται ε, στο αριστερό μέρος του φάσματος του πολιτικού και ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Τώρα να πω δύο λόγια για τις μειονότητες. Να παραθέσω το εξής τμήμα από το Σύνταγμά μας. Στο άρθρο 29 αναφέρεται ότι οι μειονότητες αποτελούν ε, τμήμα του κράτους της Ουγγαρίας και ότι ε, απολαμβάνουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα όπως οι Ούγγροι πολίτες και με τον ίδιο τρόπο ακριβώς υπερασπίζομαστε τα δικαιώματά τους. Έχουν το δικαίωμα να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομά τους και υπό τη συλλογική έννοια έχουν το δικαίωμα του πολιτισμού τους και έχουν το δικαίωμα να διδάσκονται τη γλώσσα τους. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να σχηματίζουν τοπικές και εθνικές αντιπροσωπείες. Οι λεπτομέρειες τώρα ρυθμίζονται σε έναν ε, σχετικό νόμο. Έχουμε τρεις ε, βασικές εθνικές μειονότητες. Και όπως σας είπα, ισχύει το σύστημα αυτό που σας ανέφερα. Οι μειονότητες αυτές σχηματίζουν ενώσεις ε, εκπροσώπησης. Αυτό το σύστημα λειτουργεί μια χαρά και πρόκειται να συνεχίσει μια χαρά και στο μέλλον. σε ό,τι αφορά τους άστεγους τώρα. Αποφασίσαμε στην κυβέρνηση ότι θα ε, δημιουργηθούν καταλήμματα για τους αστέγους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά τέτοια καταλήμματα τα οποία θα πρέπει να οικοδομηθούν. Πρόκειται για μια υπηρεσία που προσφέρει η κυβέρνησή μας. Δεν θέλουμε ο κόσμος αυτός ε, να εκτίθεται σε θερμοκρασίες μείον 15 βαθμούς Κελσίου, όπως επικρατούν αυτή τη στιγμή στην ε, Ουγγαρία. Και σε κάθε περίπτωση έχουν το δικαίωμα να κινούνται ελεύθερα, να μετακινούνται ελεύθερα. Τώρα, η σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχει συνένεση που και που, πολύ συχνά και αυτό συχνά με το αναφέρουμε, ότι υπάρχουν που και που και σημεία στα οποία συμφωνούν η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση. Αλλά ασφαλώς υπάρχουν και πάρα πολλά σημεία στα οποία δεν συμφωνούν. Το κόμμα μας και ο αρχηγός του κόμματος, για παράδειγμα, πρόσφατα δήλωσε ότι την Άνοιξη πρόκειται να ε, διοργανωθεί μια διαβούλευση πέντε κομμάτων σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα. Έχουμε τρία κόμματα αντιπολίτευση και το μεγαλύτερο κόμμα τη αντιπολίτευση, οι σοσιαλιστέ, ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στι διαπραγματεύσει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν τα άλλα δύο κόμματα τη αντιπολίτευση. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα γίνει ε, στι διαπραγματεύσει. Αν κάποιο λοιπόν δεν επιθυμεί να συμμετάσχει, δεν μπορούμε να τον εξαναγκάσουμε ασφαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν ξέχασα να απαντήσω σε κάποιε λεπτομέρειε. Λυπάμαι. Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί δεν απαντήσετε στι ερωτήσει τη κυρία Κρού. Ε, είστε πρόθυμο να συνεργαστείτε πλήρω ε, με το Συμβούλιο τη Ευρώπη και να εστερνιστείτε και να εφαρμόσετε τι συστάσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Αυτό θα είναι πραγματικά χρήσιμη συμβολή στη δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτά που είπα δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Εμείς στην Ουγγρική Βουλή θεωρούμε, θεωρούμε ότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι και αν κάποιο λέει κάτι, κρατάει το λόγο του. Δεν χρειάζεται να αναμασάει τα πράγματα χιλιάδε φορέ. Αλλά αν θέλετε κάθε φορά σε κάθε πάνελ να επαναλάβουμε τα ίδια, πολύ ευχαρίστω. Η Ουγγαρία και η Ουγγρική κυβέρνηση ενδιαφέρονται για συνεργασία και έχουμε συμφέρον η Ουγγρική νομοθεσία να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο και να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θέλετε κι άλλο, σα το είπα χιλιάδε φορέ και τηλεφωνικά και γραπτό και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εμεί θέλουμε ε, και να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, ε, ετοιμάζοντας τις νομοθετικές μας προτάσεις. Εγώ σας ρωτάω, θα δεχθείτε και θα εφαρμόσετε τις συγκεκριμένες συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Yes, Mr. Prime Minister. Ο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αν οι προτάσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στο Ουγγρικό Σύνταγμα και στην Ουγγρική νομοθεσία, ναι. I think that'll be a point. Would you like to comment? that, is άλλο αυτό και άλλο αυτό που μου λέγατε στο γραφείο μου. Συγγνώμη. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ακριβώς το ίδιο σας είχα πει και εκεί. Είμαι βουλευτής και ορκίστηκα πίστη στο Σύνταγμα και στο Ουγγρικό κράτος. Δεν λέω ότι αυτά που θα μας προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης θα αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στην Ουγγρική νομοθεσία. Είπα ότι αν δεν αντιβαίνουν θα τα εφαρμόσουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορεί να μας υπαγορεύσει οτιδήποτε αντιβαίνει στο Ουγγρικό Σύνταγμα και στην Ουγγρική νομοθεσία. Νομίζω ότι η αμορφιά και το μεγαλείο ακροάσεων σαν αυτή είναι ότι είναι ζωντανές, είναι ζωντανή αναμετάδοση, είναι μια κατά μέτωπο αντιπαράθεση ζωντανή και σφοδρή διαφόρων απόψεων. Και μερικές φορές είναι και απαραίτητη αυτή η αντιπαράθεση. Την εκτιμούμε ιδιαίτερως λοιπόν και λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά τα σχόλια. Είμαστε άλλωστε αυτόπτες μάρτυρες αυτής της συζήτησης και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο δεύτερο μας πάνελ. Ευχαριστώντας φυσικά θερμά τους προσκεκλημένους του πρώτου πάνελ που μας έκαναν το δώρο της παρουσίας τους και των ομιλιών τους. colleagues, dear guests, as I say, we still have a way to go. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, παρακαλώ καθίστε. We still have a way to go. And mostly. Λοιπόν, έχουμε ακόμα πολύ δουλειά και κυρίως πρέπει να προλάβουμε και την καθυστέρηση που ήδη σέρνουμε πίσω μας. Σκεφτείτε τους δερμηνείς. Σκεφτείτε το σύστημα δερμηνίας που είναι προγραμματισμένο μέχρι τις μισή. Εάν δεν, εάν δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε και να επιβαρύνουμε το τελευταίο μέρος της απόψινής ακρόασης, ας προσπαθήσουμε να προλάβουμε το χρόνο, καλωσορίζοντας τους συνέδρους που είναι εδώ τώρα στο Προεδρείο έτοιμοι να κάνουν τις συνεισβολές τους. Ανακοινώνω. Σιωπή παρακαλώ all be With all respect. Με όλο το σεβασμό παρακαλώ σιωπήστε. Σεβαστείτε του συνέδρους που είναι εδώ στο Προεδρείο, τους ομιλητές. Έχουμε τον κύριο Ουμπέρτε Βιολέη, που είναι εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, σύνδεσμος με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κύριος ε, Μόρτον Τζέραλντ, καλώς ορίσατε, Διευθυντής του, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, FRA, και την κυρία Ντούνια Μεδιάτονιτ, που είναι εκπρόσωπος της ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καλώς ήλθατε. With no delay to the first of... Και δίχως περαιτέρω καθυστέρηση να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας. 10 λεπτά! Και έπειτα γύρω στον ε, συντονιστών, δύο λεπτά έκαστος. Και κάθε μέλος που θέλει να παρέμβει, να θέσει ερώτηση, να έχει υπόψη του. Ερωτήσεις θέλουμε, όχι αγορεύσεις. Για 1,5 λεπτό. Και... Παρακαλώ, κύριε Ντουβιλέ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Υπάρχει μια αντικατάσταση εδώ στο αρχικό πάνελ που είχαμε προβλέψει. Δεν έχουμε τον κύριο Ιμπέρ Ντεβιολέ. Τον κύριο Άντριου Κάτινγκ που, που εκπροσωπεί εδώ το, την υπηρεσία σύνδεσης ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης με το την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, χτυπήθηκε το γραφείο μας από τη γρήπη που σοβίδω στο Βέλγιο τελευταίος. Επίσης, τυχώς ξέρω ότι καλέσατε κάποιον από την Επιτροπή ε, την ομάδα μάλλον των συνταγματικών εμπειρογνωμόνων να έρθουν σήμερα, αλλά δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα και εγώ δεν είμαι τεχνικός εμπειρογνώμονα, αλλά μπορώ να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης όπως, ε, και την άποψη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εσείς έχετε σίγουρα εξετάσει κάποια από αυτά τα σημεία ήδη. Θα ήθελα σύντομα να ανακεφαλαιώσω τη δική μας ε, μπλοκή μέχρι στιγμή. Στις 25 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους, ο Επίτροπός μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Τόμας Χάνομπεργκ, εκπώνησε μια γνωμοδότηση για την ελευθερία του τύπου στην Ουγγαρία, που ε, προκάλεσε ανησυχίες όσον αφορά το, πακέτο, το νομοθετικό πακέτο περί ΜΜΕ. Στον Μάρτιο του 2011 ακολούθησε μια πρώτη γνωμοδότηση από την Επιτροπή της Βενετίας που όπως είπα είναι ένα σώμα ανεξορτήτων ε, πυρογνωμόνων συνταγματολόγων και αυτή η γνωμοδότηση ζητήθηκε από τις εγκρικές αρχές και φορούσε συγκεκριμένα τη διαδικασία που οδηγεί στην υιοθέτηση του συντάγματος και όχι το ίδιο, θα αφορούσε τη διαδικασία και όχι το ίδιο το περιεχόμενο. Κάποιου μήνε αργότερα, τον Μάιο πέρυσι, η Επιτροπή τη Βενετία υιοθέτησε περαιτέρω γνωμοδότηση που αφορούσε το περιεχόμενο του συντάγματο. Προέκυψε αυτό από αίτημα τη δική μα κοινοβουλευτική συνέλευση. Όπω πιθανότατα γνωρίζετε, αυτέ οι δύο γνωμοδοτήσει έκαναν κάποια θετικά σχόλια. Καλωσόρισαν το γεγονό ότι το Σύνταγμα είχε συνταχθεί καταρχήν και έπειτα κάποιες ε, διατάξεις συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να προκαλέσει συνταγματικά κάποιος ε, ε, για κάποιο ζήτημα, πράγμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, αλλά αναφέρονταν και κάποιες ανησυχίες. Μετά τον Ιανουάριο φέτος, τον περασμένο μήνα, ο Γενικός μας ο κύριο Γιάκλαντ, έστειλε επιστολή στον Ούγγρο Υπουργό Εξωτερικών και πάλι προσφέροντας την εμπειρογνωμοσύνη και τη συμβουλή της Επιτροπής της Βενετίας σε σχέση με τρία συγκεκριμένα θέματα που ήταν το δικαστικό σώμα, η ανεξιθρησκεία και ο εκλογικό νόμος στην Ουγγαρία. Έγινε μια ανταλλαγή επιστολών με τι ουγγρικέ αρχέ, ω αποτέλεσμα τη οποία λάβαμε ένα επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή της Βενετίας για να εξετάσει αυτούς τους τρεις συνταγματικού νόμους και αυτή η εργασία είναι υπό εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μια ακόμη εξέλιξη, την 1η Φεβρουαρίου μόλις, η κοινοβουλευτική μας συνέλευση στην Σύνοδο της Ολομέλειάς της ζήτησε πέντε περαιτέρω γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή της Βενετίας για διαφορετικά ζητήματα. Έχω εδώ ένα κατάλογο που αφορούν την ε, ελευθερία ενημέρωσης, το συνταγματικό δικαστήριο, Διώξει εθνικότητα και προστασία της οικογένειας. Οχτώ διαφορετικές νομοθετήσεις έχει να εκπονήσει τώρα η Επιτροπή της Βενετίας σε σχέση με την Ουγγαρία. Μαζί με τις ε, μάλλον έχουν προετοιμαστεί, προγραμματιστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου και πιο συγκεκριμένα το ε, πρόκειται για την γνωμοδότηση του δικαστικού σώματος και την ανεξιθρησκεία. Αυτέ οι δύο γνωμοδοτήσει θα υιοθετηθούν από την Επιτροπή τη Βενετία στην Ολομέλειά τη στην Βενετία στα τέλη του Μαρτίου. Οι επόμενε πέντε γνωμοδοτήσει, μάλλον έξι, θα υιοθετηθούν τον Ιούνιο. Αλλά εκεί χρειάζεται περαιτέρω επισκέψει στη Βουδαπέστη και περαιτέρω συζητήσει με τι αρχέ. εκεί. Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονό ότι η Ουγγαρία και 46 άλλε χώρε από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο έχουν αναλάβει δεσμεύσει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μεταξύ του, και προ το Συμβούλιο τη Ευρώπη υπό, μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου, αλλά και μέσω των συστάσεων της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι σημαντικό δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όχι μόνο προς την Ένωση αλλά και προς το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και με τον καιρό το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει πολλή εμπειρία όσον αφορά την παροχή συμβουλών προς τις χώρες για το πώς μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές οι οποίες έχουν συνυπογράψει. Ε, αρρωγή μπορούν να μπορεί να προσφέρει, όπως στην σημερινή κατάσταση το Συμβούλιο είναι ανοιχτό, μπορεί να συμβουλέψει οποιοδήποτε θέμα του ζητηθεί από τις Ουγγρικές Αρχές, σε στενή συνεργασία φυσικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα και με τις αρχές ε, και με τα κράτη-μέλη, τα υπόλοιπα. Σε σχέση με το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε και όπως σας είπα θα είμαι σύντομος και θα βασιστώ μόνο σε στοιχεία. Ο Γενικός μας Γραμματέας πρόσφατα ανέφερε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι σε θέση να βοηθήσει να προχωρήσει η κατάσταση διότι έχει αυτή την προσέγγιση που βασίζεται στη σύμβαση που είναι ευρύτερη κατά κάποιο τρόπο από ότι οι αρμοδιότητες της Ένωσης και έχει επίση ε, αυτό το μη, την, μη, τον μη πολιτικοποιημένο τρόπο που βασίζεται στην συνένεση να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη για να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές. Και έτσι μπορεί να βοηθήσει όντως να προχωρήσει αυτό το θέμα. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους μας εταίρους. Η Ουγγαρία επίσης ήταν δραστήριο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από τότε που προσχώρησε τόσο για την ανάπτυξη των προδιαγραφών του Συμβουλίου της Ευρώπης όσο και για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε χώρες μεταξύ των οποίων και οι γειτονικέ της χώρες για διάφορα ε, θέματα και εμείς θα καλωσορίζαμε τον, τον ίδιο ανοιχτό πνεύμα σε σχέση με την ε, λήψη τεχνικών συμβουλών ή προτάσεων που μπορεί να προέλθουν από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως αποτέλεσμα, ως απόρρια των εργασιών που γίνονται αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κάθιν και τώρα... Να περάσουμε στο δεύτερο μέλος του πάνελ μας, Στον δεύτερο μιλητή, τον κύριο Μόρταν Τζέρομ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με που καλέσατε το Ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην ακρόαση αυτή σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις αξίες οι οποίες εστιάζονται, οι οποίες ε, ε, κατοχυρώνονται στις συνθήκες. Θα εστιαστώ σε τρία ζητήματα. Καταρχάς, σε θεσμικές ταυτότητες που, ε, όπως ξέρετε, προστατεύονται από το άρθρο 2 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης είναι αλληλεξαρτώμενα. Στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιδών δικαιωμάτων, οι αρμοδιότητε αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσφέρει λοιπόν πλήρη προστασία και έλεγχο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά ασφαλώς εξαρτάται από την ύπαρξη των κατάλληλων ασφαλιστικών δικλείδων στα κράτη-μέλη. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί και εξαρτάται από τα αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα σε επίπεδο κράτων μελών. Και γι' αυτό, λοιπόν, ο χάρτη των μεριδιανών δικαιωμάτων και η συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν όρου για την κατάλληλη νομική προστασία. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν έλλειψη των κατάλληλων νομικών μέσων σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η αλληλεξάρτηση αποτυπώνεται και σε ό,τι αφορά τις ε, βασικές αξίες, τις αξίες πυρήνα. Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών και των πολιτικών δομών των κρατών. Αλλά και στο άρθρο 2 αναφέρεται το θέμα των δικαιωμάτων των, της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου ότι αποτελούν κοινή αξία των κρατών μελών όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν εξαρτάται σε κάποιο βαθμό στην ομοιογένεια που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών όλες της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη, η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναφέρει ότι θα πρέπει τα κρατημέλη να βοηθούν το ένα το άλλο με συνθήκες πλήρους σεβασμού. Επίση αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και ο αμοιβαίο σεβασμός και τα δικαιώματα που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Θα εξαρτώνται από το κατά πόσο σέβονται τα κράτη-μέλη τις βασικές αξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 2 αναφέρονται οι πολιτισμικές ταυτότητες των κρατών μελών, αλλά αναφέρεται και η ενοποίηση. Το ότι είμαστε ενοποιημένοι, ενωμένοι στην ε, διαφοροποίησή μας. Προστατεύουμε μεν τη διαφοροποίηση, αλλά και την ενότητα ο σεβασμός η ε, υποχρέωση σεβασμού των βασικών αξιών περνάει πολύ παραπέρα από την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα νομικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τήρηση των αξιών αυτών είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πολιτική και όχι νομική διαδικασία όπως όλοι ξέρουμε. Για παράδειγμα το ΔΕΚ δεν μπορεί να αποφανθεί για το κατά πόσο μια κατάσταση ε, είναι στον τομέα αρμοδιότητας, στον πέντε αρμοδιότητας του άρθρου 7 ή όχι. Επίσης, η υπηρεσία που εκπροσώπω δεν ε, μπορεί να ξεκινήσει διαδικασίες βάσει του άρθρου 7. Ωστόσο, το Συμβούλιο το 2007 δήλωσε ούτε οι συνθήκες, ούτε οι υπηρεσίες και ο κανονισμός για τις υπηρεσίες δεν αποκλείουν τη δυνατότητα του Συμβουλίου να ζητήσει βοήθεια από την υπηρεσία μας όταν τίθεται θέμα πεδίο εφαρμογή του άρθρου 7. Και να περάσω λοιπόν στο δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω. Το κράτος δικαίου αποτελεί μία συνολική αξία η οποία σχετίζεται με όλες τις άλλες θεμελιώδεις αξίες. Και τι σημαίνει αυτό στο Ευρω... Το κράτος δικαίου προϋποθέτει ότι η η δημόσια εξουσία θα πρέπει να πληρεί κάποιες ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Την νομιμότητα, για παράδειγμα, της κυβέρνησης. Το κράτος θα πρέπει να σέβεται την αρχή της νομικής βεβαιότητας, την αρχή της αξιοπιστίας, την απαγόρευση των ε, πράξεων ε, εκ των υστέρων και την αρχή της αναλογικότητας αν δεν ε, υπάρχουν αυτοί οι όροι, υπάρχει κίνδυνο στα θεμελιώδη δικαιώματα να είναι στα βιβλία μόνο, στη θεωρία, χωρίς να εφαρμόζονται στην πράξη επιτόπου. Από την έννοια αυτή, λοιπόν, τα δυνατά και τα ανεξάρτητα σώματα δικαστικής ε, εξουσίας είναι πολύ βασικά για την ανθρώπινη κοινωνία που βασίζεται σε κράτος δικαίου έννοια αυτή της ε, ανεξαρτησίας αποκλείει οποιαδήποτε έμεση ή άμεση επιρροή που θα μπορούσε να θέσει ε, να αμφισβητήσει την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Άρα, οι δικαστές δεν δρούν μόνο ανεξάρτητα, αλλά θα πρέπει να γίνονται αντιληπτοί και ως ανεξάρτητοι από το κοινό. Η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σώμα αυξάνεται όταν το κοινό βλέπει ότι το δικαστικό σώμα εκφέρει αποφάσεις χωρίς να αναμειγνύεται η διοίκηση, η κυβέρνηση. Και στη διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικός ο διορισμός των δικαστών, η διοργάνωση του δικαστικού, το πώς συστήνονται τα δικαστήρια και πώς ανατίθενται οι υποθέσεις στα εκάστοτε δικαστήρια βασικό, βασική σημασίας είναι το δικαίωμα αποτελεσματικού ενόμου δικαιώματος και δικής δικής. Αυτό το δικαίωμα κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του χάρτη με σαφήνεια και στο άρθρο 19 της ε, Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να παρέχουν επαρκείς και σίγουρες ένομες λύσεις και δυνατότητες ε, για νομική προστασία στους πολίτες τα δικαστήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ε, τυχόν ελλείψεις σε εθνικό επίπεδο. Εξίσου σημαντικέ είναι και οι αρχέ που ελέγχουν την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω για παράδειγμα οι υπηρεσίε προστασία των δεδομένων. Και αυτέ θα πρέπει να τη εμπιστοσύνη, προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά του ανεξάρτητα από εξωτερικέ επιρροέ. Και πρόκειται για ένα από τα βασικά επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ότι εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους ε, κανόνες προστασίας των δεδομένων ελέγχεται από μια ανεξάρτητη αρχή. Κυρίες και κύριοι, και έτσι περνά στο τρίτο και τελευταίο σημείο της ομιλίας μου. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το σύνολο είναι πιο σημαντικό από κάποια μέρη του αθροίσματος. Όταν λέμε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό κίνδυνο παραβίαση κάποιων θεμελιωδών αξιών, σημαντικό είναι να εξετάσουμε όχι μόνο ένα μέσο, αλλά να συνδυαστούν διάφορε δυνατότητε. Αν για παράδειγμα η ανεξαρτησία του δικαστικού και των ε, υπηρεσιών ελέγχου αποδυναμωθεί προ όφελο τη κυβέρνηση, αυτό έχει επιπτώσεις στο συνολικό σύστημα και σε όλες τις αρμοδιότητες. άλλε εξελίξεις όπως η εισαγωγή νέων πλειοψηφιών για την εκλογή των ε, αξιωματούχων, νέε θητείε, νέοι εκλογικοί νόμοι, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συνολική αξιολόγηση. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό το σύνολο είναι σημαντικότερο από τα μέλη, από τα μέρη του. Μια τέτοια αξιολόγηση ενός κράτους μέλους δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολο εγχείρημα γιατί προϋποθέτει ε, συγκριτική, συνεχή, συνεκτική ανάλυση των διαφόρων εξελίξεων. Και με όλα αυτά υπόψη, έναντι και των 27 κρατών μελών, μπορεί να μας βοηθήσει να εγγυηθούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία θα εξασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστούμε. Και περνάμε στον τρίτο εμπειρογνώμονα, την κυρία Ντούνια Μιγιάτοβιτς. For the next 10 Σας ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στην ακρόαση αυτή. Χαίρομαι ιδιαίτερως για τη διοργάνωση αυτή, γιατί οι διεθνείς οργανώσεις όπως ε, και η ΟΑΣΕ δι, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ε, αφύπνιση και την προειδοποίηση των κυβερνήσεων ε, προκειμένου να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις και να, δείξουν, να δείξουμε ότι οι διεθνείς οργανώσεις ενδιαφέρονται για τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτές και μεριμνούν ώστε να τηρούνται έστω και προαιρετικά συμπεφωνημένες υποχρεώσεις. Από το 1957 η ΟΕΣΕ και τα μέλη τους ε, ανέλαβαν την ευθύνη να ε, εφαρμόσουν ε, διάφορες αξίες και αρχές όπως το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιδών ελευκαιριών, της ελευθεροτυπίας, της ελεύθερης έκφρασης, του πλουραλισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα είμαστε ίσως η μόνη διακυβερνητική οργάνωση ε, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, που εκπροσωπείται και στα 27 κράτη-μέλη προκειμένου να βοηθήσουν τα κράτη να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις και να τους υπενθυμίσει, να τους επαναφέρει στην τάξη, να τους ε, επισημάνει, να τους κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου σε περίπτωση που τους παραβιάζουν. Σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία, θα ήθελα να σας αναφέρω τις απόψεις μου για τη σχετική νομοθεσία της Ουγγαρίας και την επικείμενη αναθεώρηση. Από τον Ιούνιο του 2010 όταν ε, υπευλήθη το νομοσχέδιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ουγγρική Βουλή, είχα ήδη κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Σήκωσε την κόκκινη σημαία που ονομάζεται έγκαιρη προειδοποίηση. Τότε βέβαια η φωνή μου στη διεθνή σκηνή ήταν μια μοναχική φωνή. Υπέβαλα παρατηρήσεις για τα προβληματικά σκέλη αυτού του νομοσχεδίου και δημοσίου σε ομιλίες μου και σε συνομιλίες με τις Ουγγρικές Αρχές. Αυτό το 1,5 χρόνο το γραφείο μου είχε συνεχή διάλογο με τις Ουγγρικές Αρχές και μάλιστα μίλησα δημοσίω για την ετοιμότητα και την προθυμία της Ουγγρικής Κυβέρνησης να εξετάσει τα προβλήματα αυτά. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται εν εξελίξη. Επί της ουσίας δυστυχώς βέβαια διαφωνούμε. Και θα ήθελα σήμερα εν συντομία να σας παρουσιάσω ε, Πού έγκυται η διαφορά μας. Η Ουγγαρία, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμμετέχει στην ΟΑΣΕ και ανήκει και στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλες διεθνείς οργανώσεις. Κάθε συμμετοχή προϋποθέτει υποχρεώ, υποχρέωση εφαρμογής των αρχών της κάθε οργάνωσης και στην εθνική νομοθεσία. Και μάλιστα ως μέλος της ΟΑΣΕ τα, η Ουγγαρία είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τι εξή αρχέ προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τι διεθνεί σωστέ πρακτικέ. Μετά την απόφαση του Ουγγρικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που την επικροτώ γιατί έβαλε την δικαστική σφραγίδα σε όλε τι ε, ε, συστάσει που έκανε και το γραφείο μου από τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και ε, Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποίηση αυτές έπρεπε ήδη να υιοθετηθούν από την 1η Μαΐου του 2011 και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, αυτές οι συστάσεις προκειμένου να τηρηθούν οι διεθνείς προδιαγραφές και από την Ουγγαρία. Το γραφείο μου είναι πρόθυμο να βοηθήσει την Ουγγαρία σε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση και μάλιστα περιμένω το νέο νομοσχέδιο, το αναθεωρημένο νομοσχέδιο, όπως συμφωνήσαμε με τον Υπουργό Επικρατείας ε, και Επικοινωνιών στις πρόσφατες επαφές που είχαμε στη Βιέννη. Υπάρχουν όμως και άλλε διατάξει ε, του νόμου περί μέσων μαζικής ενημέρωσης που επίση θα πρέπει να τροποποιηθούν. Για παράδειγμα, η διαδικασία για την επιλογή ε, των μελών και του Προέδρου του Συμβουλίου των ε, Μίντια και της αρχής των Μίντια. Επίσης, να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των συντακτών των εφημερίδων. Υπάρχουν μερικές φορές αόριστες διαφάνεια, όριστοι ε, ορισμοί και τα θέματα των προστήμων και των κυρώσεων θα πρέπει να διευκρινιστούν. Στα θέματα καλών ε, πρακτικών, αυτό δεν είναι αμυγής υποχρέωση που απορρέει από την ΟΑΣΕ, αλλά θα πρέπει ε, να συγκεντρωθεί η συνταγματική πλειοψηφία των δύο τρίτων για να κριθεί το νομοσχέδιο αυτό. Κανένας δεν διαφυσβητεί την νομιμότητα μια τέτοια κίνηση και απέτηση τέτοια πλειοψηφία. Το θέμα είναι θα πρέπει ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο να σφυριλατηθεί με τέτοιο τρόπο μια και, ή να, να μαρμαρώσει με κάποιο τέτοιο τρόπο να βλέπουμε πόσο ραγδαίες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις στα μίδια. Είχαμε και την ε, ομιλία του αρμοδίου του ΟΗΕ και του αρμόδιου Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είδαμε ότι η Ουγγρική κυβέρνηση εφαρμόζει επιλεκτική προσέγγιση ό,τι αφορά την τήρηση των διεθνών της υποχρεώσεων. Ανταποκρίθηκε σε κάποιες επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα ε, μας διαβεβαίωσε θα ληφθούν υπόψη στάσει του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αλλά οι υποχρεώσει που παρέουν από τη συμμετοχή ε, στον ΟΗΕ, στην ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, οι υποχρεώσεις αυτές ε, δεν έχουν ε, τηρηθεί από την Ουγγαρία. Η Ευρώπη ε, και τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να γίνονται παραδείγματα προς μίμηση αν θέλουν και άλλες χώρες να ακολουθήσουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Αν κανείς συμμετέχει σε μια ε, επίλεκτη λέσχη όπως είναι η ΟΑΣΕ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε τα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτήν την ε, επίλεκτη λέσχη να είναι πραγματικά υποδείγματα και σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία και σε ό,τι αφορά τον πλουραλισμό και τα ελεύθερα μέσα μαζική ενημέρωση. Κάτι άλλο. Μερικέ φορέ έχω την αίσθηση ότι αυτή η επίλεκτη λέσχη, αυτή η ελίτ, ξεχνάει ότι πολλέ χώρε στην Ευρώπη γνωρίζουν ότι όπω και η δημοκρατία, η ελευθεροτυπία και η ελευθερία έκφραση δεν είναι κάτι δεδομένο που κατοχυρώνεται άπαξ και διαπαντός. Θα πρέπει συνεχώ να δικαιολογούνται, να επανεπιβεβαιώνονται και να ενισχύονται. Γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι και οι ευρωπαϊκέ χώρε θα πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα σε τέτοια περίπτωση και να γίνονται υπόδειγμα και παράδειγμα προ μίμηση. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τι ε, συστάσει και το του Συνταγματικού Δικαστηρίου, θα κάνουμε μία ανάλυση, νομική ανάλυση και θα ετοιμάσουμε συστάσει για να ληφθούν υπόψη από του ε, Ούγγρου νομοθέτε κατά την τροποποίηση τη νομοθεσία. Μάλιστα, πρότεινα εμπειρογνώμονες από το γραφείο μου να μεταβούν στην Ουγγαρία για να βοηθήσουν με την τεχνογνωσία τους στην προσπάθεια τροποποίησης νομοθεσίας. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης αν τηρηθούν οι συστάσεις, οι απαιτήσει μάλλον του Συνταγματικού Δικαστήριου. Για παράδειγμα, ε, ο τύπος να αφαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογή ε, του νέου νόμου. Εγώ ζητώ από την Ουγγρική κυβέρνηση να μην περιοριστεί στις ελάχιστες προδιαγραφές που απέτησε το Συνταγματικό Δικαστήριο και να ευθυγραμμίσει την, την νομοθεσία για τα μίδια με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και το τελευταίο μήνυμα ε, ευκαιρία της συμμετοχής μου σε αυτή την δημόσια κρόση θα ήθελα να στείλουμε ένα μήνυμα προς τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών προκειμένου να κάνουν ό,τι μπορούν και να μην θεσπίζουν νομοθεσίες που καταστέλουν ή περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση, τις ε, θέματα ταμπού, τις ε, αντίθετες φωνές. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα δημοκρατικού διαλόγου σε μια δημοκρατική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε και τώρα να προτείνω να περάσουμε κατευθείαν στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Να προτείνω κάθε πολιτική ομάδα να να πάρει το λόγο και μετά να μιλήσουν άλλοι τέσσερις βουλευτές και να προτείνω οι συντονιστές ε, να πάρουν το λόγο αν το θέλουν ή αν θέλουν μπορεί να ορίσουν κάποιον να, ε, να τους εκπροσωπήσει. Η κυρία Γκάλα, λοιπόν, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Να σας πω καταρχάς, ένα φαινόμενο το οποίο έχουμε βιώσει και προηγουμένως. Εγώ να σας πω ότι είμαι πολλά χρόνια εδώ, 6,5 χρόνια και ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί αυτό που θα σας περιγράψω τώρα. Μία επιτρόπος να θέλει να επιβάλλει στην Ουγγαρία και συγκεκριμένα σε έναν αντιπρόεδρο ένα κείμενο το οποίο δεν το έχει δει κανένας. Ε, είναι κάτι που υπερβαίνει πάρα πολύ ε, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτρόπου. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχω γνώση του να έχει γίνει απόπειρα να γίνει κάτι τέτοιο ποτέ στο παρελθόν σε έναν πρωθυπουργό ή σε έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και θέλω να γραφεί στα πρακτικά παρακαλώ ότι πρόκειται για ανευπροηγουμένου παρέμβαση της Επιτρόπου. Δεύτερον, πράγματι Άμα ψάξει θα βρει προβλήματα η Κομισιόν. Ε, εδώ μιλάμε για ε, συγκεκριμένους ε, νόμους που λέω ότι δεν είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι στο κοινοτικό κεκτημένο. Αυτά τα προβληματικά κομμάτια της νομοθεσίας και η Ουγγαρία, θέλει να τα διορθώσει και γίνονται οι σχετικές προσπάθειες. Δεν νομίζω όμως ότι σήμερα αυτό ενδιαφέρει τους ελεύθερους και τους σοσιαλιστές. Δεν είναι αυτό για αυτούς το πραγματικό θέμα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να εκτοξεύουν προσβάσιμες κατηγορίες που βασίζονται απλά και μόνο σε πληροφορίες που έχουν από ε, δημοσιεύματα του τύπου ή από επιστολές που έχουν λάβει. Λένε ότι είναι το τέλος της δημοκρατίας, το τέλος της ελευθερίας έκφρασης. Ε, να σας πω κάτι, δεν πάτε καλύτερα στην Ουγγαρία, δεν κλείνετε την τηλεόραση, δεν πάτε καλύτερα να τα δείτε από κοντά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος τον οποίο να εμποδίζουν να εκφράσει την άποψή του. Και τώρα στρέφομαι στο Επίτροπο των Μέσων Επικοινωνίας. Πριν από κάποια χρόνια στην Ουγγαρία, πράγματι η κυβέρνηση προηγούμενη είχε αποκλείσει ορισμένους ε, τομείς, ε, ορισμένους δημοσιογράφους από τις συνεντεύξεις τύπου. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για κάτι αντίστοιχο. Αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε σοσιαλιστές και φιλελευθέρους στην κυβέρνηση πάει και δημοκρατία. Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν έχουμε, αυτή η συζήτηση δεν έχει καμία σημασία, κανένα το μόνο που έχει να κάνει είναι να ε, οξύνει ε, τον ευρωσκεπτικισμό, την ε, αντιπάθεια προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση πραγματικά ξυλοκοπά τους αθώους διαδηλωτές. Το έχουμε δει. Και συγκεκριμένα συνέβη στην Βουδαπέστη το φθινόπωρο του 2006 τότε υπήρξε ένα σοσιαλιστής φιλελεύθερος ε, κύριος ή κυρία που να προάσπισε τα δικαιώματα των δημοσιογράφων ή των απλών ανθρώπων. Ουδής. Εγώ μπορώ να σας δώσω εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα. Άρα μιλάμε για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και τι κάνει αυτή η τακτική. Το μόνο που κάνει, επαναλαμβάνω, είναι να οξύνει ε, τον ευρωσκεπτικισμό και τον εξτρεμισμό με τον τρόπο αυτό τελικά τίθεται ε, σε κίνδυνο ε, όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να πω ότι αυτό που θέλουν να κάνουν οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές είναι να κάνουν αδύνατη ε, την εργασία της ουγγρικής κυβέρνησης. Το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των Ούγγρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, βεβαίως. make... Κάθε μέλος μπορεί να πει αυτό που θέλει. Προτείνω όμως να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε στο θέμα και να υποβάλουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Κάλιο αυτό παρά ομιλίες, γιατί θέλουμε να σεβαστούμε το χρονικό μας πλαίσιο. Έχουμε άρα δύο πάνελ που πρέπει να περάσουν και θα συσσωρεύσουμε καθυστερήσεις αν δεν αλλάξουμε τρόπους. Κύριε Βάλτεν Χόλτσα, έχετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω, να ζητήσω από την κυρία Γκάλ να μου πει αν άκουσα αυτά που είπε η κυρία Μπεάτοβιτς. Πρόεδρε, από ό,τι ξέρω από το προηγούμενο κομμάτι, υπήρχαν συνάδελφοι που ήθελαν να παρέμβουν σηκώντα τη γαλάζια κάρτα και δεν του επιτράπει. Άρα δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα. Άκουσα, βεβαίως, βεβαίως άκουσα αυτά που υπόθηκαν. Καλώς λέει ο πρόεδρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, κανένα μέλο δεν στερήθηκε το δικαίωμά του να σηκώσει το χέρι του ή να πει κάτι στον προηγούμενο γύρο. Εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο ανοιχτό γίνεται. Αλλά βοηθήστε με για να μπορέσουμε να προλάβουμε το χρόνο. Η κυρία Γκόντ για το SD έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη και δεν θα ακολουθήσω αυτή τη διαμάχη. Έχω κάποιες σύντομε παρατηρήσει σχετικά με αυτά που μόλι υπόθηκαν. Άντας Μπόκα δεν είναι πλέον πρόεδρος διότι δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες. Να μιλήσω αγγλικά, λέει ο κύριος. Η, η, κυρία. Α, η κυρία μάλλον, συγχωρείτε. Πολύ σύντομα σχόλια. Αυτά που είπε ο Γιάννος θέλω να σχολιάσω. Ότι ο Μπόκολντας που ήταν πρόεδρος του πρώην ανωτέρου, ανωτάτου δικαστηρίου δεν πληρεί τα κριτήρια του νέου νόμου, άρα δεν μπορεί να μείνει στη θέση του. Αυτό ήθελα να πω. 17 χρόνια υπηρετούσε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Άρα νομίζω θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός. Σύντομο σχόλιο ήταν αυτό. Έχω και ερώτηση προς τους ε, εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο κ. Κέρου είπε το σύστημα είναι κάτι παραπάνω από το άθισμα των συστατικών μερών. Είπατε ότι η Επιτροπή της Βενετίας έρευνα ή μελέτα οκτώ νόμους. Θα ήταν σημαντικότατο να δούμε το πακέτο συνολικά. Τις προσωρινές διατάξεις, το βασικό νόμο και το βασικό δίκαιο. Αν μιλάμε για δίκες εκλογές δεν αρκεί να μελετήσουμε τον εκλογικό νόμο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, τον νόμο για σταθερότητα που καθορίζει με δύο τρίτα πλειοψηφία το φορολογικό σύστημα και οι προσωρινές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα ποινικοποίησεως του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολιτεύσεως. Αν αναφερόμαστε σε αυτού του είδους το πλαίσιο θα ήταν πολύ σημαντικό μελετήσουμε όλη τη δέσμη μέτρων και όχι ξεχωριστούς νόμους. Το Συμβούλιο της Ευρώπης σκοπεύει να το κάνει αυτό. Η Επιτροπή της Βενετίας σκοπεύει να το κάνει αυτό. κυρία Βέλε, ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία για τον κύριο Κέτιν σχετικά με αυτά που θα πρέπει να κάνει η Επιτροπή της Βενετίας. Ερώτηση. Πόσες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πέρασαν Τέτοιε διαδικασίες για το σύνταγμά του, να αναλύνεται το σύνταγμά του. και οκτώ βασικούς κύριο σώμα νομοθεσία να εξετάζεται. Υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το αντιμετώπισε αυτό. Και δύο ερωτήσει για τον κύριο Κέρουγκ. Αναφερθήκατε στη γενική εικόνα που είναι σημαντική Αναφερθήκατε στην ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και το κράτος δικαίου. Ερώτηση. Μία χώρα όπου γενικός εισαγγελεύς μπορεί να αναθέτει υποθέσεις σε κάποια δικαστήρια. Οπότε δεν έχουμε τυχαία ανάθεση. Αλλά ένας γενικός αγγελέας να αναθέτει αυτός τις υποθέσεις. Το θεωρείτε ότι ταιριάζει με το κράτος δικαίου. Και άλλη ερώτηση. θεωρείται απάντηση εκτό μικροφώνου, δεν να ακούει Μία χώρα με ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος ασχολείται με τα δικαστικά, το δικαστικό κλάδο, με τους δικαστέ και όπου το προσωπικό διορίζεται από το κοινοβούλιο, από τα δύο τρίτα του κοινοβουλίου. Και κατά σύμπτωση διορίζεται η γυναίκα ενό επιφανούς μέλους του κυβερνώντος κόμματος σε αυτή τη θέση. Θεωρείτε ότι αυτό είναι σωστό, συνάδει, υπάρχει ηθική βάση. Μπορεί να μην είναι νομικό σωστό, αλλά θεωρείται ηθικό ότι είναι σωστό. Για του πρασίνου ο κ. Σταλαβάρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπε κάτι ο κύριος Κίρμε, που αναφέρθηκε από κάποιον άλλον, ότι το άθισμα είναι κάτι παραπάνω από το άθισμα των συστατικών μερών, το σύνολο δεν αφορά ένα άρθρο και ένα νόμο αυτή η συζήτηση. Όταν αλλάζει το λόζο, το, συγγνώμη, το νόμο για τα μέσα ενημέρωση, αλλάζει το Σύνταγμα, αλλάζει τη βασική νομοθεσία, κάνει πολύ βαθιέ τομέ στο δικαστικό τομέα, έχουμε ένα ολόκληρο αστερισμό, συστάδα πολιτικών κινήσεων που αλλάζουν την οτροπία, τα, θεμέλια τα ίδια του πολιτικού προσκυνίου, της πολιτικής σφαίρας στην Ουγγαρία. Είπατε επίσης ότι η χρήση του άρθρου 7 ε, είναι πολιτική κίνηση και όχι νομική. Υπάρχουν δύο ειδών πολιτικές χρήσεις, στο άρθρο 7.1 για το Κοινοβούλιο και στο 7.2 για το Συμβούλιο. Ας κάνουμε μια διάκριση, διότι αυτό είναι ένα επιχείρημα που έχει χρησιμοποιήσει η Ουγγρική κυβέρνηση μεταξύ πολιτικού τομέα και ιδεολογικού. Πολιτική χρήση δεν είναι ιδεολογική. Η πολιτική χρήση σχετίζεται με τα θεμέλια της πολιτικής. Δεν είναι θέμα συντηρητικών κατά σοσιαλιστών, υφερελευθέρων και προοδευτικών κατά κάποιον άλλων. Η δημοκρατία τους χωράει όλους. Έκκληση απευθύνω προς συναδέλφους του ΕΛΚ. Μην το κάνετε αυτό θέμα διαμάχης συντηρητικών κατά σοσιαλιστών ή συντηρητικών κατά προοδευτικών. Αρκεί αυτό σε δύο χρόνια να συζητούμε κάποια μέτρα αριστερή κυβέρνηση που τα δεξιά κόμματα θα είναι αντίθετα με αυτά και ελπίζω τα μέλη του Κοινοβουλίου θα είναι συνεπή εν τη αυτή περίπτωση. Όπως κατά το παρελθόν συζητήσαμε με πολλές άλλε χώρε. Ιταλία, Ιρλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία και θα μπορούσα να λέω και να λέω και να λέω. Πρέπει να είμαστε συνεπεί στο Κοινοβούλιο και απευθύνω έκκληση προ την Ουγγρική κυβέρνηση. Και η Ουγγρική κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεπή όσον αφορά αυτά που λέει, τη στάση τη και τι πράξει τη. Αρκετά τακτικέ υποχωρήσει είδαμε, αρκετέ. Θέλουμε να ξέρουμε, η Ουγγρική κυβέρνηση είναι έτοιμη να είναι αξιόπιστο εταίρο στο διάλογο που ξεκινά. Διότι αν δεν είναι, τότε θα πρέπει αυτός ο διάλογος να κινηθεί σε ανώτερο επίπεδο, όπως προβλέπει το άρθρο 7.1 που εναπόκειται στο κοινοβούλιο να το χρησιμοποιήσει. ECR, εκπρόσωπο του ECR θέλει να πάρει το λόγο. ECR, εκπρόσωπο του ECR, εσεί, ορίστε. ECR, ECR. Η κυρία Βοητσόφσκι. Ο κύριο Βοητσόφσκι. ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά που παρίσταμε. Είμαι αναπληρωματικό μέλος ε, στην Επιτροπή αυτή. Πρέπει να σα πω ότι παρακολούθησα τη συζήτηση μέχρι τώρα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά μου έχει αφήσει μια πικρή γεύση. Δεν γνωρίζω βέβαια την κατάσταση στην Ουγγαρία με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά εξακολουθώ να αποκομίσω την εντύπωση ότι κάτι πολύ στραβό συμβαίνει με την θέση και την προσέγγιση μας απέναντι στη δημοκρατία. Από ό,τι φαίνεται, με την Ουγγαρία ισχύει το εξή. Το κυβερνών κόμμα έχει ε, τη συντριπτική πλειοψηφία, ε, όχι ε, ό,τι ισχύει σε αλλε χωρε αλλά αυτό αποφάσισε ο Ουγγρικό λαο στι εκλογέ. Να στηρίξει το κυβερνών κόμμα που προφανώς αυτό είναι στα υπέρ του και είναι λάθος των άλλων κομμάτων που ε, γι' αυτό έχασαν και πολλές ψήφους προφανώς. Έρχομαι τώρα στο γκρικό θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να υπερβούμε το ουγγρικό θέμα. Η πολιτική ανεξαρτησία είναι ένα, αλλά η δημοκρατία ουσιαστικά είναι η απόφαση να δοθούν εξουσίες σε κάποιους πολιτικούς. Υπάρχει τάση κάποιες φορές να μιλάμε για την ανεξαρτησία φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Εισαγγελείς, κεντρικές τράπεζες, φυσικά, συμφωνώ. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να καταλήγουμε στα λάθος συμπεράσματα. Ότι καλό είναι να έχουμε δηλαδή ορισμούς και όχι εκλογές σε αυτές τις θέσεις. Όχι. Οι αιρετοί εκπρόσωποι, τα αιρετά όργανα είναι αυτό που πρέπει να υποστηρίξουμε. Άκουσα κάποιε επικρίσει για κάποια θέματα, αλλά νομίζω ότι εδώ μιλάμε ουσιαστικά για τη δημοκρατία στην Ουγγαρία και βλέπουμε ότι δεν γίνεται σεβαστή αρκετά. Ωραία, δεν έχουμε να ακούσουμε άλλε παρεμβάσει από τι προσώπου των πολιτικών ομάδων και θα ακούσουμε τώρα του διαφόρου συναδέλφου. Ο κύριο Ζάγερ θα είναι ο πρώτο ομιλητή από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη θέση για να, το λόγο για να θέσω μια ερώτηση. Άκουσα την κυρία Ανίλη Κρούς ότι πρέπει οι απόψεις μας να βασίζονται στα γεγονότα. Με χαροποίηση δήλωση, αλλά ξέρετε αυτό πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Ας μην περιπλέκουμε λοιπόν τη συζήτηση, ας περιοριστούμε στα γεγονότα. Νομίζω ότι θα πρέπει και ε, του τύπου να μελετήσει την κατάσταση και το παρελθόν. Υπήρξαν ε, κάποιες διαδικασίες για την ε, ανανέωση των αδειών των ε, σταθμών. Δεν ξέρω, μιλήσατε τότε για την ε, ελευθερία του τύπου, για την ελευθεροτυπία. Τι είχατε πει τότε, θα ήθελα να δω τις δηλώσεις σας. Γιατί μεταξύ των δύο γύρων των εκλογών του 2010 ανανεώθηκαν οι άδειες ε, κάποιων σταθμών όπως του Group Radio. Τότε είχατε μιλήσει εσείς, είχατε πει τίποτα. τι είπατε ή τι δεν είπατε όταν στις αρχές της χιλιετίας με την σοσιαλιστική κυβέρνηση τότε στην Ουγγαρία δεν επέτρεπε η κυβέρνηση των σοσιαλιστών και των φιλελευθέρων οι συντηρητικοί να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες όταν συμμετείχαν στα ΔΣ. Τότε είχατε υψώσει τη φωνή σας. Και αν ναι, σας παρακαλώ να μου διαβιβάσετε εγγράφος τις δηλώσεις σας, εάν υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, θα ήθελα να λάβετε υπόψη και αυτό που είπε η Σόφι Ιντβέλτ. Σε ό,τι αφορά την μειονότητα των Ρωμά που επί της κυβέρνησης ε, έφυγαν μαζικά από τη χώρα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τελικά για να καταλάβω αν υπάρχουν δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Βλέπουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, τον Πρόεδρο Παρόσο, την ε, Επίτροπο Ρέντινγκ, την Επίτροπο Κρούς. Όλοι έχουν αναφέρει ανησυχίες και έχουν θέσει ερωτήματα σε σχέση με τη λειτουργία της δημοκρατίας ε, στην Ουγγαρία από συνταγματικής πλευράς ε, καθώς και όσον αφορά την ανεξαρτησία ε, της ε, δικαιοσύνης. Η Χίλαρη Κλίντον, ο Έλεν Ζιπέ επίσης έχουν αναφέρει προβλήματα τα οποία υπάρχουν εντός των δημοκρατικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην Ουγγαρία. Έχω ακούσει στο Στρασβούργο και άκουσα και εδώ ε, την ε, αιμονή που έχει να κάνει με την ε, παγκόσμια συνωμοσία των σοσιαλιστών και φιλελεύθερων κατά της Ουγγαρίας. Νομίζω ότι αυτό πλήττει την αξιοπιστία την, ε, της Ουγγαρίας και των ηγετών της, ε, αυτών που προωθούν δηλαδή την ιδέα αυτή. Και επίσης όλα αυτά τα ονόματα σοσιαλιστές είναι, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, κάποιοι από αυτούς είναι μέλη του ΕΛΚ. Και και έχουν διοριστεί ή έχουν προταθεί από το ΕΛΚ. Ο Έλμαρ Μπρόκ σε γερμανική εφημερίδα τον Ιανουάριο του 2011 δημοσίευσε δίστηλο άρθρο για την κακή λειτουργία της δημοκρατίας ε, στην ε, Ουγγαρία. Στις αρχές του 90 ήταν φιλελεύθερος όπως ε, και ο κύριος Ορμπάν. Τώρα είναι όλοι αυτοί οι σοσιαλιστές. Και Τελική ερώτηση. Αν οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι αυτομάτως είναι ένοχοι, θα πρέπει θα πρέπει να φοράμε αστέρι για να φέρει τη διαφορά ανάμεσα σε εμά και σε αυτού. Ε, κάτι σάπιο υπάρχει και όχι στο βασίλειο τη Δανία. Ευχαριστώ. Κύριε Κώστα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι Mm. πολύ συγκεκριμένη στην παρέμβασή μου. Καταρχήν μια ε, σύντομη ε, ε, παρατήρηση. Ήθελα να πάρω το λόγο νωρίτερα, αλλά ε, τώρα ήθελα οπωσδήποτε να πάρω το λόγο. Τον Γενάρη του 2011 άκουσα την παρουσίαση της Ουγγρικής Προεδρίας και έκανα και μία ομιλία στην οποία καταδίκασα το κυνήγι μαγισσών κατά της κυβέρνησης ε, της Ουγγαρίας. Και τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε. Δεν ε, κρίνεται τη χώρα μας με βάση τα γεγονότα. Και ακούω τους συναδέλφους μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νιώθω ότι δεν έχει νόημα να γυρίσω στην πατρίδα μου, τα παιδιά μου να μην τα στείλω στο σχολείο, διότι είναι τόσο κακή η κατάσταση. Οι δηλώσεις που κάνετε είναι γελίες. Ε, ε σοκάρομαι που ακούω αυτά που μου λέτε. Και όταν επιστρέφω στην πατρίδα μου, τι βλέπω. Βλέπω δημοκρατία, βλέπω ελευθερία λόγου και βλέπω ότι δεν ε, είναι βάσιμες ε, οι ανησυχίες σας. Και όταν μιλάμε για πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρίες, ε, όταν μιλάμε για διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πού είσαστε εσείς. Ακούω τους εκπροσώπους του πάνελ. Δείξτε μου μία χώρα που να έχει ενσωματώσει στο δίκαιό της ε, το χάρτη θεμελιωτών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ε, χρήση της ε, νοηματικής στην νομοθεσία. Ποιε είναι οι σα, σα, ε, λοιπόν όταν μιλάμε για τα δικαιώματα ανθρώπων με ε, αναπηρίες ε, και όταν μιλάμε για την επικύρωση τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει επικυρώσει, τέσσερι χώρε όμω όχι. Και επίση όσον αφορά την Ουγγαρία, ο νόμο εκεί προστατεύει τα παιδιά, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένου και του ανθρώπου με αναπηρίες. Αυτά αναφέρονται στο Σύνταγμα μόνο, μία, μόνο σε άλλη μία χώρα προστατεύονται οι άνθρωποι με αναπηρία, στη Γερμανία. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ε, ευχαριστώ κύριε Μπρόμς. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, αναρωτιέμαι μήπως το Συμβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα έπρεπε να ε, κυνηγάει το, Βέλγιο που απαγόρευσε ένα μεγάλο κόμμα ή τη Γερμανία που θέλει να απαγορεύσει ένα μικρό. Ε, τι γίνεται με την γενοκτονία των ε, Αρμενίων και την, τι γίνεται με, όταν καταδικάζονται ερετικές ιστορικές θέσεις. Έχω πολύ λίγο χρόνο, αλλά ε, υπάρχουν ε, κάποιοι που ε, αναφέρονται και στο Ισλάμ. Το Συμβούλιο ή η ευρωπαικη Ένωση επέκριναν την βία κατά των, αυτών που διαμαρτύρονταν των διαδηλωτών στην Ουγγαρία. Επέκρινε το το Ηνωμένο Βασίλειο που άφησε ένα κόμμα να ε, διορίσει υψηλούς δικαστικού εξωματούχου. Οι απαντήσεις όλα αυτά είναι όχι. Ε, δεν μιλάμε για την υπεράσπιση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ε, εάν εγώ ήμουνα η κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα έλεγε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης να συγγυρίσουν πρώτα το δικό του σπίτι και τα κράτη-μέλη και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των διαφωνούντων στα κράτη-μέλη και μετά να κοιτάξουν την Ουγγαρία. Μέχρι τότε θα πρέπει να θα πρέπει η Ουγγαρία να, ε, να περιφρονεί όπως, ε, όπως τους αξίζει ε, τα θεσμικά αυτά όργανα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έχουμε μείνει πίσω τουλάχιστον μια ώρα στο πρόγραμμα. Παρακαλώ. Ωραία, μόνο ερωτήσει θα κάνω. Σα το υπόσχομαι. Σα δείχνω κάποια άρθρα του τύπου. Είναι από ένα χρόνο πριν. ουσιαστικά κενά. Και μετά βλέπετε να γράφουν τέρμα φημώθηκε ο τύπος, η ελευθερία ε, έκφρασης δεν υπάρχει πλέον στην Ουγγαρία. Κανένα από τα έγγραφα κανούν. Καμία εφημερίδα που ε, ασκεί κριτική, ασκούσε κριτική δεν έχει κλείσει. Εξακολουθούν να εκφράζουν τις απόψει τους. Κυρία Γκέντς που δεν τη βλέπω εδώ. Ε, ήθελα να της απαντήσω. Οι σοσιαλιστές είχαν ε, υποστηρίξει για την ε, θητεία του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου και ότι έλεγαν ότι έπρεπε να έχει πενταετή εμπειρία κτλ. Τώρα γιατί λένε ε, άλλα πράγματα. Α, ήρθε η κυρία Γκέντς για να απαντήσει και στο ερώτημά μου. Γιατί, επαναλαμβάνω, είχαν υπερψηφίσει την πρόταση στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου Σοσιαλιστές. Επίσης, ο κύριος Βέμπερ θέλω να μου απαντήσει. Ξέρετε ε, πώς λειτουργεί το δικαστικό σώμα, τι λέει ο νόμος και αν όχι διαβάστε το γιατί για 30 χρόνια μπορεί η εισαγγελία να ε, μεταφέρει σε ένα άλλο δικαστήριο μια υπόθεση εφόσον το επιθυμεί. Και όπως ε, την κυρία Βέμπερ άλλο ένα ερώτημα. Υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό νομοθέτημα που να απαγορεύει την άσκηση δημόσιου αξιώματο από οποιονδήποτε επειδή είναι νυφημένο ή νυφευμένη με ευρωβουλευτή. Υπάρχει νομοθεσία. Αν ναι, να σας ζητήσω δημοσία συγγνώμη, εδώ και τώρα. Αν όχι όμως, πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη στους θυγόμενους από αυτό. Προσβάλλετε συνεχώ τη δημοκρατία, ακούγεται μια φωνή. Η κυρία Ιντεβέλτ. Θα ήθελα συντομία να απαντήσω στον κύριο Σάιερ. Θα του στείλω την πηγή. Είναι το περιοδικό της καναδικής κυβερνήσεως ή των καναδικών πρεσβειών, πιο ακριβώς. Δεν ήταν δήλωση, εγώ έβαλα ερώτηση που υπέβαλα στον αντιπρόεδρο τη κυβερνήσεω δεν πήρα απάντηση. Δύο ερωτήσει το έθεσα και δεν απαντήθηκαν. Οπότε ψάχνω στοιχεία αλλά δεν παίρνω απαντήσει. Και θα εξακολουθώ να ψάχνω. Δεύτερον, πολλέ παρεμβάσει έκαναν συνάδελφοι του ΕΛΚ που διατείνονται ότι αυτό αυτό το θέμα κινείται για πολιτικούς σκοπούς και στρέφεται κατά της Ουγγαρίας. Ίσως εν μέρη να έχουν δίκιο. Δεν νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ήταν 100% συνεπέ καταγγέλλοντα κάθε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν δείτε το δικό μου ιστορικό και του κόμματό μου, ε, θα δείτε ότι έχουμε υποβάλει αμέτρητες κοινοβουλευτικές ερωτήσει για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος και αρκετές αφορούν την ίδια τη χώρα μου. Άρα είμαστε πολύ συνεπείς και νομίζω ότι πρέπει να εκφράσω τη λύπη μου που αφορά μόνο την Ουγγαρία. Υπάρχουν και σε άλλε χώρε προβλήματα, δίκιο έχετε. Αλλά τα προβλήματα που έχουν σωρευτεί στην Ουγγαρία είναι πολύ σοβαρότερα. Και ότι, ότι μόλις τώρα τα συζητάμε δείχνει ότι η Ευρώπη οριμάζει σαν κοινότητα αξιών. Έπρεπε να το είχαμε κάνει κατά το παρελθόν, κάλιο αργά παρά ποτέ όμως. Θα πρέπει να αρχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Εντφέλτ. Κύριε Ζάιερ, ήμουν ηρωνικός όταν ανέφερα την τεχνική της γαλάζιας κάρτας που ε, ισχύει για όλο το κοινοβούλιο, για την Ολομέλεια και όχι για την Επιτροπή. Πρέπει κάπως να συμμαζέψουμε την κατάσταση. Αν επιτρέπαμε τώρα γαλάζιες κάρτες, θα χάναμε τον έλεγχο της συνεδριάς, θέλει να πει ο Πρόεδρος. Και γίνεται και διάλογος εκτός μικροφώνου που δεν ακούμε. Πρόεδρος, δεχόσαστε απάντηση. Θα απαντήσω αγγλιστή για να μην έχουμε προβλήματα και παρεξηγήσεις. Το ερώτημά μου δεν ήταν αυτό. Αμφισβητώ ότι αμφισβητώ τις πηγές σας. Ερώτηση. Πριν από πέντε χρόνια, όταν η Καναδέζικη κυβέρνηση εισήγαγε την απέτηση για θεωρήσεις διαβατηρίων κατά των Ούγγρων και των Ούγγρων πολιτών λόγω των χιλιάδων Ρώμα που πήγαν στον Καναδά στα, όταν ήταν η σοσιαλιστική φιλελεύθερη κυβέρνηση. Πώς θέσατε τότε το πρόβλημα. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Το καινούριο φαινόμενο ότι ο αριθμός εκείνων που πηγαίνανε ε, μειώθηκε. Τι σχόλια κάνετε τότε θέλω να ακούσω. Επεκρίνατε τη σοσιαλιστική φιλελεύθερη ε, ουγγρική κυβέρνηση που προξένησε τη φυγή των Ρωμά πρόεδρος. Νομίζω ότι αναφέρθηκε, δεν χρειάζεται απάντηση αυτό που είπατε. Παρακαλώ, λέει ο πρόεδρο, η κυρία Ιντβελτ, που άμα πολύ σύντομη. Θα είστε σύντομοι. Πρώτα απ' όλα, γενικό σχόλιο. Δέχομαι ότι δεν καταγγείλαμε κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και δεν έχουμε πάντα επίγνωση όλων των παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε λησμονήσει, δεν έχουμε δει πολλά με την πάρα των ετών. Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, τα στοιχεία που έχω προέρχονται από το 2008 μέχρι το 2011, Νοέμβριο 2000, μέχρι Νοέμβριο 2011. Άρα επί του Φίντις ε, περισσότερο. Φέντης. Επί του Φίντες, επί κυβερνήσεως Φίντες, το περισσότερο κομμάτι. Όσον αφορά τη Βίζα, ε, πάντα λέγαμε ότι θα έπρεπε ε, είτε είπα είτε ο Καναδάς να αντιμετωπίζουν όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τον ίδιο τρόπο. Ήμασταν στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης δεν κάναμε ποτέ διάκριση κατά κανενό. Κυρία Λούνατσεκ, μισή λεπτό παρακαλώ, είστε σύντομη. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Λοιπόν, θα ήθελα σαν πράσινη να πω ότι θέλω να μιλήσω στεναρά κατά της παράλογης ιδέας του να υπάρχει συνωμοσία φιλελεύθερη σοσιαλιστική κατά ζωγκαρία. Είμαι πράσινη, ποτέ μου ποτέ φιλελεύθερη, ποτέ συντηρητική. Αλλά διατείνομαι ότι εκείνοι που δεν είναι από αυτές τις δύο ιδεολογικές ε, τάξεις μπορεί να είναι κατά αυτών που συμβαίνουν στην Ουγγαρία. γιατί αυτά από το... Λόγω αυτών που ακούμε από αυτούς που είναι στην Ουγγαρία. Και το LNP, η πράσινη της Ουγγαρίας, ε, που μπήκε το 2006, ε, της η κυβέρνηση γιατί την επέκρινε. Είναι αδελφό μας κόμμα και επέκριναν. Πήγαν στο κοινοβούλιο στις 23 Δεκεμβρίου και είπαν το Κοινοβούλιο εξαιρείται και αντιπολίτευση εξαιρούνται από τη δυνατότητα συμμετοχή. Λοιπόν, μην μιλάτε για αυτή την ιδέα τη συνωμοσία ε, φιλελευθέρων σοσιαλιστών. Ή περίφημο ε, καλλιτέχνε, Άνταν Φίσερ ή το Γκεφι, που έστειλαν επιστολέ στο ΕΛΚ. Ανήκουν σε ιδεολογική ομάδα οι καλλιτέχνε αυτοί. Όχι, είναι διάσημοι καλλιτέχνε που φοβούνται για τα τεκτενόμενα στην Ουγγαρία και ζητούν να γίνει κάτι. Λοιπόν, μην μιλάτε για αυτό σα παρακαλώ. Και ο Μπαρόσο, η Άσο κόρη κυρία Μέρκελ ε, και πολλοί άλλοι αναφέρθηκαν, οι οποίοι είναι από του συντηρητικού, από τη δική σα πολιτική ομάδα που επεκρέθησαν. Λοιπόν, ακούστε και αυτού αν δεν θέλετε να ακούσετε του άλλου. Αλλά εφόσον έχουμε εδώ κόσμο στο πάνελ, θα ήθελα να σα ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, προ τον κύριο Κάτινγκ, αναφερθήκατε στο εκλογικό, στον εκλογικό νόμο. Μπορείτε να μα πείτε τι απάντηση σας εδόθη. Από ό,τι κατάλαβα είναι απλώς κολυσιεργία, κολυσιεργία ε, κάνουν. Προσπαθούν και δύο επόμενες αγορές. Κύριε Ζερόμ, αναφερθήκατε στη διαδικασία του άρθρου 7. Είπατε ότι είναι πολιτική απόφαση. Θα μας συμβουλεύατε να προχωρήσουμε, γιατί νομίζω θα έπρεπε, αλλά θα ήθελα να ακούσω... Εσείς τι έχετε να μας πείτε. Κυρία Μπάουερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ ουγγρικά. Θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω ότι θα μάθουμε πολλά από τούτη την ακρόαση. Νομίζω ότι το Προεδρείο της Επιτροπής ε, θα πρέπει να μάθει κάποια πράγματα. Αυτό που με εκπλήσει, που δεν το γνώριζα, είναι ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης εκδίδει έγγραφα τα οποία θεωρούνται υψηλότερα στην ιεραρχία από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την Επιτροπή της Βενετίας, τι γίνεται με τις άλλες ε, με τα άλλα ε, ψηφίσματα της Επιτροπής αυτής. Θα πρέπει να εφαρμοστούν και αυτά και η Κομισιόν θα ζητήσει και εφαρμογή των άλλων συστάσεων της Επιτροπής της ε, Βενετίας. Ε, τότε θα χαρώ πολύ διότι έτσι θα δούμε θετικές αλλαγές. Μια άλλη ερώτηση που θα ήθελα να θέσω είναι η εξής. Μέχρι σήμερα πίστευα ότι η Ουγγρική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επικοινωνούν πολύ καλά μεταξύ τους με βάση αυτά που άκουσα από την Έλλη Κρούς. Και αποδεικνύεται τελικά ότι ναι, επικοινωνούν. Εγώ νόμιζα ότι εμείς είμαστε διαμεσολαβητές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αλλά αποκαλύπτεται τελικά ότι εμείς είμαστε ε, παράγοντες σε ένα πολύ περίεργο έργο, σε ένα, ότι είμαστε ηθοποιοί σε ένα περίεργο έργο. Δεν ξέρω πόσες φορές θα πρέπει να το ανεβάσουμε, αλλά όλα αυτά είναι ταπεινωτικά. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό. Η Επιτροπή μας τι ρόλο παίζει διότι δεν νομίζω ότι πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται οι ε, συνεδριάσεις ε, των επιτροπών ε, για τέτοιους στόχους. Κυρία Μπάουερ, είμαστε κοινοβούλιο και ακούμε αυτά που θέλουν να πούνε τα πολιτικά, οι πολιτικές ομάδες που συμμετέχουν. Συζητάμε είναι δημοκρατική απόφαση να συζητάμε τα θέματα αυτά και αυτός είναι ο τρόπος που τα συζητάμε. Έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει η κατάχρηση αυτής της ε, ακρόασης και της Επιτροπής μας. Βλέπω την κυρία Κόνς και την κυρία Βέμπερ. Σας παρακαλώ να είστε σύντομες, διότι ε, απαντάτε σε ερώτηση που σας τέθηκε. Θα απαντήσω στην ερώτηση που μου τέθηκε. Δεν ήμουν παρούσα, αν κατάλαβα σωστά όμως ε, τον κύριο Άντρας. Ε, το ερώτημα ήταν γιατί εμείς οι σοσιαλιστές ε, στηρίζουμε την τροποποίηση του συντάγματος σχετικά με την πενταετία και τους δικαστές. Το θέμα αυτό αφορά τον κύριο Μπόκο. Ε, η Τίλα τη οποία το όνομα αναφέρθηκε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική εμπειρογνώμονα. Ε, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα γραφείο στο οποίο έχει συγκεντρωθεί πολλή εξουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα με το Εθνικό Δικαστικό Γραφείο και έχει διοριστεί ε, κάποιο, κάποιο πρόσωπο που βρίσκεται πολύ κοντά στο κόμμα του Φίντες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε με ρώτησαν σχετικά με το παράδειγμα της Γερμανίας και νομίζω ότι η διαφορά είναι ακριβώς αυτή που ανέφερε ο κύριος Χίρου. Ας κοιτάξουμε την ευρύτερη εικόνα, όχι μόνο τα μικρά κομματάκια της εικόνας, διότι αν συνδέσουμε τα κομμάτια νομίζω η εικόνα είναι διαφορετική από ό,τι στη Γερμανία. Το γεγονός ότι αναφέρθηκα στον διορισμό του Πρόεδρου του Εθνικού Δικαστικού Γραφείου Ανέφερα ότι αυτό μπορεί να μην είναι νόμιμο, αλλά ε, πού είναι η ηθική νομιμότητα. Μπορεί να μην υπάρχει νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει όμως ε, ε, κάποια ε, ηθική όσον αφορά τον διορισμό ανθρώπων σε δημόσιες θέσεις. Και όταν ρώτησα πώς αντέδρασε το Κοινοβούλιο σε κάποια άλλα θέματα. Να πω ότι η κυρία Κίνεγκαρτ ήταν ε, ε, η συγγήτρια για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί αποφάσισε να μην εξετάσει όλες τις περιπτώσεις ε, και να σοπάσει για τα θέματα αυτά. Είδα κάποια χέρια. Κυρία μαλαβεζάτ; ζητήσατε το λόγο, κυρία βεζάτ; Είναι διαδικαστικό. Πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι. Επιμένω. Κύριε Φερξιά, εμείς δεν κάναμε του του αγόρευσης. Ε, αντιθέτως, ε, άλλες ομάδες το έπραξαν. Είναι λίγο τη τέτοιου είδου ε, ακροάσει, αν μετατρέπονται σε διάλογο μεταξύ ΕΛΚΑ σοσιαλιστών. Α σεβαστούμε έστω κατά το ελάχιστο του ανθρώπου που έχουμε προσκαλέσει. Διότι είναι ε, πραγματικά σουρεαλιστική αυτή η συζήτηση. Και μάλιστα βλέπουμε συναδέλφου ε, που δεν βλέπαμε συχνά στην Επιτροπή μα να παίρνουν για το λόγο. Ο πρόεδρος. Εμείς πρέπει να ε, αναλάβουμε την ευθύνη για τη δεξαγωγή των ακροάσεων. Και πρέπει να σας πω ότι δεν μίλησε μόνο η Σοσιαλιστική Ομάδα και το ΕΛΚ, μίλησαν πράσινοι, μίλησαν φιλελεύθεροι, ε, μίλησε η Γκούε. Έχει δοθεί ο λόγος σε όλους. Σας υπενθυμίζω, και όλοι θα λάβουν το λόγο, σας υπενθυμίζω ότι είναι σημαντικό να μένουμε σε ερωτήσεις και να μην κάνουμε διαλέξεις. Επανέρχομαι στο πάνελ στα μέλη του πάνελ. Με την ίδια σειρά όπως και την πρώτη φορά. Ναι, να απαντήσω για την Επιτροπή της Βενετίας πρώτα απ' όλα κάποιες ερωτήσεις και πώς αποφασίζουμε τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Είτε λαμβάνουμε άμεσα αιτήματα από την οικία χώρα σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο νομοθέτημα ή η κοινοβουλευτική συνέλευση, την οποία απαρτίζουν αιρετοί βουλευτές από την κάτω ή άνω βουλή, μας ζητά να κάνουμε ε, γνωμοδότηση. Με αυτό στους δύο τρόπους επιλέγει η Επιτροπή της Βενετίας ποια θέματα θα την απασχολήσουν και κάνει ανεξάρτητη επιλογή μάλλον δεν κάνει ανεξάρτητη επιλογή και επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη χώρα. Τώρα το κατά πόσον έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στην Ουγγαρία. Ουσιαστικά δεν λειτουργεί έτσι η Επιτροπή της Βενετίας. Αφού γνωμοδοτήσει για το Σύνταγμα, γιατί αυτό μα ζητήθηκε τότε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, μετά, ε, αφού έγινε αυτό, λάβαμε οκτώ αιτήματα. Τρία από τι Ουγγρικέ αρχέ υπήρξε ανταλλαγή επιστολών με το Γενικό Γραμματέα και πέντε αιτήματα από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση. ουσιαστικά κοινοβουλευτική συνέλευση είναι αυτή που αν μπορούμε να πούμε μας ζητά να, αποκομίσουμε, να ε, δημιουργήσουμε μια συνολική εικόνα. Θα επισκεφθούμε τη Βουδαπέστη στις 16 και 17 Φεβρουαρίου για να τεκμηριώσουμε την απόφαση και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τη διαδικασία. Νομίζω ότι κάλυψα αυτά που με ρώτησαν. Να πω και κάτι γενικότερο. Φυσικά το Συμβούλιο της Ευρώπης παράγει εκθέσεις, δηλώσεις ε, και κρίσεις και ε, από το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, σε σχέση με υποθέσει που αφορούν και τα 47 κράτη-μέλη μας. Ε, ίσως να μην ε, την χάνουν τις ίδιες προσοχές, τις προσοχές που θα άρμοζε όλες αυτές οι ε, υποθέσεις. Αλλά δεν επικεντρωνόμαστε εμείς σε συγκεκριμένα... Α, για το εκλογικό νόμο. Θέλετε να αναφερθώ στον εκλογικό νόμο, ναι. Ο εκλογικός νόμος ήταν ένας από τους τρεις τομείς που πρότεινε ο Γενικός μας γραμματέα στι Ουγγρικές Αρχές ε, να προσφύγουν στη βοήθεια της Επιτροπή Βενετίας και συμφώνησαν οι Ουγγρικέ Αρχές, άρα ε, θα έχουμε σχετική γνωμοδότηση και θα εγκριθεί μάλλον τον Ιούνιο η γνωμοδότηση από την Επιτροπή της Βενετίας. Ζερόμ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας ε, και κάποιες ε, ερωτήσεις. Καταρχήν η Ρανάτε Βέμπερ ε, ρώτησε πολύ συγκεκριμένα σχετικά με τον Ισαγγελέα και την περίπτωση να ανατίθενται υποθέσεις καθώς και τις διαδικασίες διορισμού. Νομίζω ότι αυτό που αναφέρατε εδώ είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί και ήταν και η ουσία της παρέμβασής μου. Ε, έχουμε την ε, πολυπλοκότητα όλων αυτών των διαφορετικών στοιχείων και ναι, αν, καν, ε, κάνει κανείς κάποια σύγκριση σε όλη την Ευρώπη θα, δει, θα βρει χώρες όπου γίνονται τα πράγματα αυτά με το συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορεί να αποφύγει λοιπόν κανείς να εξετάσει τη συνολική εικόνα. Και ήλπιζα ότι η Επιτροπή της Βενετίας θα είχε εξετάσει τα θέματα αυτά μπορεί να διαπιστώσουμε ότι έχουμε κενό εδώ. Αν δούμε ότι έχουμε ετήσια υποβολή εκθέσεων σε κάποιες από τις ε, βασικές ε, τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 2, ώστε να μπορεί να εξετάσει κανείς τις βασικές τάσεις. Μπορούμε να αντιστρέψουμε και τα θέματα. να πούμε ότι κάποια τέτοια ε, στοιχεία τα βρίσκουμε και σε άλλες χώρες, αλλά μπορεί η νομική του τάξη να έχει καθιερωθεί πριν 10, 20, 30 χρόνια. Τι μπορεί να κάνει κανείς σε μια νέα δημοκρατική εποχή όπου έχουμε μάθει πολλά από το παρελθόν. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κενό, ε, δεν μπορούμε όμως να αποφύγουμε την συνολική εικόνα. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, που είχε να κάνει με τις συμβουλές μου προς το Κοινοβούλιο, δεν νομίζω ότι θα έδινα πολύ αναλυτικές ε, συμβουλές είναι σε μεγάλο βαθμό δική σας απόφαση, αλλά κοιτώντας το θέμα από τη δική μου θέση, νομίζω ότι είναι, πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τονίστηκε και από αρκετούς από τους ομιλητές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα ε, κράτους δικαίου να συζητιούνται σε τούτο εδώ το φόρουμ και να ε, τα εξετάζουμε σοβαρά. Ε, υποβάλλουμε κάθε χρόνο ε, από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, μία ογκώδη έκθεση όπου εξετάζουμε διάφορα θέματα και θέλουμε να προσθέσουμε έτσι, να συνεισφέρουμε στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση όμως δημοσιεύουμε και εκθέσεις για συγκεκριμένα θέματα. Πέρα από τη γενική συζήτηση εδώ υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένε διαδικασίες ε, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει το άρθρο 7, η διαδικασία ε, παρέμβασης το αν ε, θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένε διαδικασίες, νομίζω ότι θα το αφήσω σε εσά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόρεν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε. Είπατε ότι πρέπει να εργαστούμε, ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα βάσει στοιχείων. Αλλά μετά μπήκατε σε πολιτικά επιχειρήματα, είπατε τι γινόταν την περίοδο των σοσιαλιστών, πώς είναι η κατάσταση τώρα. Για μένα αυτό δεν παίζει ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι ποτέ δεν θα έπεφτα σε αυτή την παγίδα των συγκρίσεων διαφόρων πολιτικών κομμάτων ή κυβερνήσεων για να θέσω θέματα ελεύθερης έκφρασης, ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και ελεύθερη ροής πληροφοριών. Ο Μίκρος Χαράστη, προκατοχό μου, έθεσε θέματα που σχετίζονται με την ελευθερία του λόγου κατά διάρκεια της εντολή του, της θητεία του. Εγώ πήγα στη θέση μου το 2010 και σας διαβεβαιώ ότι κάθε θέμα που συζητούμε σήμερα, και όχι μόνο για την Ουγγαρία, για την άρνηση της γενοκτονίας στη Γαλλία, εκφράσαμε κάποια θέση και για άλλα θέματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση που δεν εξετάσαμε. Δεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τα κράτη-μέλη, τα κράτη που συμμετέχουν ε, στον ΟΑΣΕ. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιστρέψουμε στα στοιχεία και να μην δίνουμε πολιτικό χαρακτήρα. Ελεύθερη έκφραση, ελεύθερη ροή πληροφοριών, ελεύθερα μέση, μέσα ενημέρωση είναι όλα σημαντικά ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και πολιτικών κομμάτων που δημιουργούν προβλήματα Αυτά και ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο. Στη δεύτερη ομάδα, στο δεύτερο πάνελ, δεν θα είναι λιγότερο έντονο από το πρώτο το πάνελ. Πάμε παρευθύς στο τρίτο και τέταρτο πάνελ, αυτό το δεύτερο πάνελ. Σε συνδυασμό, σε κοινό, μεικτό συνδυασμό. Αλλιώς μπλέξαμε δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Καλό λοιπόν τους εξή. Τους διακεκριμένους τους κεκλημένους μας. Mr. Lajos Association. Πρόεδρο της Ένωσης των Ουγγρών Δικαστών. Mr. Sultan sociologist. Κοινωνιολόγο και νομικό. Mr. Andras Arato, ναι. President of Πρόεδρο του Κουμπλεατόρ του Κουμπ Ράδιο. Του Κλουμπ Ράδιο. Mr. Balas Denes, representative of the Hungarian... Εκπροσωπεί την Ένωση, την Ουγγρική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών. Και ο Τίλα Κόπιας, ο κ. Ατήλα Κόπιας, δραστήριο μέλος, ακτιβιστής Προσπαθούμε να οργανώσουμε εδώ το πάνελ, ούτω ώστε όλοι οι διακεκριμένοι προσκεκλημένοι που μας συνοδεύουν να χωρέσουν. Να μπορέσουν να μιλήσουν. Παρακαλώ ησυχία όμως, ε. Θα ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό. Τρίτο και τέταρτο πάνελ, ομού. Θα τους δώσω με τη σειρά το λόγο και μετά θα έχουμε τελικό γύρο ρώτα απαντήσεων. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Κάθε πολιτική ομάδα θα έχει την ευκαιρία, θα έχει λόγο και μετά να σας θυμίσω ότι πρέπει να τηρούμε το χρόνο. Ο κύριος Μπάλας δεν ξεκινά, γιατί πρέπει να φύγει βλέπετε. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Μην του φύγει μάλλον η πτήση, μην του ξεφύγει η πτήση. Λοιπόν, ο πρώτος θα μιλήσει, ο κύριος Μπάλας Ντένες, και μετά θα ακολουθήσουμε την προβλεπόμενη σειρά, όπως την είχαμε στην μέση διάταξη. Ο κύριος Μπάλας Ντένες εκπροσωπεί την Ουγγρική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών. Κύριε Ντένες, έχετε το λόγο. Το πολύ δέκα λεπτά, ε. Αλλά αν μπορείτε και λιγότερο χρόνο, χάρη θα μας κάνετε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Να συνοψίσω τι γίνεται με το κράτο δικαίου και τα διάφορα προβλήματα στην Ουγγαρία σε 10 λεπτά είναι σαν να παρουσιάσω Σέξπιρ όλο το έργο του Σέξπιρ σε 10 λεπτά. Περνάμε δύσκολου καιρού όλη στην Ευρώπη και στην Ουγγαρία. Ποιο είναι το θλιβερότερο. Ότι ένα ογκρικό κόμμα είναι στο κοινοβούλιο και οι διάφορε οργανώσει που σχετίζονται με το κόμμα μιλάνε συστηματικά ε, για τους Ούγγρους Ρωμά ότι είναι εγκληματίες ή ότι δεν βλέπουμε κάποια δράση νομική, πολιτική ή ηθική εναντίον του φαινομένου αυτού ούτε από την Ουγγρική κυβέρνηση ούτε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποιο είναι το πιο θλιβερό ότι μετά από 22 χρόνια μετά το τέλος του κομμουνισμού ένα μεγάλο ποσοστό από τα παιδιά των Ρωμά ε, είναι χωριστά από τον στα σχολεία. Και παρά αυτά που λέει η κυβέρνηση για τη σημασία που έχει ένταξη και ολοκλήρωση, είναι κανόνε για τη δημόσια παιδεία στην πράξη απλώ θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Η Ουγγρική κυβέρνηση και υπεύθυνοι των σχολείων εξακολουθούν θεωρούν ότι ξεχωριστή αλλά ισότιμη παιδεία είναι μια λύση. Όχι, δεν είναι. Και η μείωση του, της περίοδους υποχρεωτικής παιδείας απλώς θα κρατήσει ζωντανό το διαχωρισμό στην Ουγγαρία. Δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή τεράστια ποσοστά από την Ουγγρική κοινωνία είναι ρατσιστές και ξενόφοβοι και λένε έγκλημα τσιγκάνων και έχει γίνει σε καθημερινή χρήση. Ή όποιος τολμήσει να μιλήσει ή να δράσει κατά αυτής τοποθέτησης θεωρείται ότι είναι κατά της Ουγγαρίας. Αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση και θυμό για τους Ρωμά των ε, Ούγγρων. Ακούγομαι γιατί έτσι αισθάνομαι. Παρά τα στοιχεία, παρά την κοινή λογική, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας. Το θέμα των Ούγγρων Ρωμά. Είναι απελπιστική κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Παρά τούτο, κανείς εδώ σήμερα α, δεν υπάρχει που να εκπροσωπεί τους Ρωμά και να μιλήσει ειλικρινά. Και η νέα στρατηγική της κυβερνήσεως Ρωμά δεν ακολουθεί προσέγγιση και εργαλεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποιο είναι πιο ανησυχητικό λοιπόν, ότι η κυβέρνηση με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου του τελευταίους 20 μήνες συστηματικά επετέθηκε, σε κάποιες περιπτώσεις κατέστρεψε το σύστημα, το οικονομικό και τον ισολογισμό της χώρας και διόρισε τους ανθρώπους της επικεφαλής των ανεξαρτήτων φορέων ή διότι όλα αυτά έγιναν στο όνομα της αντιδιαφθοράς, κατά πολλής διαφορά τη πολιτική. Αν μιλάμε για νομοθεσία, Ποιο είναι το πιο απογοητευτικό και εκνευριστικό το, το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση έχουν, κενό, έχουν κάνει ένα κενό πλαίσιο νομοθεσία στην Ουγγαρία και έχουν σταματήσει την... δεν έχουν περιεχόμενο συζητήσει στο Κοινοβούλιο ή περηφανεύονται με τον χρόνο ρεκόρ με τον οποίο θεσπίζουν δευτερογενή και τριτογενή νομοθεσία. Τεράστια ταχύτητα θέση τη νομοθεσία και είναι αυτό, καθε αυτό τεράστιο πρόβλημα. Εννέα μέρε συζήτησε το νέο σύνταγμα το Κοινοβούλιο. Μας θυμίζει η δεκαετία του 50 η προπαγάνδα που ακούμε και η προπαγάνδα θα δώσει μεγαλύτερη νομιμότητα στο Σύνταγμα. Το 2011, μιλώντα ειλικρινά, το πρόβλημα δεν ήταν οι διαβουλευσει, το πρόβλημα ήταν να παρακολουθήσει κανείς τα τεκτενόμενα στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια από τα εξή είναι πιο συμβολικά. Ότι ο πρόεδρο του Ουγγρικού Κοινοβουλίου το περασμένο φθινόπωρο κάλεσε είπε ότι είναι μερικοί ε, τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Στασβούργο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι είναι ηλίθιοι ή ότι δεν κάνει τις νομοθετικές ε, αλλαγές που απέτησε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, μπορούν σε μερικές εβδομάδες με αυτή την ταχύτητα να αλλάξουν πολλές φορές το, το ε, Σύνταγμα. Τι είναι χειρότερο, το ότι κυβερνηση δεν μιλά ανοιχτά για τις νομικές συνέπειες της προστασίας, το διάταξη προστασία των εμβρίων στο Σύνταγμα ή που κάνει ελάχιστα για να βοηθήσει τις οικογένειες και τους εφήβους στις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Τι να πρωτοπώ. 15.000 άνθρωποι με πνευματικά προβλήματα ζουν σε μεγάλα ιδρύματα. Παρά τη δέσμευση που ανελήφθηκε πριν από 14 χρόνια για την να κλείσουν αυτά τα ιδρύματα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με πνευματικά προβλήματα δεν μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους ποιος θα τους φυλάει. Και έχει ποινικοποίησει ε, το, τους αστέγους η χώρα στην πράξη. 115 νέους νόμους θέσπισε και τροποποίησε 200. Αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση δεν δείχνει ότι θέλει να ρυθμίσει τη δραστηριότητα των λομπιστών. Κινούνται στη μαύρη και φαιά οι λομπίστες. Ο νόμος για τα λόμπι, ο παλιός, ήταν ο πρώτος που διαγράφει από το γκρικό σύστημα. Talking about the role of Europe. Τώρα όσον αφορά το ρόλο της Ευρώπης, σαν Ούγγρος και Ευρωπαίος πολίτης, δεν ξέρω τι είναι το πιο προβληματικό. Το ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να πιστεύει ότι ε, η διπλή γλώσσα, δηλαδή άλλα να λες και άλλα να εννοείς, μπορεί να ισχύει ή ότι τι πιστεύουν αυτά που λέει η οτι πιστευουν αυτα που λεει η κυβερνηση οι πολυψηφοφόροι. Ε, το να λέμε άλλα και να κάνουμε άλλα εξακολουθεί να ισχύει. Ο αντιπρόεδρο τη κυβερνήσεω τη χώρα φαίνεται να συμμορφώνεται με τα πάντα που του ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αυτό κατάλαβε τη συζήτηση. Χτε ο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν με, με οργή είπε ότι βασικά αυτό που συνέβη του πρόσφατου μήνε ήταν μια συνωμοσία κατά αυτού που συντονίστηκε από τους διεθνείς διπλωματικούς κύκλους που χρησιμοποίησαν τις διπλωματικές σχέσεις και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το CNN. Θεωρώ ότι αυτή είναι γλώσσα ψεύτικη, λέει ψέματα. Το πρώτο εξάμεινο του 2011 ήταν πολύ απογοητευτικό. Οι προσπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προάσπιση τη ελεύθερη έκφραση το Συμβούλιο τη Ευρώπη του ΑΣΕ και του ΟΗΕ στους περίφημους νόμους για τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, αλλά δεν κατάφεραν να κινητοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτό. Η κατάσταση τώρα είναι διαφορετική. Η προσοχή είναι η συμμετοχή, η πίεση χρειάζεται. Στο κάτω-κάτω, αν η, η Ουγγαρία ήταν τώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις με τη χώρα αυτή θα είχαν διακοπεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να καταλάβουμε τα εξή χωρίς τα σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα της χώρας και την απελπιστική ανάγκη βοήθειας του Δούνου του, δεν θα άκουγε τις επικρίσεις η Ουγγαρία. Δεύτερον, η χώρα θα πρέπει να λύσει τα πολιτικά της προβλήματα πρώτα απ' όλα, να λύσει τα του οίκου της. Χρειάζεται ψηφοφόρους που θυμούνται η Ουγγρική κοινωνία. Χρειάζεται κόμματα που δεν είναι διαφθαρμένα, χρειάζεται ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση και πρέπει να οργανωθεί βάση των αρχών της ανοιχτής κοινωνίας. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργό και κλείνω, πριν από λίγες μέρες στη Βουδαπέστη, σύγκρινε και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν το ενόπνευμα, το αλκοόλ. Δεν νομίζω ότι είχε δίκιο. Η κυβέρνηση και το κόμμα της Ουγγαρίας θεωρώ ότι είναι μεθυσμένοι σήμερα. Αλλά η χώρα θα αισθανθεί τον πονοκέφαλο μετά. Ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η νυφάλια φωνή σε αυτή την ιστορία. Και αν κρατήσουμε αυτή τη μεταφορά, φοβούμαι ότι σε αυτή τη φάση στην Ουγγαρία φαίνεται ότι η πολιτική εξουσία σε κάποιε περιπτώσει μοιάζει με ε, παρεστησιογόνα. Και όταν υποστηρίζεται από τα δύο του Κοινοβουλίου αυτή η εξουσία είναι σαν τα σκληρά ναρκωτικά. Και τα σκληρά ναρκωτικά, κυρίε και κύριοι, είναι εύκολο να τα αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρηση και πολύ εύκολο να προξενήσουν εθισμό. Η νυφάλια φωνή σα, χρειάζεται αυτέ τι μέρε. Ευχαριστώ την προσοχή σα. Ακούσαμε τον κύριο Ντενές και μου είπαν ότι θα πρέπει να αποχωρήσει πριν το τέλος της συνάντησης. Προχωράμε ε, με την αρχική ε, σειρά. Ο Λάγιος Μακάη, ε, πρόεδρος των Ούγγρων δικαστών. Το πολύ 10 λεπτά, αν μπορείτε να είσαστε πιο σύντομος, αυτό θα είναι καλό, διότι έχουμε λίγο πολύ μία ώρα και έχουμε έξι ομιλητές στο πάνελ και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό. Ε, θα θέλαμε να ακούσουμε και ερωτήσεις και απαντήσεις σας. Παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόκληση, πρόσκληση και την δυνατότητα να ε, ενημερώσω την ε, Επιτροπή Πολιτικών ε, Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με το δικαστικό σύστημα. Θα τονίσω κάποια σημαντικά θέματα. Η Ένωσή μας εργάζεται με βάση την εντολή που αναφέρεται στο καταστατικό της και το σχέδιο δράσης που υιοθετήθηκε το 2009. Ε, ε, ε, είχαμε μια συμφωνία με, την, με το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης και γι' αυτό μπορέσαμε να υποβάλουμε τη θέση μας σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Η Ένωσή μας ε, οργανώνει μια σειρά δημοσίων διασκέψεων για να ε, μάθει τη γνώμη των δικαστών και με βάση τις ε, θέσεις αυτές υποβάλλουμε προτάσεις στο Κοινοβούλιο. Εκατοντάδες δικαστή, δικαστές ήταν παρόντες στις διασκέψεις αυτές και πολλοί άλλοι μας έστειλαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις προτάσεις τους. Αρκετές προτάσεις έχουν υιοθετηθεί, υπάρχουν όμως και κάποια θέματα, κάποιες νομοθετικές λεπτομέρειες όπου η θέση της Ένωσής ήταν διαφορετική από από τα νομοθετήματα που τελικά υιοθετήθηκαν. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ένωσή μα ε, δεν ε, συμμετείχε στην σύνταξη του συντάγματο. Ε, διατυπώσαμε τις προτάσεις μας για το, τους κανόνες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των των δικαστηρίων ε, καθώς και άλλους κανόνες αφού ε, ολοκληρώθηκε το Σύνταγμα και γι' αυτό η Ένωση, ε, η Ένωση μας δεν είχε τη δυνατότητα να υποβάλει τη θέση της στους νομοθετές εκ των προτέρων όσον αφορά για παράδειγμα την μείωση του, ε, της ηλικίας συνταξιδότησης των δικαστών. και μάλιστα αυτό το μέτρο δεν το περιμέναμε, ήταν αναπάντεχο γνωρίζοντας ε, τη νέα νομοθεσία. Μαζί με τους επικεφαλής ε, των ε, δικαστηρίων υποβάλαμε τη θέση μας, στην οποία διαμαρτυρόμασταν κατά του μέτρου αυτού. Έχουμε κατά νου το Έχουμε κατά νου το ενδιαφέρον των ε, δικαστών ε, και γι' αυτό ζητήσαμε μεταβατική περίοδο ε, και ζητήσαμε κάποιο αντιστάθμισμα επειδή οι συντάξει των δικαστών είναι πολύ χαμηλές. Η πρότασή μας δεν έγινε δεχτή από τους νομοθέτες. Εμείς διατηρούμε την πρότασή μας. Θα ήθελα να πω ότι επειδή οι γενικοί κανόνες για, του, για ισχύουν και για τους δικαστές, οι δικαστές ε, που είδαν μείωση του χρόνου υπηρεσίας τους ε, είχαν ε, εδραιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και αρκετοί δικαστές ζήτησαν λοιπόν σύνταξη. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, όσον αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων και τις, αλλαγές, και τις σχετικές αλλαγές, η Ένωσή μας όπως ε, και ε, πανεπιστήμια και άλλα φόρουμ ε, επέκριναν την λειτουργία. Η Ένωσή μας συμφώνησε με τις επικρίσεις αυτές. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος Ζόλταν Φλέκ επέκρινε την λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Είπαμε ότι ούτε η σύνθεσή του ε, ούτε άλλοι παράγοντες ε, δεν καθιστούν ε, ικανό το Συμβούλιο αυτό να διαχειρίζεται σωστά τα δικαστηρία και γι' αυτό των δικαστηρίων και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Όσον αφορά την λειτουργία αυτού του φορέα, δεν είχε κατά νου το συμφέρον του του Κερσίνη στο σύνολό του, αλλά ατομικά συμφέροντα. Κατά 14 χρόνια λειτουργίας ε, δεν ήταν ε, δυνατόν να λυθούν τα προβλήματα που υπήρχαν. Για παράδειγμα, στην πρωτεύουσα και σε μια γειτονική περιφέρεια, οι δικαστικέ διαδικασίε ε, κρατάνε περισσότερο χρόνο από ό,τι σε άλλα μέρη τη χώρα Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που είναι η καθυστέρηση στις υποθέσεις, ο φόρτο από παλιέ υποθέσει ε, και ε, ο άνισος φόρτο εργασία δικαστών. Η προηγούμενη κυβέρνηση γνώριζε επίση τι ανομαλίε αυτέ και υπέβαλε διάφορε προτάσει σχετικά με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο. Είχαν ληφθεί κάποια βήματα για να ε, ε, αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Ε, προτάθηκε μια μεταφορά εξουσιών στον πρόεδρο της Ένωσης, κάτι που έγινε με τροποποίηση της πράξης για τη λειτουργία των δικαστηρίων το 2010. Το μέτρο αυτό σήμαινε ότι η ατομική ευθύνη ήρθε στο προσκήνιο. Ε, ο πρόεδρος του Γενικού Δικαστικού του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου ε, ανέλαβε τα, δικαιο, τις εξουσίες ε, με τη νέα νομοθεσία. Γι' αυτό το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο έχει μειωμένες εξουσίες. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου ε, Δικαστών και του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν κάτι που επίσης επικρίθηκε. Η ανάγκη να διαχωριστούν αυτές οι δύο θέσεις ε, ε, έγινε πιο πιεστική με το πέρασμα του χρόνου. Η πείρα μας μας δείχνει ότι το ε, ουγγρικό δικαστικό σύστημα δεν είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη και γι' αυτό Μάλλον δεν μπορέσαμε να βρούμε παρόμοιο σύστημα με το δικό μας στην Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη τις επικρίσεις αυτές, η Ένωσή μας πρότεινε μια νέα δικαστική δομή, όπου το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κεντρική διαχείριση των δικαστηρίων δεν είναι ο πρόεδρος του ανωτατάτου δικαστηρίου. Επίσης προτείναμε ένα σώμα που να εκλέγεται, το να αποτελείται από δικαστές ε, που να ε, είναι υπεύθυνο για την ε, εποπτεία. Ένας τέτοιος φορέας θα είχε δικαίωμα συνένεση σε κάποιε περιπτώσει, για παράδειγμα τους διορισμούς σε υψηλέ θέσει. Αυτή η δικαστική δομή αντικατοπτρίζεται στην νομοθεσία που υιοθετήθηκε. Από εδώ και μπρο, ε, ο πρόεδρος ε, του ε, Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου θα είναι υπεύθυνο για πολλά άλλα θέματα. Το Εθνικό Συμβούλιο Δικαστών είναι επίση ένα νέο φορέας που δημιουργήθηκε και είναι υπεύθυνο για την εποπτεία ε, των ε, δραστηριοτήτων ε, διαχείριση του Προέδρου του Εθνικού Δικαστικού Γραφείου. Η πρόταση της ένωσή μα ε, δεν έγινε αποδεκτή στο σύνολό τη, διότι εμείς προτείναμε να υπάρχει δικαίωμα συνένεση. Ε, στην ε, νομοθεσία όμως δίδεται μόνο δικαίωμα υποβολής νομοδότησης. Ενώ διάφορα δικαστικά σώματα διατηρούν το ε, δικαίωμά τους ε, να υποβάλουν ε, γνωμοδότηση όσον αφορά τον διορισμό δικαστών και άλλων. Αυτό σημαίνει ότι ακούγεται η φωνή των δικαστών. Σημαντικό είναι να πούμε ότι κατά τη διάρκεια υποβολής αίτησης, προτού να διοριστεί ένας δικαστής, ετοιμάζεται ένας σύντομος κατάλογος με βάση κάποια αντικειμενικά κριτήρια και ο πρόεδρος του Γενικού του, Εθνικού Δικαστικού Γραφείου, του, Εθνικού Γραφείου Δικαιοσύνη, ε, μπορεί να ε, επιλέξει έναν από τους ε, τρεις κορυφαίους δικαστές στον κατάλογο αυτών. Κανέναν άλλον. Πρέπει το πρόσωπο που τελικά θα διοριστεί να είναι ένας από τους τρεις στον κατάλογο αυτών. Επίσης, η διάσκεψη των δικαστών ε, υποβάλλει γνωμοδότηση σχετικά με τις ε, ίδιε τι αιτήσει. Πιστεύουμε ότι η ε, υποστήριξη της πλειοψηφία αυτών των φορέων εξασφαλίζει την νομιμότητα του ατόμου που διορίζεται και γι' αυτό η Ένωσή μας πρότεινε οποιοδήποτε δεν έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας να μπορεί να διοριστεί μόνο με μια προκαταρκτική συμφωνία του Εθνικού Συμβουλίου Δικαστών. Αντί για το δικαίωμα συγκατάθεση, ε, η νομοθεσία ε, συμπεριλαμβάνει δικαίωμα υποβολή νομοδότηση. Εμεί πιστεύουμε ότι. Όσον αφορά τους διορισμούς, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο να μπορούμε να συλλέξουμε εμπειρίε. Ε, αυτό δεν συμπεριλήφθηκε στη νομοθεσία στο παρελθόν. Πρόκειται για νέο αίτημα. Και συνήθως ε, κάποιος ε, πρέπει να έχει τριετή εμπειρία. οι πιο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο πρόεδρος ε, της Κούρια, πρέπει να έχουν εμπειρία πιο μακρά των τριών ετών. Εμείς προτείναμε οκταετή πείρα ως δικαστής. Αυτό όμως μειώθηκε στα πέντε χρόνια στην ε, νομοθεσία που ισχύει. Η Ένωσή μας ε, συμφώνησε τα δικαστήρια ε, να βοηθηθούν επειδή υπάρχει μεγάλος φόρτος παλιών υποθέσεων ε, ο οποίος θα πρέπει να μειωθεί. Και γι' αυτό πρέπει κάποιες περιπτώσεις ε, να ε, διαβαστούν σε άλλα δικαστήρια. Κάτι τέτοιο θα έδινε πολλές εξουσίες στην Κούρια. Δόθηκαν όμως πολλές εξουσίες τελικά στον πρόεδρο του Εθνικού Δικαστικού Γραφείου. Εμείς ε, δεν συμφωνούμε με την δυνατότητα του εισαγγελέα να, ε, ε να ε, παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε δικαστήριο, αλλά δεν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο περιορίζει την αντικειμενικότητα. Κατά τη γνώμη της Ένωσής μας, η παρούσα νομοθεσία που έχει να κάνει με το δικαστικό σύστημα δεν παρεμβαίνει στην ανεξαρτησία των δικαστών. Αυτό ισχύει παρότι δεν έχουν υιοθετηθεί όλες οι προτάσεις μας. Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι ε, σε τακτική βάση ε, γίνονται επιθέσεις στο δικαστικό σύστημα χωρίς αιτιολόγηση ε, και χωρίς αντικειμενική βάση. Η Ένωσή μας ε, εκπροσωπεί τα συμφέροντα του κλάδου και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τους ε, νομοθέτες στο μέλλον για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στον επόμενο μιλητή. Σας ευχαριστώ που κάνατε προσπάθεια να συνοψίσετε γιατί ήταν μεγάλη η αναφορά. Ο κύριος Σολτάν Φλέκ τώρα που είναι κοινωνιολόγος και νομικός. Παρακαλώ 10 λεπτά το πολύ. Μακάρι να τα περικόψετε κι εσείς τα 10 λεπτά. Θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερως. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που έχω επιλεγεί να μιλήσω σε αυτό το πάνελ εδώ στο επίκεντρο της ε, δημοκρατίας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στον τομέα που γνώριζω καλύτερα. Καταρχάς να πω ότι εδώ δεν μιλάμε συνολικά για την Ουγγαρία. Μιλάμε για τα μέτρα της Ουγγρικής κυβέρνησης. Μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά η Ουγγρική κυβέρνηση, τι αλλαγές έχει εισαγάγει στο πολιτικό σύστημα και, όπως λέει και ο τίτλος της ακρόασης, κατάσταση στην Ουγγαρία. Δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε νομικά ε, και νομικιστικά ζητήματα, αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική, τη δημόσια πολιτική. Γι' αυτό και πολύ σωστά συζητούνται αυτά τα θέματα σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Τη δική σας επιτροπή. Πρέπει να πω ότι στην ευρύτερη περιοχή έχουμε διάφορες περίεργες παραδόσεις και συνήθειες, κάποιες ε, είναι αξιέπαινες, κάποιες άλλες παραδόσεις όμως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κάποια προσοχή. Σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα, απαρτίζεται από δικαιώματα. Έχουμε την ε, αρχιτεκτονική που φαίνεται να είναι εντάξει. Υπάρχουν όμως μικρές στρεβλώσεις στους θεσμούς. Και αυτό το πρόβλημα είναι που οδηγεί σε αμφισβήτηση του όλου συστήματος, του όλου συντάγματος. Μια άλλη παράδοση είναι πώς χρησιμοποιούμε τον νόμο ως εργαλείο. Στους τελευταίους 18 μήνες, αλλά και τα τελευταία 20 χρόνια, αυτό έχει χαρακτηρίσει και την ουγγρική πολιτική. αν το επιθυμούν τα κόμματα που είναι στην κυβέρνηση, μπορούν να τροποποιούν το Σύνταγμα. Και το πράττουν αν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό. Τώρα λοιπόν που έχουν την πλειοψηφία των δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο, ε, οι κυβερνώντες του κόμματος Φίντες φυσικά είναι πολύ εύκολο να το κάνουν. Δεν μπορούμε βέβαια να τα βλέπουμε απομονωμένα ορισμένα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Είναι πολλοί αυτοί που και εδώ αλλά και στο διεθνή τύπο υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση ευρύτερη συνολική, ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα δηλαδή σφαιρικά. Και συμφωνώ και εγώ, όπως και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πει επανειλημμένω, ότι δεν είναι σωστό να γίνεται κατάχρηση τη πλειοψηφία των δύο τρίτων από το κυβερνών κόμμα Φιντές. Βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε απλουστευτικέ συγκρίσει. Για να έρθω σε κάποια πραγματικά περιστατικά, το 2010 το Γραφείο για τα Ανθρωπινά Δικαιώματα και το Ινστιτούτο Max Planck σε μια δήλωση. Μια δήλωση όπου γιατί πονάνε συστάσεις και υποδείξεις και έλεγαν ότι η, η ε, Ανατολική Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και ο Νότιος Κάφκος πρέπει να ακολουθήσουν ε, τις υποδείξεις για μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι θα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις μεταρρυθμίσεις αυτές, αν και όχι αποκλειστικό, όπως ισχύει σε άλλε χώρε, οι δικαστές. Οι συλλογικοί δικαστικοί φορεί. ότι θα έπρεπε, θα έπρεπε να διαδραματίσουν ρόλο στη διαχείριση τη δικαστική. Ποια είναι η λύση που θα μπορούσαμε να προτείνουμε. Οι διάφορες εξουσίες να επιμερίζονται σε διαφορετικούς φορείς. Αλλά δεν σκέφτηκε κανείς να συγκεντρώσει τις εξουσίες, όλες τις εξουσίες, μόνο σε ένα φορέα δημόσιο. Επανέρχομαι τώρα στο δικαστικό σύστημα της Ουγγαρίας, που είναι και ο ακρογωνίος λίθος της ένομης σε κάθε χώρα που κρίνει κατά πόσον υπάρχει κράτος δικαίου σε κάποια χώρα. Βέβαια, για να απαντήσουμε το ερώτημα αυτό, πρέπει να βλέπουμε γενικότερα πώς γίνεται η άσκηση της εξουσίας στη δεδομένη χώρα. Υπάρχει αλλαγή στην ανεξαρτησία ή στο καθεστώς αντικαθίστα επικεφαλής κάποιων οργανισμών. Γίνεται προσπάθεια να μην μπορούν να γίνουν αλλαγές στο μέλλον. Αυτά τα δύο τρίτα που ελέγχει αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο το κόμμα ε, ΦΙΝΤΕΣ πράγματι μπορεί να καθορίσει την αρχιτεκτονική ορισμένων δικαστικών φορέων. Σε ό,τι αφορά τώρα το δικαστικό σύστημα στην Ουγγαρία. Υπήρχε ένα συλλογικό σώμα λήψης αποφάσεων που έχει αντικατασταθεί από την ε, κεντρική πλέον διαχείριση. Και έχουμε ένα επικεφαλής που ελέγχεται για εννέα εκλέγεται, για, μάλλον ορίζεται για εννέα χρόνια και συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες που πριν το, τις είχε το συλλογικό ε, σώμα των δικαστών. Και φυσικά αυτό συνιστά αδιαφανή τρόπο λήψεως αποφάσεων. Αυτό αποφάσισε βέβαια η πλειοψηφία των δύο τρίτων. Δεν μπορεί κανείς όμως να το δεχθεί. Ο πρόεδρος της Κούρια και αυτός εκλέγεται από τα δύο τρίτα της πλειοψηφίας, όπως είπαμε, για εννέα χρόνια, αλλά μπορεί να παραμείνει αφού λήξει η εννέα του θητεία μέχρι ότου βρεθεί ο αντικαταστάτης του. σε ό,τι αφορά κάποιες κατώτερες βαθμίδες υποτίθεται ότι ελέγχουν τον πρόεδρο της Κούρια οι δικαστές αυτοί, αλλά το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να διατυπώσουν κάποια άποψη, κάποια γνώμη. Δεν υπάρχει διαβούλευση. στην Ουγγαρία, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κάποιο συλλογικό σώμα το οποίο να μπορεί να μεταφέρει τις επιθυμίες των δικαστών σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση των δικαστηρίων. Δεν υπάρχει τέτοιο φορές αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε. Μιλάω για τους δικαστέ πάντοτε. Δεν είναι θέμα διάκρισης σε σχέση δηλαδή με το υποχρεωτικό όριο συνταξιοδότησης. Απλά πρέπει να θυμίσουμε ότι ο δικαστής είναι ένα λειτουργήμα προστατευμένο. Την χάνει ιδιαίτερη ειδική προστασία. Φυσικά όλα μπορούν να αλλάξουν. Οι όροι εντολή των δικαστών μπορούν να τροποποιηθούν. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι θέτοντας σε κίνδυνο τα ίδια τα δικαστήρια. Το ίδιο ισχύει και με την αντικατάσταση του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, αυτού που αποκαλούμε Κούρια στη χώρα μου, που είναι και η ψηλότερη θέση στο δικαστικό σύστημα της Ουγγαρίας. Φυσικά και κάποιος μπορεί ε, να απομακρυνθεί από το αξιωμά του, αλλά στο μέσο της θητείας είναι σαν να παραγνωρίζονται όλοι οι νόμοι. Η ακαιρεότητα των δικαστών ουσιαστικά τίθεται σε κίνδυνο με αυτή την κίνηση. Η δικαστική εξουσία λοιπόν, που όπως είπα είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους, ίσως ο σημαντικότερος πυλώνας του συστήματος, αντιμετωπίζει τώρα τα ίδια προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζουν ε, άλλοι δημόσιοι λειτουργοί, με, δηλαδή χαρακτηριστικά την πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Τον έντονο κεντρικό χαρακτήρα. Το Κοινοβούλιο εκλέγει όλους τους ε, λειτουργούς, Φαίνεται όμως ότι τελικά ε, έχουμε την ε, ένωση των και όχι τη διάκριση των εξουσιών. Γυρίσαμε σε ελληνιστικές εποχές. Τώρα περνάμε στον κύριο ε, Λάνατο που είναι ο πρόεδρος του Club Radio. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ελπίδα παρά την τεράστια καθυστέρηση υπάρχει και ζωντανή μετάδοση στο Group Radio στη Βουδαπέστη Α μιλήσω ουγγρικά, διότι υπάρχουν κάποιοι ακροατέ του ραδιοφώνου που δεν κατανοούν τα αγγλικά και ζητώ συγγνώμη θα μιλήσω ουγγρικά. Σας ευχαριστώ. Πρώτη φορά όταν πέρασα τα σύνορα Ουγγαρίας και Αυστρία ήταν πάρα πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου. Δεν χρειάστηκε ούτε να γίνει έλεγχος διαβατηρίων ούτε να καθυστερήσω. Φαντάζεστε πόσο τιμή είναι για μένα να είμαι εδώ στην καρδιά ε, της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Είναι τιμή, αλλά όχι και ευχαρίστηση απαραίτητα που είμαι εδώ, διότι σε κανονικές περιστάσεις ένας μικρός επιχειρηματίας όπως εγώ από τη Βουδαπέστη δεν θα παρευρισκόταν εδώ για να συναντά τόσο διακεκριμένους πολιτικούς. Ο απλός άνθρωπος στο δρόμο ε, μπορεί να μοιραστεί ε, το φως των προβολέων μόνο σε κάποιο σοου σε reality. Ε, και το Κομπ ράδιο πολεμά για την επιβίωσή του. Στο reality του νόμου της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης. Όταν το Συμβούλιο το Παντοδύναμο για τα μέσα ενημέρωσης για να δώσει τις άδειες και να επιβάλλει κυρώσεις, αυτό ήταν προβλεπόμενο θα γίνει. Είχε μόνο μέλη ε, που ήταν υπέρ της κυβερνήσεως. Ε, και ενώ νομοθεσία ε, η Ευρωπαϊκή απαγορεύει μονομερή έλεγχο των μέσων ενημέρωση για να αποφευχθεί αυτό που μα συνέβη εμά στο Ράντιο. Ε, κεντρική μεροληπτική εποπτεία φημώνει τι ανεξάρτητε φωνέ των μέσων ενημέρωση. Βέβαια, μπορείτε να δώσετε παραδείγματα αντιπαραδείγματα θα έλεγα όμως, είναι φρικτό αυτό συμβαίνει. Το Κομπ δεν είναι το μόνο παράδειγμα του προβλήματος ασυνήθιστων φαινόμενων για την υπόλοιπη Ευρώπη ή την πολιτισμένη Ευρώπη, ας το πω έτσι. Θα ήθελα να εστιαστώ στο παράδειγμά μας. Να παρουσιάσω κάποιες ιδέες. Η οι δημοσιογραφικές υπηρεσίες ε, μπορούν να παρουσιάσουν ειδήσει που προέρχονται από επίσημε πηγές. Και αυτοί που απασχολούνται εκεί εξαρτώνται άμεσα από την εξουσία. Και παρουσιάζονται με μεροληπτικά ειδήσει όπως οι διαδηλώσεις κλπ. της αντιπολίτευσης. Συνήθως οι εταιρείε που είναι υπέρ τη κυβερνήσεω παίρνουν συχνότητε ραδιοφωνικέ. Οι κρατικοί φορεί, κυβερνητικοί φορεί δεν διαφημίζουν στου ανεξάρτητου σταθμού και οι ιδιωτικοί διαφημιστέ, αυτοί που θέλουν να διαφημίσουν οι ιδιωτικέ εταιρείε επειδή φοβούνται, ακολουθούν αυτή την προσέγγιση όσον αφορά τι διαφημίσει. Να συνοψίσω το τι συνέβη στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και έτσι θα καταλάβετε καλύτερα ποια είναι όλη η κατάσταση πιστεύω. Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως μου ζήτησε, μου έθεσε ένα ερώτημα μάλλον, να του πω κατά πόσο το Club Radio είναι ε, φωνή της αντιπολίτευσης. Όλα τα μέσα ενημέρωσης θα έπρεπε να είναι πηγές έκφρασης της αντιπολίτευσης ανεξάρτητα από το κόμμα που κυβερνά. Να συνοψίσω τι μας συνέβη. Τι είναι το Club Radio καταρχάς. Θεωρούν ότι είναι ο μόνος σταθμός, δημόσιος σταθμός στην Ουγγαρία που παρουσιάζει πολιτικά σχόλια, ο μόνος σταθμός, πολύ διακεκριμένοι δημοσιογράφοι έχουν τα προγράμματά τους, επικρίνουμε και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ασχολούμαστε με όλους τους τομείς της ζωής, από αθλητισμό μέχρι πολιτιστικά. Η μουσική είναι περίπου το 20% του συνολικού περιεχομένου και είναι δημοφιλής στους σταθμούς γιατί εκατοντάδες χιλιάδες συντονίζονται στη συχνότητά μας καθημερινά. Η άδειά μας η δωδεκαετής εξέπνευσε το Φεβρουάριο του 2011. Σύμφωνα με τον νόμο. Και τον παλιό και τον νέο. Αλλά η αρχή για τα μέσα ενημέρωσης θα έπρεπε να ξεκινήσει τη διαδικασία ανάθεσης πριν από 14 μήνες. Καθυστέρησε 14 μήνες, το κάνει 14 μήνες μετά και αυτό είναι κατά του νόμου. Λόγω της καθυστέρησης, της αδειοδότησης, αρχές του 2010 ζητήσαμε στο Club Radio άλλη συχνότητα στη Βουδαπέστη. Ενεκρίθη, νικήσαμε, αλλά το Συμβούλιο, το ραδιοτηλεοπτικό, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 2010. Τα αποτελέσματα και δεν ξέραμε αν θα επιβιώσουμε ή όχι. Είμαστε εν κενό. Προσφύγαμε στο δικαστήριο. Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου τέλος Φεβρουαρίου στο πρωτοδικείο, στην πρωτοβάθμια δικαιοσύνη. Κύριε Σάγερ, δεν ανανεώθηκε καμία συχνότητα του σταθμού μας. Έχουμε μια άδεια προσωρινή δίμηνη που αν, θα ανανεωθεί, αν ανανεωθεί. Μέχρι το φθινόπωρο του 2011 εκπέμπαμε σε 10 πόλεις περιφερειακές και σε 7 περιπτώσεις με διαφορετικές με διαφορετικές τεχνικές δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Σε τοπικό σταθμό έδωσαν πέντε συχνότητες, σε εμά κανένα. Αυτό ο ιδιωτικό σταθμό είναι κοινοτικό σταθμό και δεν πληρώνει άδεια. Και εκεί ακούγονται ομιλίε, συνομιλίε κλπ. Όταν ζητήσαμε ισότιμη αντιμετώπιση, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο είπε ότι δεν ε, τίθεται καν θέμα τέτοιο, δεν μπορούσαν να μα δώσουν παρόμοια αντιμετώπιση. Δεν ήταν σοβαρό το αίτημά μα. Α πάμε τώρα στο επίμαχο θέμα των 95,3 MHz ε, της συχνότητας αυτής και του διαγωνισμού για τη χορήγηση αυτής της συχνότητας. Χρησιμοποιούσαμε αυτή τη συχνότητα με δίμηνη προσωρινή άδεια, ανανεώσιμη. Άμα έχει δίμηνη άδεια, τι επιχειρηματικό μοντέλο να φτιάξει. Τον Ιούλιο του 2011 το Ραδιοτηλεπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία ανάθεση, αλλά υπό ποιου όρου, ποια κριτήρια τα κριτήρια ήταν τέτοια που θα καθιστούσαν ανέφικτοι, δεν θα ήμασταν επιλέξιμοι. Τα κριτήρια προτιμούσαν τοπικά νέα, μουσικό ραδιόφωνο, όσο χαμηλότερο το πνευματικό περιεχόμενο, περισσότεροι βαθμοί. Και το τέλος διπλασιάστηκε για την άδεια. 200.000 ευρώ το χρόνο. Βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε, ήμασταν έτοιμοι να συμβιβαστούμε. Κάναμε μια προσφορά και κανονικά το ραδιοτηλεπτικό συμβούλιο ακόμα και υπό τις αυστηρές συνθήκες θα μπορούσε να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε. Ε, δεν συμπεριλάβαμε περιεχόμενο 60% μουσικής, μόνο 40% αλλά εισμάτιν. Αλλά μια μικρή εταιρεία βλέπετε με 3.000 ευρώ κεφάλαιο κέρδισε το διαγωνισμό με ένα βαθμό διαφορά. Μυστήριο επικρατεί πώ έγινε η επιλογή, η προσφορά είναι στη, η δική μα είναι στο σελίδα, η δική του δεν απεκαλύφθη. Ε, το του Συμβούλιο βγήκε στην επίθεση όταν δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα. Εμεί είπε ότι ήταν προκλητική προσφορά μα, που είναι ψευδέ, και ότι έπρεπε να δώσουμε περισσότερα για την άδεια, είπαν. Προσφύγαμε δικαστικά και το ροδιατηλεπτικό Συμβούλιο κολυσιεργεί και παρεμποδίζει την απόδοση δικαιοσύνης. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι και οι δύο περιπτώσεις θα μπορούσαν να καταλήξουν συμβιβασμό αν και τα δύο μέρη ε, μπορούν, θέλουν να συμβιβαστούν. Η, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο προσπαθεί να φημώσει τις διάφορες φωνές με διοικητικά μέσα, αλλά έχουν και οικονομικά όπλα το πλωστάσιο τους. Το καλοκαίρι του 2010 κάθε δημόσια και κρατική, φορή και και οι διαφημίσεις με το Cobb Radio μπλοκαρίστηκαν. Δεν έδωσαν διαφημίσεις σε εμάς. Ε, έδωσαν σε σταθμούς που είναι υπέρ της κυβερνήσεως. Αλλά μιλάμε για δημόσια χρήματα εδώ. Και οι ιδιωτικοί διαφημιστικοί φορείς ευθυγραμμίστηκαν και ακολούθησαν το παράδειγμα των κρατικών διαφημιστικών φορέων. Είμαστε κατά πολύ ο δεύτερος ε, σε προτίμηση σταθμούς ε, για, για συζητήσεις κλπ. Τριπλασιάστηκαν ε, τριπλασιάστηκε το ακροατήριό μας αλλά μειώθηκαν ε, κατά το ένα, στο 1 τρίτο τα έσοδά μας λόγω λήψης των διαφημίσεων. Η μοίρα του Globe Radio είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον πλουραλισμό των μέσων και την ελευθεροτυπία, αλλά υπογραμμίζει και την ανάγκη, τη θεμελιώδη ανάγκη που υπάρχει, ε, να υπάρχει ένας νόμος για τα μέσα ενημέρωσης που απαγορεύει αυθαίρετες αποφάσεις. Ο νόμος ο Ουγγρικός για τα μέσα ενημέρωσης δεν εξυπηρετεί την ανάπτυξη ελεύθερων μέσων ενημέρωσης πλουραλιστικών μέσων, είναι απλώς ένα εργαλείο στην εργαλειοθήκη ε, της κεντρικής εξουσίας για τα μέσα ενημέρωσης. Να σας ευχαριστήσω τέλος για την υπέροχη αλληλεγγύη και την προσοχή που δώσατε και έγινε ο πιο φημισμένος ε, ο σταθμός στο έγινε ο πιο φημισμένος άσημος σταθμός στον κόσμο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Λάτοφ. Ένα δεκάλεπτο πέρασε και σας προτείνω λοιπόν να πάμε στους εξής, στα εξής μέλη του πάνελ, να έρθουν εδώ για να έχουμε τέσσερα μέλη του πάνελ θα μιλήσουν. Ο τελευταίος γύρος θα είναι ξανά για τον κύριο Ναυράξης. Και θα ακολουθήσουν και ερωτήσεις με απαντήσεις. Ε, καλό λοιπόν να έρθουν οι εξής. Ακτιβιστής. Mr. Thomas Frist Εκπρόσωπος της κοινωνίας των, του Civil Unity Forum, ο κύριος Ανδρέας Οπλάτκας έρθει, πρώην εκδότης του Νόια Τσίτσα Σάιτουνγκ και μετά θα υπάρχει και περιθώριο να πάρει το λόγο ο κύριος Λαβράξης για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Παρακαλώ, καθίστε. Θα συνεχίσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τον λόγο έχει λοιπόν ο κύριος Ατήλα Κόπιας, ο οποίος είναι ακτιβιστής και έχει οργανώσει διάφορες ε, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Έχετε το λόγο. Δέκα λεπτά έχετε. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας όμως, συνοψίστε, να είστε ακόμα πιο σύντομος, διότι αλλιώς δεν θα υπάρχει καθόλου ώρα για συζήτηση. Ε, καλησπέρα σε όλους. Ε, λέγομαι Ατήλα Κόπιας, ε, είμαι ακτιβιστής. Θα προσπαθήσω να μιλήσω γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Είναι πολύ σημαντική ημέρα για μας σήμερα. Ήθελα σήμερα να σας μιλήσω για τη δημοκρατία και πώς οι κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες υποφέρουν. Ε, θέλω να μιλήσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα ε, σημαντικά ε, θέματα για μια τέτοια ακρόαση. Σε 10 λεπτά όμως δεν προλάβω να πω πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να υποθούν. Για παράδειγμα, καταστρέφονται κατοικίες, οι άνθρωποι με αναπηρίες στερούνται τις συντάξεις τους ε, ε, άνθρωποι θύματα καταστροφών ε, έχουν εγκαταλειφθεί από το κράτος, αυξάνονται οι άστεγοι. Θα μπορούσα να σας τα απαριθμώ αυτά όλη μέρα. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα, ιδιαίτερα αν κοιτάξουμε τη στρατηγική 2020 και τα όσα λέει σχετικά με την ε, ένταξη των ε, κοινωνικά μειονεκτικών ομάδων. Σημαντικέ είναι οι συνέπειε όλων αυτών ε, στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν αρκούν τα 10 λεπτά. Θα μιλήσω λοιπόν για του άστεγου και πώ ποινικοποιήθηκε το να είναι κανεί άστεγο στην Ουγγαρία. Τον τελευταίο χρόνο αρκετές ε, τοπικές αρχές ανέλαβαν δράση κατά των αστέγων. Κάποιοι τους ονομάζουν ε, άστεγους εγκληματίες. Ε, εξώθησαν τους ε, αστέγους, κατέστρεψαν τα σπίτια τους παρά το γεγονός ότι έχουμε θερμοκρασίες σε μείον 10 ή μείον 20 βαθμούς κάτω από το μηδέν. υιοθέτησαν νέους κανονισμούς ε, κατά των αστέγων, απαγόρευσαν ε, το κάπνισμα. Ε, γενικά έχουν λάβει πολλά μέτρα κατά των αστέγων σε δημόσιους χώρους. Τον Μάιο του 2011, από τον Μάιο του 2011 είναι έγκλημα να, χρησιμοποιεί, να, να κατοικεί κανείς σε κάποιο δημόσιο χώρο και μπορεί κανείς να πρέπει να πληρώσει πρόστιμο για κάτι τέτοιο. Αυτό έχει ε, εξαπλωθεί τώρα σε εθνικό επίπεδο και οι νομικές συνέπειες είναι πολύ πιο σημαντικές από το να πληρώσει απλά κανείς κάποιο πρόστιμο. Εάν λοιπόν ε, χρησιμοποιεί κανείς ως χώρο κατοικίας κάποιο δημόσιο χώρο ε, μπορεί να σταλεί στην φυλακή για 60 μέρες και να λάβει πρόστιμο 500 ευρώ. Βρισκόμαστε στην Ευρώπη, στην Ουγγαρία και το γεγονός ότι, ότι είναι κανείς τόσο φτωχός που δεν έχει σπίτι και γι' αυτό τον στέλνει κανεί στη φυλακή, αυτή είναι η πραγματικότητα είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι μόνο παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι και ε, σημαντικό, σημαντική παραβίαση του κράτους δικαίου. Ε, ποια είναι η βάση του κράτους δικαίου. Κάποιες ε, πράξεις τιμωρούνται και ο κόσμος μπορείτε να αποφύγει ε, να διαπράττει τις πράξεις αυτές είναι ότι πράξη. Αλλά το να είναι κανεί άστεγο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει κανεί πολύ εύκολα και αυτό ε, τιμωρείται με τον νόμο. Ε, εγώ ε, έχω δικέ μου ε, εμπειρίε σχετικά με το θέμα αυτό. Πέρσι το φθινόπωρο εξάπλωσα σε ένα παγκάκι σε ένα πάρκο και 20 λεπτά αργότερα κατόπιν επειδή κάποιο ε, το είπε στην αστυνομία, ε, με πήραν από εκεί με ε, χειροπέδες. Δεν έκανα τίποτα άλλο, σαν ένα παγκάκι ξάπλωσα, αλλά επειδή οι αρχές θεώρησαν ότι είμαι άστεγος, αποφάσισαν οι αρχέ να παρενεύουν και με πήραν από εκεί με χειροπέδε. Το ίδιο ακριβώ έκανα τρει μέρε μετά, πήρα και κουβέρτα μαζί μου. Αυτή τη φορά όμω φορούσα κουστούμι. Και μάλιστα πήγα στην αστυνομία για να παραδοθώ. αλλά τίποτα δεν έγινε μετά από αυτό. Σε αντίθεση με την ε, προηγούμενη φορά που είχα τηθεί ως άστεγος ε, και ακριβώς επειδή ήξεραν ότι δεν είμαι άστεγος ακόμα και αν ήθελα λοιπόν ε, δεν μπορούσα να συλληφθώ για το έγκλημα αυτό παρότι τρεις μέρες πριν οι ίδιοι άνθρωποι με είχαν πάρει από εκεί με χειροπέδες. Άλλο θέμα. Τι μπορεί να κάνει ένα κίνημα κοινωνικής πολιτικής αν θέλει να διαμαρτυρηθεί κατά μιας τέτοιας κατάστασης. Η Ουγγαρία ποτέ δεν ήταν το καλύτερο παράδειγμα δημοκρατίας ε, και δημοκρατικών θεσμών. Αλλά εάν ε, ε, υπήρξε παραβίαση του νόμου, πάντα μπορούσε να στραφεί κανείς προς κάποιον, να πάει στον εισαγγελέα, να πάει στον διαδιαπροσωλαβητή του πολίτη. Σήμερα δεν μπορεί να πάει κανείς σε κανέναν από αυτούς τους φορείς. Είτε έχουν εξαλειφθεί αυτοί οι θεσμοί ή ε, έχουν επικεφαλείς ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί στην κυβέρνηση. Εάν λοιπόν οποιοδήποτε άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα με κάποιο μέτρο που λαμβάνει η εχουν επικεφαλης ανθρωπους οι οποιοι ειναι πιστοι στην κυβερνηση εαν λοιπον οποιοδηποτε ανθρωπος εχει καποιο προβλημα με καποιο μετρο που λαμβανει η κυβερνηση του κόμματος Φιντές, ε, το, το καλύτερο μέρος που μπορεί να προσφύγει κανείς είναι κάποιος φίλος του εντός του Φιντές. Ε, μπορεί βέβαια κανείς να διαμαρτύρεται, να διαδηλώνει στον δρόμο ή μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωση. Αυτό κάναμε στις 15 Μαρτίου, την ε, επέτειο ε, του, του Ουγγρικού Απελευθερωτικού Αγώνα. Οργανώσαμε λοιπόν μη κυβερνητικέ διαδηλώσεις. Δεν έχουμε λάβει όμως σχετική άδεια. Ε, για τα επόμενα δύο χρόνια ο Δήμος ε, της Βουδαπέστης έχει ε, κλείσει όλους τους χώρους για διαδηλώσεις. Δηλαδή, θεωρητικά μπορεί κανείς να κάνει διαδήλωση, δεν υπάρχει όμως χώρος να το κάνει αυτό. Στις 2 Ιανουαρίου όμως, μπροστά από την όπερα της Βουδαπέστης, διαδηλώσαμε για υπέρ της δικαιοσύνης και και των ε, κοινωνικών θεσμών ε, για ε, το κοινό. Μπορείτε στο διαδίκτυο να δείτε Μπορείτε στο διαδίκτυο να δείτε πώς το παρουσίασαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κρατική τηλεόραση παρουσίασε μια, έναν άδειο χώρο μπροστά από την όπερα. ότι θεωρούσαν, δηλαδή, μάλλον διάδωσαν ότι δεν έγινε διαδήλωση. Λοιπόν, ε, οι δύο ομάδες, οι ακτιβιστές ε, και οι άνθρωποι που είναι όλο και πιο ευάλωτοι και βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας ε, συναντώνται τώρα. Την μέρα του, στις 23 Δεκεμβρίου το ΦΙΤΕΣ υιοθέτησε νέα νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ στις 15 Απριλίου. Εάν μέσα εάν εντό ενό εξαμήνου ε, διαπράξει κανεί κάποιο έγκλημα, μπορεί να λάβει πρόστιμο είτε ε, χιλίων ευρώ ή να ε, μπει στη φυλακή για 75 μέρε. Και αυτό αφορά οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου κατ' επανάληψη. Δηλαδή, είτε πετάξει κανεί τσιγάρο στο δρόμο, είτε κάνει κάτι ακόμα πιο ασήμαντο κανεί. Αν το κάνει αυτό δύο φορέ, ή πάει φυλακή ή, πληρώνει πρόστιμο. Εγώ το, το τελευταίο εξάμεινο Έξι φορές παραβίασα τον νόμο με τον τρόπο αυτό και εάν είχε οργανωθεί η ακρόαση αυτή μετά τις 15 Απριλίου, τότε η κυβέρνηση Ορμπάν θα μπορούσε να με έχει εμποδίσει να, έρθω να παρευρεθώ εδώ σήμερα. Βλέπω ότι είναι παρόν ο κ. Ναυραξής και θα έχει ε, την τελευταία λέξη. Ε, σας παρακαλώ, ε, βάλτε το χέρι, με το χέρι στην καρδιά, πείτε μου, θεωρείτε τη χώρα αυτή δημοκρατική και πιστεύετε ότι ανήκει στην Ευρώπη της κοινωνικής ασφάλειας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή σας τη μαρτυρία. Την, την ακούσαμε με ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια διευκρίνηση που νομίζω ότι είναι πολύ σωστή και επίκαιρη. Ε, αναφερθήκατε στην κατάσταση και όταν, σας, όταν κρατηθήκατε με χειροπέδες μπορείτε να μας πείτε μετά από πόση ώρα απελευθερωθήκατε. 8 ώρες, διότι αυτή είναι η κανονική διαδικασία. Ο κύριος Τόμας Φρίξ τώρα είναι εκπρόσωπος ε, του ε, Φόρουμ ε, Πολιτικών Ελευθεριών που θα πάρει το λόγο το πολύ για 10 λεπτά. Όπως όμως έκανε και ο κύριος Κόπιας, θα εκτιμήσουμε και εμείς αν είσαστε πιο σύντομος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είμαι εκπρόσωπος ε, των μη κυβερνητικών οργανισμών της Ουγγαρίας αλλά και πολιτικός επιστήμων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, εκφράσω τις δικές μου απόψεις για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Το Civil Unity Forum είναι μη κυβερνητική οργάνωση, όπως σας είπα. Είμαι και εκπρόσωπος τύπου αυτής της ε, οργάνωσης που συγκροτήθηκε το 2009 και από τότε προσπαθεί να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία. Έχουμε οργανώσει διάφορες ε, εκδηλώσεις, διαδηλώσεις. Αυτές συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες ε, πολίτες. Επίσης, συνδιοργανώσαμε την ε, πορεία ειρήνης. Μπορεί να την ακούσατε το Γενάρη συγκεκριμένα. 400.000 ήταν οι παρότες σύμφωνα με την αστυνομία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Νομίζω ότι πολλοί από εσάς έχετε μία στρεβλή εικόνα της κατάστασης στην Ουγγαρία. Επί σειρά μηνών, πολλοί ασκούν κριτικές κατά της Ουγγαρίας, του συντάγματος, ε, των θεμελιωδών νόμων, της κυβέρνησης, του πολιτικού συστήματος ε, συνολικά και μεροληπτούν. Μεροληπτούν, βασίζονται σε ατεκμηρίωτες ε, κατηγορίες ότι η κυβέρνηση του Φίντες ε, είναι φασιστική. Τον ε, συγκρίνουν τον ε, Πρωθυπουργό με τον Ούγκο Τσάβης μέχρι και με τον Χίτλερ. Πραγματικά εμείς μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Εσείς μπορεί να βλέπετε εξωτερικά την Ουγγαρία ως δικτατορία, αλλά εμεί εντό Ουγγαρία έχουμε την τύψη ότι ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα όπου υπάρχει κράτο δικαίου, υπάρχουν πολιτικέ ελευθερίε, υπάρχει ελευθερία του τύπου, των μέσων ενημέρωση, μπορούν οι άνθρωποι να βγουν στο δρόμο, να ασκήσουν κριτική κατά τη κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Άρα, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος έχει δίκιο τελικά. Έχουν δίκιο αυτοί οι οποίοι όντα εκτό Ουγγαρία μα βλέπουν ω δικτατορία, ή οι μη κυβερνητικέ οργανώσει που είμαστε μέσα στην Ουγγαρία και βλέπουμε τη χώρα μα ω μια δημοκρατική χώρα, όπου υπάρχει κράτο δικαίου. Το Γενάρη, στην πορεία αυτή, 21 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, εκατοντάδε χιλιάδε ήταν οι άνθρωποι που θεωρούσαν ότι είμαστε δημοκρατία. Τελικά ποιοι έχουν δίκιο, οι λίγοι που είναι έξω από τη χώρα ή οι πολλοί που είναι μέσα στη χώρα. Αν το σκεφτείτε, νομίζω η απάντηση είναι προφανή. Και θα πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη ότι αυτή η φαρσοκομιδία, αυτή η λαροτραγική επίθεση κατά τη Ουγγαρία ουσιαστικά αποπροσανατολίζει και αντί να αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα, στρέφεται σε άλλες θα πρέπει η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι οι επιθέσεις κατά της Ουγγαρία ξεκίνησαν λόγω των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση, τα οποία στράφηκαν κατά των ε, οικονομικών συμφερόντων. Γιατί μιλώ. Τα λεγόμενα ανορθόδοξα οικονομικά μέτρα του 2010, παραδείγματο χάρη ο φόρο στι τράπεζε ή ο φόρο αλληλεγγύη για την κρίση πραγματικά έχω υποψίες πολλές. Από πού προήλθαν οι επιθέσεις, από αυτούς που ένιωσαν να κινδυνεύουν ε, τα συμφέροντά τους, από τους οικονομικούς κύκλους. Η πεποίθηση μου είναι ότι Η χώρα αυτή που είναι μέλος της Ένωσης εδώ και χρόνια, που είναι δεσμευμένη υπέρ της δημοκρατίας για ε, χιλιετίες, δεν είναι αυτή η οποία αποτελεί απειλή για την ε, δημοκρατική και την Ευρώπη. Αντίθετα, απειλή είναι η τεράστια οικονομική όμιλη με τεράστια δύναμη που προσπαθούν να επηρεάσουν και αυτά τα οικονομικά συμφέροντα προσπαθούν να επηρεάσουν χωρίς καν να έχουν εντολή και αρμοδιότητα. Η βασική πρόκληση λοιπόν που έχει να αντιμετωπίσει η δημοκρατία είναι οι παγκόσμιες αγορές που γίνονται ισχυρότερε και από δημοκρατικά εκλεγμένου πολιτικού. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι πολίτες δεν έχουν πλέον λόγο. Μόνο οι παγκόσμιε αγορές. Θα πρέπει λοιπόν να τους ε, αντιμετωπίσουμε. Και αν αποφασίσετε να το πράξετε και να σταθείτε απέναντι σε αυτούς, τότε θα μας βρείτε στο πλευρό σας εμάς, ε, τη μη κυβερνητική οργάνωση αυτή που εκπροσωπώ. Φυσικά και δεν θέλω να υπεκφύγω σε κανένα από τα θέματα που αφορούν την Ουγγαρία και το κράτος δικαίου και μάλιστα τον αντίον θέλω να, να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα γιατί νομίζω ότι από εκεί πηγάζουν και οι παρανοήσεις. Τα μέσα, οι διανοούμενοι, οι πολιτικοί, επιστήμονες πολλές φορές ε, αδυνατούν να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα προβλήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Φυσικά η Ουγγαρία, για να μην παρεξηγηθώ, απορραπέχει απέχει να αποτελεί την τέλεια δημοκρατία. Κάποιοι δηλαδή, ε, κάποιες από τις επικρίσεις είναι δικαιολογημένες και εμείς οι ίδιες οι μη οργανώσεις ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Υπάρχει όμως κάτι σαν τέλεια δημοκρατία, οπουδήποτε στον κόσμο. Κάπου υπάρχει. Παρά τις ε, αδυναμίες και τα σφάλματα, η Ουγγαρία εξακολουθεί να είναι μια δημοκρατία που λειτουργεί. Να σα πω ένα παράδειγμα. Ένα Ολλανδό πολιτικός επιστήμονας έκανε μια διάκριση μεταξύ της ε, δημοκρατίας της πλειοψηφίας και της, ε, μάλλον της πλειοψηφικής δημοκρατίας και της συνενετικής δημοκρατίας. Η συνενετική δημοκρατία είναι αρκετά δεδομένη στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση δηλαδή προσπαθεί να συνεργάζεται με τις μειονότητες του πολιτικού φάσματος για να εξευρεθεί συνένεση. Στον αγγλοσαξονικό κόσμο όμως, που έχουμε δύο ουσιαστικά κόμματα που εναλλάσσονται, ο νικητής τα παίρνει όλα και οι αποφάσεις τελικά λαμβάνονται από το, την κυβέρνηση και δεν συμμερίζεται, μάλλον δεν μοιράζεται το φόρτο να αποφάσουν η αντιπολίτευση. Άλλο ε, μοντέλο μπορεί να ακολουθείτε στις ε, χώρες αυτές και άλλο σε εμά που ίσως ακολουθούμε και το μοντέλο των ε, πρώην κομμουνιστικών χωρών. Προσπαθούμε βέβαια να το αντιμετωπίσουμε, να το εξεργαστούμε το παρελθόν και να αποστασιοποιηθούμε από αυτό τον μπλοκ. Σλοβενία, άλλες χώρες μπορεί να είναι πιο τυχερές. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, από αυτή την πλευρά είμαστε λιγότερο τυχερές, τυχερές χώρες. αυτοί που απέφυγαν 40 χρόνια τώρα τουλάχιστον ε, την κομμουνιστική δικτατορία και ήταν τόσο πιο τυχεροί από εμάς που δεν το καταφέραμε νωρίτερα, νομίζω ότι ίσως να μην καταλαβαίνουν τι βαριά κληρονομιά φέρουμε στους ώμους. Δεν μπορούμε να εξαγνιστούμε εντό αγωγικών εντελώ από το παρελθόν. Υπάρχουν ε, κάποιες παλιές διαδικασίες, υπάρχουν ε, οι παλιοπολιτικοί, πολιτικοί, παλιά σκοπής, κάποιες διαδικασίες παλαιοκομματικέ. Έρχομαι σιγά σιγά στο ε, συμπέρασμα. Γιατί έχουμε μια πλειοψηφική δημοκρατία και όχι μια συναντική δημοκρατία. Παρακαλώ, να έχετε υπόψη σας και τους λόγους και αυτό που λέω και μην πιστεύετε τα πάντα. Μην πιστεύετε αυτά που προσπαθούν να σα περάσουν αυτοί που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη από τη Δύση. Και επειδή προέρχομαι από μια μη κυβερνητική οργάνωση, πρέπει να σα πω ότι οι φιλοδοξίε και οι προθέσει τη κυβέρνηση βρίσκουν σύμφωνου του περισσότερου ψηφοφόρου την, ε, το μεγαλύτερο μέρος της κοινή γνώμης και αυτό το απέδειξε και η πορεία της ειρήνης που κάναμε τον Ιανουάριο. Έχουμε ε, βάλει ε, στόχο, έχουμε το κίνημα το πατριωτικό που το έχουμε ονομάσει και έχουμε φτιάξει και ένα, ένα badge το οποίο φορώ και εγώ στο σακάκι μου Είμαστε κατά του εθνικισμού, αλλά τις εθνικές παραδόσεις τις στηρούμε και είμαστε υπερήφανοι. Είναι εκδότη του Νόια Zeitung, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Εγώ, κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, είμαι ξένος εδώ. Είμαι Ελβετο-Ούγγρος. Εγώ θεωρώ ότι είμαι ε, φιλελεύθερος άνθρωπος. Δεν, δεν εκπροσωπώ όμως κανένα κόμμα, ε, ούτε καμία ε, μη κυβερνητική οργάνωση. Τον ε, αυτό μου μόνο εκπροσωπώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ε, πολλά μέτρα της Ουγγρικής κυβέρνησης τον τελευταίο 1,5 χρόνο ε, τα επικρίνω. Ε, θεωρώ ότι πολλά μέρη της νομοθεσίας είναι λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν τόσο απαραίτητο ο γρήγορος ρυθμός ώστε να αλλάξει το Σύνταγμα και δύο άλλοι βασικοί νόμοι και επίσης ε, πιστεύω ότι μια κυβερνητική οργάνωση ότι ένα κυβερνητικό κόμμα με πλειοψηφία δύο ε, τρίτων ε, θα έπρεπε να δείχνει μεγαλύτερη μεγαλοψυχία απέναντι στην αντιπολίτευση. Σήμερα Δεν θα αναφερθώ στους διορισμούς σε διάφορους ε, φορείς. Ε, δεν θα αναφερθώ σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό νομίζω ήδη έχει γίνει επαρκώς. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Φρίτς ή να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα που έθιξε. Θα ήθελα να μιλήσω για την γενική δυτική κριτική ε, απέναντι στην Ουγγαρία μια κριτική την οποία ε, δεν θα δίσταζα να την ε, περιγράψω ως εκστρατεία. Πολλά θέματα που αναφέρατε ε, θα ήθελα να τα αναφέρω, τα οποία δεν αναφέρθηκαν σήμερα εδώ, θέματα όμως που έχουμε ακούσει από τα στόματα πολιτικών και που έχουμε δει και σε δυτικά δημοσιεύματα για λόγους χρόνου θα σας αναφέρω μόνο κάποια παραδείγματα. Αυτήν την εκστρατεία την θεωρώ λανθασμένη, ε, μη αντικειμενική ε, και τελείως υπερβολική σε χοντρό βαθμό. Καταρχήν ε, επειδή σε μεγάλο βαθμό ε, έχει ξεκινήσει ε, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους της ε, Ουγγαρίας. Στις τελευταίες εκλογές η αντιπολίτευση έχασε με μεγάλο ποσοστό και ε, δεν δέχτηκε το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών. Δεν εκπροσωπώ πια την Zürcher Zeitung, ωστόσο μπορώ ε, να σας πω ότι ήδη τρεις μέρες ε, μετά τις εκλογές ε, με την πένα του κυρίου Κόνραντ ε, δημοσιεύθηκε ένα πολύ επικριτικό άρθρο στο, στην εφημερίδα που εκπροσωπώ. Πολλοί από εσά τους δυτικούς πολιτικούς Ε, δεν γνωρίζουν τα όρια της δικαιολογημένη και μη δικαιολογημένη κριτικής και είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα δεν καταλαβαίνετε ότι, στον, ε, ότι ουσιαστικά δίνεται συνέχεια σε ε, έναν αγώνα ε, εσωτερικοπολιτικό της Ουγγαρίας. Ε, έχει αναφερθεί η κατάργηση της δημοκρατίας ε, στο Σύνταγμα. Ε, στο Σύνταγμα λέει ότι το όνομα του κράτους είναι Ουγγαρία και δύο σειρές πιο κάτω λέει ότι η δομή του κράτους είναι δημοκρατία. Ε, συχνά διαβάσαμε δημοσιεύματα που συγκρίνουν την Ουγγαρία με δικτατορία. Μια εφημερίδα στην ε, Βουδαπέστη πριν λίγες μέρες ε, δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή. Πρόκειται για εφημερίδα της αντιπολίτευσης. Μια επιστολή προς τούτο το κοινοβούλιο με την έκκληση το, κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο να παρέμβει κατά ε, του αυθαίρετου καθεστώτος. Πιστεύετε ότι είναι απόλυτα αρχικό καθεστώς όταν κάποιος μπορεί να δημοσιεύσει κάτι τέτοιο χωρίς ε, να τιμωρηθεί. Ε, εμένα μου φαίνεται, δόξα τω Θεώ, ότι απέχουμε πολύ από δικτατορία και λογοκρισία. Δυστυχώς ε, συχνά η ε, άγνοια πολύ συχνά συνοδεύεται ε, από κακοβουλία. Η Λεμόντ στο Παρίσι δημοσίευσε μία καρικατούρα του Πρωθυπουργού Όρμπαν με στολή Ναζί. Ξέρει κάποιος από σας τι έκανε η πρώτη κυβέρνηση Ορμπάν ε, το 2000 εισήγαγε μέρα ε, ε, για το ολοκαύτωμα στα σχολεία. Η σημερινή κυβέρνηση σε μεγάλο βαθμό έχει ε, περιορίσει ε, και δυστυχώς κατά τη γνώμη μου δεν έχει περιορίσει αρκετά ε, τα κινήματα των δεξιών. Ξέρετε ότι μέχρι τη σημερινή κυβέρνηση οι Ναζί είχαν μνημείο στην Βουδαπέστη ε, πώς επετράπησαν αυτοί οι νεοναζί στη Βουδαπέστη μέχρι να παρεύει η σημερινή κυβέρνηση. Ε, λέγεται συχνά ότι μετράμε με διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Για παράδειγμα, συχνά δεν αναφέρεται συχνά Ε, μιλάνε πολύ για τον εθνικισμό της σημερινή κυβέρνησης και ένα ε, επιχείρημα είναι συχνά ότι η Ουγγρική κυβέρνηση ε, είναι διατεθειμένη να δώσει διαβατήρια ε, στις μειονότητες των γειτονικών χωρών. Να επιτρέπει δηλαδή την ε, διπλή υπηκότητα. Αυτό είναι τόσο τρομερό. Είναι τόσο τρομερό τότε ότι και η Γερμανία ε, στην Πολωνία έχει δώσει υπηκότητα σε 300.000 γερμανόφωνους Πολωνούς. Το πρόβλημα των Ρωμά είναι, έχει πολλές πτυχές. Ε, όταν η Ουγγαρία είχε την προτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήθελε να προτείνει μια ε, ευρωπαϊκή πρόταση. Μπορεί κανείς σίγουρα να επικρίνει πολλά όσον αφορά τη μοίρα των, Ρώμα, των Ρωμά στην Ουγγαρία. Νομίζω όμως ότι η Γαλλία και η Ιταλία όταν αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα δεν είχαν καλύτερο τρόπο ε, αντιμετώπισης. Γι' αυτό η τελευταία μου λέξη θα είναι η εξής. Σας παρακαλώ προσπαθήστε να γνωρίσετε καλύτερα τη χώρα και προσπαθήστε να ε, επιδεικνύετε λιγότερη επιθετικότητα απέναντι στη χώρα. Για τους Ούγγρους λένε ότι έχουν πολύ ισχυρή εθνική συνείδηση. Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Λιγότερο γνωστό είναι ότι μεγάλο μέρος της ουγγρικής κοινωνίας αφενός από τη μία πλευρά ε, θαυμάζουν τον δυτικό κόσμο, από την άλλη μεριά όμως ε, ε, νιώθουν και πίκρα απέναντι στο δυτικό κόσμο και αυτό οφείλεται σε ιστορικούς λόγους, ε, τους οποίους δεν έχω το χρόνο να απαριθμίσω εδώ. Η εκστρατεία αυτή ε, όμως θα πρέπει να ε, συνεχιστεί με αντικειμενική βάση. Εάν συνεχίσετε με αυτήν την αλόγιστη κριτική της χώρας, τότε ε, οι μάζε στην Ουγγαρία που ήδη είναι ε, επιφυλακτικές απέναντι στην ε, ε, Δύση θα εξωθηθούν πιο, πιο πολύ προ τα δεξιά. Το αποτέλεσμα αυτή τη εκστρατεία δεν θα είναι η ενίσχυση της Ουγγαρία στην Ουγγαρία, θα είναι η ενίσχυση του, των αντιευρωπαϊκών εξτρεμιστικών δυνάμεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα προτείνω τον τελικό γύρο που πρέπει να είναι πολύ σύντομο. Για να κάνουμε τουλάχιστον ένα γύρο ερωτήσεων και τα τελικά, τις τελικές δηλώσεις και ανακοινώσεις. Ο κ. Ναυράσκης, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εν τη αυτή περιπτώσει για να επιτρέψω χρόνο για ερωτήσεις, για τελικό γύρο ερωτήσεων και παρατηρήσεων, θα είμαι λακωνικότατος. Δεν θα αρχίσω να αμφισβητώ τα όσα άκουσα. Σέβομαι τις απόψεις που ακούστηκαν, ακόμα και αν δεν ήταν όλες δικαιολογημένες. Και αν κάποιοι δήλωσαν λάθος στοιχεία. Για μία ακόμη φορά να πω ότι θέλουμε εμείς να δεσμευτούμε να συνεργαστούμε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η παρουσία μου εδώ είναι ε, δείγμα της δεσμεύσεως. Όπως και ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δείγμα αυτής της δέσμευσης. Είμαστε δεσμευμένοι για τη συνεργασία μας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Ουγγρική κυβέρνηση είναι πρόθυμη να διεξαγάγει επαγγελματικού τύπου συζητήσεις επί κάθε θέματος νομικού και άλλων, αλλά παρακαλώ ας αποφευθούν οι επιφανειακές επικρίσεις και οι πολιτικές ε, γνώμες να βασίζεται στα στοιχεία της κρίσης σας και να παίρνετε πρώτα τα στοιχεία από όσο των δυνατόν πιο πολλές πηγές και βάσει των στοιχείων αυτών να παίρνετε την απόφασή σας. Και με τα χαρά σας σας βοηθήσουμε, να σας δώσουμε πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε να κάνουμε αυτό που θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για την πραγματική προσπάθεια που κάνετε να συνοψίσετε. Ας ακούσουμε λοιπόν γύρω ερωτήσεων. Ένα, δύο λεπτά το πολύ ο καθένας. Είδε μη, θα έχουμε προβλήματα. Κυρίως με τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κύριε Γιανόκα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ντένις. Ήθελα να σας πω καταρχάς, σας άκουσα προσεκτικότατα. Α, έφυγε. Λυπάμαι που έφυγε ο κύριος Τενής, γιατί ε, είναι πολύ σημαντικό οι εκπρόσωποι των μειονοτικών ομάδων να εισακούονται. Η Ρώμα, οι Εβραίοι και άλλοι. Δυστυχώς δεν υπήρξε αυτή η δυνατότητα. Η Ουγγρική Ένωση ε, Πολιτικών Ελευθεριών επελέγει. Ερώτηση προς αυτούς και αυτοί θέλουν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Ρωμά στην Ουγγαρία μετά το 2010. Γιατί δεν μίλησαν, γιατί δεν κατήγγυλαν αυτή την φρικτή κατάσταση, προσπάθησαν να διορθώσουν την κατάσταση η κυβέρνηση Ορμπάν. Είναι μικρό πρόβλημα περιφερειακό, ανεργία, ελλείψεω, σωστή παιδεία κλπ. Θα χρειαζόταν σωστή στρατηγική για την παιδεία και την απασχόληση. Αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει διαμορφωθεί την τελευταία οκταετία 120 δισεκατομμύρια φιωρίνια εξόδεψε η κυβέρνηση για να ανταχθούν οι Ρώμα ανεπιτυχώς. Όλα επί χάρτου ήταν άριστα, αλλά στην πραγματικότητα δεν πετύχαμε την ένταξη. Θα ήθελα να ξέρω ποια ήταν η άποψη του κ. Ντερές και των εκπροσώπων άλλων μειονοτήτων, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τους ακούσουμε τώρα και δεν μπορέσαμε να αναφερθούμε και στη φτώχεια των παιδιών και το πρόγραμμα καταπολεμήσεως της φτώχειας των παιδιών εφαρμόστηκε ή παρετήθηκε, αφέθηκε το πρόγραμμα πριν αναλάβει την εξουσία η κυβέρνηση Φιντές. Ε, η κυρία Γκούντς που ήταν υπουργό ίσων ευκαιριών είναι εδώ στην αίθουσα πάντα έλεγαν ότι θέλει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα κατά της ένδυας των παιδιών και τώρα έχουμε και ένα ίδρυμα, μάλιστα, προσπαθεί να βοηθήσει τα φτωχά παιδιά να έχουν τουλάχιστον ζεστό γεύμα την ημέρα. Έτσι έχει η κατάσταση σήμερα. Η τελευταία κυβέρνηση είπε πολλά, περισσότερα λόγια, παρά πράξεις, και για τα άτομα με αναπηρίε, τα άτομα με ψυχικές ασθένειες. Κανείς δεν έκανε τίποτα τελευταία οκταετία. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα για να ξοδέψει 7 δισεκατομμύρια φιωρίνια για την βελτίωση της καταστάσεως για την στήριξη των μεγάλων ιδρυμάτων καταργήθηκαν τα μεγάλα ιδρύματα για πάνω από 50 άτομα ε, και βοηθούνται καλύτερα τα άτομα με ε, ψυχικές ασθένειες. Πιο επιστημονική προσέγγιση θα μας βοηθούσε, πιστεύω, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και των Ρωμά και τις στόχες. Δυστυχώς δεν ακούσαμε, όπως σας είπα, επανειλημμένα τους εκπροσώπους αυτής της μειονότητας και δεν είχα τη δυνατότητα να α, θέσουν ερωτήσεις. Θα μας εγκαταλείψουν σε λίγα λεπτά, λέει ο Πρόεδρος. Οι παρακαλώ κυρία Γκόντς, να είσαστε σύντομοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ελπίζω να μην γίνει ουγγρο-ουγγρική αυτή η συζήτηση, να μην καταλήξει ουγγρο-ουγγρική βρίσκω δύσκολο να συμφωνήσω με τα επιχειρήματα που ακούστηκαν, δηλαδή ότι υπάρχει μια συνωμοσία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κόσμου. Ο Ατήλα Κόπιας πώς μπορεί να θεωρείται ε, διεθνής ε, χρηματιστής ο ακτιβιστής αυτός. Και ο κ. Φρίτς αναφέρθηκε στις Ουγγρικές παραδόσεις. Πάντα, ε, εμείς πάντα ψάχνουμε να βρούμε εξωτερικούς αποδιπομπέους τράγους. Από αυτό πάσχουμε. Πάντα κατηγορούμε τους άλλους. Ξέρω και στρέχομαι στη Λίβη ότι είναι περίπλοκο το θέμα των τσιγκάνων. το έχω επεξεργαστεί επί σειρά ετών, επί μακρών Χρειαζόμαστε κατανόηση. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που θα είναι πρόθυμη και ανοιχτή και θα θέλει να αλλάξει τις, τους τρόπους της και την προσέγγιση. Ο άντρε Σόπατκα μας προειδοποιούσε για τα συναισθήματα κατά της Ευρώπης που αρχίζουν και αναπτύσσονται που όλο και περισσότερο ε, γιγαντώνεται αυτό το συνέστημα. Η, η ειρηνική αυτή διαδήλωση οργανώθηκε από το Φιντές και από διάφορες φορείς που στηρίζουν το Φιντές. Αν πάτε στο Facebook μπορείτε να δείτε ποιες οργανώσεις του Φιντές οργάνωσαν την ειρηνική αυτή ε, διαδήλωση και δυστυχώς γίνονται πολλές ομιλίες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε απικία όπως έγραφε ένα πάνω στη διαδήλωση αυτή. Αυτό το συνέστημα, τη του συναισθήματος που αποφύγουμε πάση θυσία και το Φίντες και η κυβέρνηση δημιουργούν τα συναισθήματα κατά της Ευρώπης ενώ στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δούνο του για στήριξη. Καταρχά να ευχαριστήσω τον κύριο Κόπιας για την θαραλέα παρουσίαση του ακτιβισμού και αυτά που έκανε εκείνος και άλλοι πολλοί για να δείξουν λεπτομερώς πώς έχουν τα πράγματα. Σύντομο ερώτημα που να σας εξηγήσετε. Ποια ήταν η διαμαρτυρία, γιατί έγινε διαμαρτυρία μπροστά στο Κοινοβούλιο. Σαν βουλευτές αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να καταλάβουμε γιατί εσείς και άλλοι διαμαρτυρηθήκατε ενώπιον του Κοινοβουλίου. Προς τον κύριο Φρίτς και κάποιον άλλον που είπε ότι ήταν μεγάλη διαδήλωση. Είμαστε υπε... Είπατε ότι είσαστε υπε... υπερήφανοι για την εθνική σα ιστορία. Αυτό που είδα εγώ στι φωτογραφίε ήταν πολύ ισχυρά συνθήματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως και αντισημητικά συνθήματα και πανώ. Σε αυτή την ειρηνική διαδήλωση υπήρχαν αντισημητικά συνθήματα και αντιευρωπαϊκά. Προβληματικό αυτό. Αν διοργάνωνα κάτι θα παρακαλούσα αυτού να φύγουν. Τέλο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν πρέπει να μιλάμε για ιδεολογικά θέματα δεξιά κατά της αριστεράς. Αυτές οι επικρίσεις που κάνω δεν αφορούν ταπείνωση της Ουγγαρίας, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αφορά τις κοινέ ευρωπαϊκές αξίες που ε, ε, συμπεριλαμβάνονται στη, θεμελιώδη, στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η κυρία Φράγερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο τώρα στο τέλος της συνεδρίασης. Γενικά βρήκα Θεώρησα ότι η ε, ακρόαση αυτή δεν ήταν από τις πιο καλές ε, στιγμές ε, του Κοινοβουλίου. Σπάνια έχω δει τόση επιθετικότητα απέναντι σε ένα κράτος μέλος. συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Οπλάτσκα. Ε, νιώθω ότι πολλά που κάνει η κυβέρνηση μπορεί να μην είναι σωστά, αλλά και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και την Ελλάδα και στη Γαλλία και στην ε, Αγγλία, την ε, Γερμανία, πολλές πολιτικές αποφάσεις ε, που λαμβάνονται δεν είναι πάντα σωστές. Βρίσκω λοιπόν ότι αυτό που είπε ο κύριος Οπλάτκα είναι πολύ σωστό ότι με τέτοια στάση θα έχουν ξαφνικά αύξηση οι εθνικιστικές ιδέες. στη Γερμανία δεν συζητήθηκαν ποτέ ως πρόβλημα οι πρόορες συντάξεις. Εδώ και 25 ε, χρόνια έχουμε στη Γερμανία κανόνες ε, για τις πρόορες συντάξεις και θεωρούμε ότι αυτό είναι ε, απαραίτητο. Δεν θέλω να τα εξισώσω όλα αυτά, θέλω όμως αντικειμενική συζήτηση για την Ουγγαρία και θεωρώ ότι το θέμα του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι σημαντικό για μας δεν είναι το μόνο, ε, δεν είναι το μόνο μέτρο, διότι εκεί συμμετέχουν και ε, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Τουρκία, που δεν αποτελούν απαραίτητα μέτρο ε, για μας εδώ ε, στην Ευρώπη. Μια ερώτηση προς τον κύριο Πλάτκα. Πώς πιστεύετε ότι στον δικό μας ε, κόσμο μέσω μαζικής ενημέρωσης και εντός του Κοινοβουλίου ε, πώς, μπορείτε, ε, πώς μπορούμε να κάνουμε πιο αντικειμενική τη συζήτηση. Κυρία Χέσκο, ένα λεπτό παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά διότι παρόλο που είμαι ε, θέλω Ουγγαρέζα θέλαμε ίσω ευρωπαϊκό θέμα. Οι σοσιαλιστέ δημοκράτε, οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν το φθινόπωρο να κάνουν πολιτική διαφήμιση για την ανάγκη για εποπτεία των δημοσ... αγορών και να προωθηθεί ο, φορο... ο συναλλαγών σε όλη την Ευρώπη. Στι 26 χώρε δεν υπήρξαν νομικά εμπόδια. Στην Ουγγαρία λόγω των νέων αυτών, του νέου νόμου για τα μέσα ενημέρωση δεν έγινε αυτή η διαφήμιση. Πώ θα προωθηθούν τα ευρωπαϊκά θέματα ποτέ δεν μπορεί κανείς να ζητήσει να μπει πολιτική διαφήμιση με ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Θα με ενδιέφερε να ξέρω ποια είναι η απάντηση που θα έδιναν ε, τα 26 άλλα κρατημέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σταβάρε, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτή η ακρόαση ήταν χρησιμότατη ε, πλουραλιστική, ποικιλόμορφη. Τώρα ήρθε η ώρα τη περίσκεψη. Ίσως ε, θα πρέπει να επιτόπου να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να δούμε ποια θα είναι τα συμπεράσματά μα τα οποία θα αναφέρουμε. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθήσει ε, Κάποιο έγκυση μετά τη Λισαβόνα έχουμε νέε ευθύνε και εξουσίε για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Νέα Η νέα δομή για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι αρχιτεκτονική, έτσι την αποκαλούμε. Και εδώ και ένα χρόνο βελτιώσαμε την έκθεση στο Κοινοβούλιο και λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι φορεί για τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν βασικό στόχο για να προωθούν του εκείνου που παίρνουν αποφάσει με στοιχεία και δεδομένα. Και μετά παραθέτω. Και μετά οι θεσμοί που παίρνουν τι αποφάσει θα πρέπει να τι λάβουν και να αποφασίσουν σύμφωνα με τι λέει έκθεση, μηδέν ανοχή παραβιώσεων της θεμελιώδους χάρτας, συγκεκριμένες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλα τα θεσμικά όργανα χρειάζεται να ακολουθούν διαφανή και συνεκτικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν δεχόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω, και προσέξτε το αυτό, σχετική σχέσεως, ε, χρήσεως του άρθρου 7 της Συνδίκης Ευρωπαϊκής Ενώσεως επί τη βάση της νέας αρχιτεκτονικής των μελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να είμαστε συνεπείς με αυτά που λέμε και που έχουμε γίνει στην έκθεση που έχει τίτλο Θεμελιώδη δικαιώμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποτελεσματική εφαρμογή μετέθεση θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Αβώνα. Ε, Συνάδελφο Κίνγκεργκαλ είναι ο συντάκτη τη εκθέσεω. Εκτό μικροφώνου ο πρόεδρο. Κύριο Άντε, εσεί το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντικαθιστώ ένα συνάδελφο που έπρεπε να αποχωρήσει και θα ήθελα να πω το εξή. Για μερικού μήνε ακούγαμε διάφορε κατηγορίε που απευθυνόταν κατά της κυβερνήσεως στη Βουδαπέστη και όλες αυτές οι κατηγορίες ίσως να είναι δικαιολογημένε. Λέγεται ότι είναι αυταρχική κυβέρνηση, ακούμε κατηγορίες για αντισημιτισμό, αλλά άμα εξετάσουμε προσεκτικότερα τις κατηγορίες φαίνονται ότι είναι Μιλάμε για θέματα τα οποία είναι εκτός των προνομίων και της δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπως συνταξιοδότηση ή που αφορούν τον εθνικό τομέα όπως νόμο για τα μέσα ενημέρωσης ή θέματα που εμπίπτουν πλήρως στον τομέα της εθνικής αρμοδιότητας όπως είναι το Σύνταγμα και πρέπει να πω ότι εκπλήσω με τα μάλα διότι αυτό το κοινοβούλιο προκαλείται τόσο εύκολα. Αυτό συνέβη κατά το παρελθόν στην περίπτωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας και τώρα έρθει η σειρά του Ουγγαρίας και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το κοινοβούλιο θα, θα την πληρώσουν υπονομεύοντας τελικά την αξιοπιστία τους. Μόνο ένα λεπτό, ο επόμενος αγορητής, λέει ο πρόεδρος, ξεκινάει ο επόμενος αγορητής και λέει ευχαριστώ πρόεδρε, ένα σχόλιο απευθυνόμενος προς την κυρία Λούνατσεκ. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ε, εάν Μα πυροβολείτε με αντισημιτισμό αν δεν έχετε α, αντισημιτική στάση όταν δεν έχετε άλλα επιχειρήματα. Ακούστηκαν κάποια για τον εκλογικό νόμο στην Ουγγαρία. Να πω το εξή. Πρώτον, ο εκλογικό νόμο τη Ουγγαρίας διευκολύνει το εκλέγεστε. Δεύτερον, το νέο σύστημα διευκολύνει τα μικρά κόμματα να καταρτήσουν λίστες. Τρίτον, είναι πιο εύκολο να ξεπεραστεί το 5% για τα κόμματα, το όριο. Τέταρτον, το νέο, ο, νέο, το νέο, ο νέος εκλογικός νόμος απειλάχθηκε από την αναλογική. Αυτό το πρώτο είναι η Επιτροπή της Βενετίας. Υπάρχει κάποιος στην αίθουσα που αμφισβητεί αυτά που σας είπα. Ότι είναι αληθή, αν αμφισβητείτε σηκώστε το χέρι σας. Και αν υπάρχει κάποιος μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής θα τον ενημερώσω για τα στοιχεία. Να κοιτάξτε, για σήκωστε το χέρι, αν τα αφισβητείτε. Χέρι να δω. Δεν μπορώ να το βοηθήσω. Ήμουν αυστηρό όσον αφορά την τελευταία ομάδα παρεμβάσεων των ε, των μελών. Δεν μπορώ να είμαι λιγότερο αυστηρό με το πάνελ. Λοιπόν, ένα λεπτό καθένα, παρακαλώ, για να συνοψίσετε. Με τη σειρά, κύριε Κόπιο, θέλετε να ξεκινήσετε. Όχι, δεν θέλετε, δεν χρειάζεται. Αν όμω το αισθάνεστε, μιλήστε. Δεν απαραίτητο, σα υποχρεώνουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λεπτό, σα χρειάζεται, ορίστε. Λέει ο πρόεδρο, πάρτε το ένα λεπτό σα. Έτσι, ε, έτσι ένα ερώτημα συγκεκριμένο σε μένα και θέλω να απαντήσω. Και να κάνω και μια σύντομη παρατήρηση σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμού ότι οι επικρίσεις κατά τη ε, σημερινή κυβέρνηση η κριτική προέρχεται από το διεθνή χρηματοπιστωτικό κόσμο. Πρέπει να σα πω ότι δεν με πειράζει η χώρα μου. Η κυβέρνηση που έχουμε με πειράζει. Τη χώρα μου την αγαπώ. Τα μέτρα είναι αυτά για τα οποία διαμαρτυρηθήκαμε, διαδηλώσαμε ενώπιον του μπροστά στο Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο, γιατί εγκρίθηκαν κάποιοι νόμοι τότε. Μπορώ να σας δώσω μέρα στα στοιχεία, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Λυπούμε πάρα πολύ που κάνουμε μια συζήτηση για την Ουγγαρία, αλλά τη βασίζουμε μόνο σε φήμες και λόγια. Η, η ειρηνική διαδήλωση ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη βάση. Το λέω εγώ γιατί ήμουν μέλος αυτής της πορείας, αυτής της διαδήλωσης. Δεύτερο και τελευταίο. Νομίζω ότι το πρόβλημα με τη σημερινή συζήτηση είναι ότι έχουμε σήμερα στην Ουγγαρία φιλελεύθερους και μετακομμουνιστές που είναι στην μειοψηφία. Αυτοί επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Και εσείς τους δίνετε βήμα, τους δίνετε φωνή, αλλά δεν ακούτε άλλες φωνές που είναι και οι φωνές της Το 2010 Ολόκληρη η χώρα εξέλεξε το Φίντε και τους Χριστιανοδημοκράτε στην κυβέρνηση. Πήραν την πλειοψηφία, πήραν τα δύο τρίτα. Ίσως να έχει πέσει λίγο τώρα βέβαια, αλλά εξακολουθούν να έχουν την πλειοψηφία. Είναι λοιπόν ε, οι λάθο φωνέ αυτέ που ακούτε. Δεν ακούτε τι φωνέ τη πλειοψηφία των Ούγγρων. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε ίσως να δώσουμε μια άλλη καμπή στη συζήτηση αν ακούγαμε και την πλειοψηφία. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι το κοινοβούλιο ούτε ε, ο δυτικός κόσμος που ε, επιτίθεται στην κυβέρνηση μάλλον είναι οι αντιευρωπαϊστές εντός ε, της Ουγγαρίας. ένα τροχός είναι που ε, γυρνάει και οι δύο πλευρές ε, δείχνουν ε, η μία την άλλη και λένε ότι όχι εσείς φταίτε. Μήπως θα πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω και εσείς και εμείς. Ε, παρότι είμαι πρώην δημοσιογράφος δεν έχω απάντηση 35 ε, χρόνια έκανα τη δουλειά αυτή. Με, με ρωτήσατε τι θα μπορούσε να γίνει για να ε, ε, μπορέσουν τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να βοηθήσουν την κατάσταση. Να βοηθήσουν την κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος καλύτερα και Γι' αυτό απευθύνομαι και στους εκπροσώπους εδώ ε, της ε, κυβέρνησης. Η σημερινή κυβέρνηση θα πρέπει να φροντίσει καλύτερα την ε, πολιτική επικοινωνία της, διότι πραγματικά δεν κάνει πολλά. Final word. Ο κύριος Ναυράξης, τελευταία κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και λάβετε μέρος σε αυτή την συζήτηση. Πρόεδρος, και εγώ ως πρώτος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, τα μέλη του πάνελ, όλους όσους μίλησαν. Να ευχαριστήσω όλους ε, το καθένα από σας ξεχωριστά και αυτά που είπατε. Και να σας πω ότι σίγουρα αυτά θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα εμπνευστούμε σε σχέση με το ψήφισμα. Το οποίο θα πρέπει να ψηφίσουμε στο Στρασβούρο την επόμενη εβδομάδα στην Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας